έπρεπε. άρχεται η Σύνοδος. Θα ξεκινήσω με μία ανακοίνωση. Ε, σε ό,τι αφορά τα πορίσματα της Διευρεμητικής ε, Επιτροπής ε, για τις αιτιάσει παρενόχλησης κάποιων ε, βοηθών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την εξέταση των γραπτών δηλώσεων των ενδιαφερομένων και μετά από ακρόαση με την καταγγέλουσα, επιβάλλεται κύρωση με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 6 και το 166 επιβάλλει κύρωση προς την Μαρία Ζάο Ροντρίγκε για τη συμπεριφορά της προς τη βοηθό που συνιστά ηθική παρενόχληση, ψυχολογική παρενόχληση. Μάλιστα ενημερώθηκε η κυρία Ροντρίγκε δυνάμει του άρθρου 167 του εσωτερικού κανονισμού μπορεί να υποβάλει ε, προσφυγή στο Προεδρείο για την κύρωση. Ε, σε περίπτωση που ασκήσει τέτοια προσφυγή θα ανασταλεί η επιβολή τη κύρωση. Δυστυχώ δεν είναι και πολύ ευχάριστη η ανακοίνωση για την έναρξη τη ολομέλεια. Περνάμε τώρα στο πρώτο σημείο της ημερήσια διάταξη του πρωινού, το ολοκληρωμένο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του ενδοκρινικούς διαταράκτε. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι δεν προβλέπεται διαδικασία catch the για τη συζήτηση αυτή, ούτε ερωτήσεις με την μπλε Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, πριν από 20 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτησε την πρώτη στρατηγική για του οδοκρινικού διαταράκτε. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει από κοινού έκτοτε. Και μάλιστα σήμερα είμαστε παγκόσμιοι ηγέτε στην αντιμετώπιση αυτών των χημικών ουσιών. Από το 1999 απαγορεύσαμε ή περιορίσαμε πολλούς ενδοκρινικούς διαταράκτες. Επιπλέον, είμαστε οι πρώτοι που προβλέψαμε κάποια κανονιστικά κριτήρια για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στην ε, νομοθεσία που υιοθετήσαμε για τα βιοκτώνα και τα φυτοφάρμακα. Επίσης, ε, χρηματοδοτήσαμε την έρευνα και στηρίξαμε διεθνείς οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Βέβαια, δεν αρκούν όλα αυτά. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες ε, εξακολουθούν να αποτελούν παγκόσμια πρόκληση και πηγή ανησυχία και προβληματισμού για πολλούς πολίτες. Δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε τον περασμένο Νοέμβριο την ολοκληρωμένη της ανακοίνωση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Και μάλιστα ε, αυτό είναι έμπρακτη απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσιλωμένη στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος. Και επίση τηρούμε την υπόσχεσή μα να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα κριτήρια για τα βιοκτώνα και φυτοφάρμακα. Η προσέγγιση μας θα πρέπει να συνεχίσει να εδράζεται στα επιστημονικά πορίσματα και στην εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης. Τρεις είναι οι στόχοι που έχουμε κατά νου. Πρώτον, η ελαχιστοποίηση της γενικής έκθεσης στους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Δεύτερον, η επιτάχυση της επιστημονικής πρόοδου. Και τρίτον, η προώθηση εκτενού διαλόγου με όλους τους ενδιαφερομένους. Και μάλιστα καταλήξαμε σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των στόχων που σας ανέφερα. Όλα αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωσή μας και ε, οφείλω να σας ενημερώσω με ιδιαίτερη χαρά ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει το έργο για όλα αυτά τα θέματα και μάλιστα ο εγκάρσιος έλεγχος ε, καταλληλότητας των ενδοκρινικών διαταρακτών θα υιοθετηθεί κατά το πρώτο εξάμεινο του 2020 με 12 ε, δημόσιες διαβουλεύσεις που προβλέπονται για φέτος. Και το 2019 επίσης, φέτος, θα οργανώσουμε την πρώτη της διάσκεψη του Φόρουμ Ενδιαφερομένων και θα εγκαινιάσουμε και την, τον, δικτυακό μας, τον διαδικτυακό μας τόπο, διαδικτυακή πύλη και θα στηρίξουμε φυσικά την σχετική επιστημονική έρευνα. Γνωρίζω ότι μερικοί από εσά απογοητευτήκατε από την ιδέα αυτού του fitness check, του ελέγχου της κατάστασης και της διάγνωσης της κατάστασης. Αυτό δεν είναι συνιστά αναβλητικότητα Απλώς θέλουμε να κάνουμε μια καλή αξιολόγηση και σίγουρα με αυτό το fitness check ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε διάγνωση κατάστασης για να χαράξουμε κατάλληλες πολιτικές. Και μάλιστα έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις για τους οδοκρινικούς διαταράκτες σε διάφορους τομείς. Θέλουμε λοιπόν μία συνοχή σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτών των χημικών ουσιών. Πριν όμω προτείνουμε κάποιε νομοθετικέ αλλαγέ, θα πρέπει προηγουμένω να δούμε τι είδου αλλαγέ χρειάζονται. Γιατί διαφορετική μεταχείριση των διαφόρων ε, ουσιών δεν σημαίνει κατά ανάγκη ε, μη συνεκτική προσέγγιση. Έχουμε κάνει διαφορετικές αξιολογήσεις, αλλά καμία δεν ήταν ε, γενική και δεν κάλυπτε όλα τα ζητήματα. Θα πρέπει μερικά ζητήματα να τα δούμε εγκάρσια. Καταρχήν τα κριτήρια για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών και τις νομοθετικές του συνέπειες. Αυτός ο έλεγχος που θα κάνουμε τις διάγνωση το fitness check, θα ε, πληρώσει αυτά τα κενά και θα μας επιτρέψει να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε νομοθετικά κάποια προϊόντα καθημερινής χρήσης, τα συγκεκριμένα παιχνίδια, καλλιτικά, τρόφιμα και άλλα τέτοια προϊόντα. Ήδη ε, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμή συγκεντρώσει, θα ξεκινήσουμε εκ των μηδενός και Αφού ολοκληρώσουμε αυτόν τον έλεγχο, θα έχουμε όλα τα στοιχεία για να κάνουμε εμπεριστατωμένα ε, την απόφασή μας. Επίσης, ε, οι ευρωπαϊκές ε, υπηρεσίες και τις Ευρωπαϊκές Επιτροπές κάνουν ό,τι μπορούν για να συγκεντρώσουν τα στοιχεία και να εφαρμόσουν απαραίτητες πολιτικές για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Δύο παραδείγματα. Ε, τώρα ολοκληρώνουμε τον κατάλογο δυνητικών ενδοκρινικών διαταρακτών που χρησιμοποιούνται για τα καλλιτικά ε, και μάλιστα θα προσπαθήσουμε πολύ γρήγορα να, να καταθέσουμε και ε, πρόταση νομοθετική. Σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα θα συγκεντρώσουμε μελέτες για τις θελικές ενώσεις και τη σοφενόλη 1 και μόλις ολοκληρώσουμε τις μελέτες θα καταθέσουμε σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Ελπίζουμε έτσι να υλοποιήσουμε τον κοινό μας στόχο και περιμένω τα σχόλιά σας για την, στη συζήτηση. Ευχαριστώ. πολύ και τώρα ακούμε τους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ελ κυρία Γκέρλινγκ, τρία λεπτά. Καλημέρα σας. Εκπροσωπώ τον κύριο Γκίζικερ σήμερα, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο όμω θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μας για την πρόταση του Κοινοβουλίου ε, που είναι ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της εξασφάλισης ενός πλαισίου για την ρύθμιση των ενδοκρινικών διακαταρακτών. Έχουμε να κάνουμε με μια επισκόπηση σημείων στα οποία χρειάζεται περισσότερη δουλειά ε, και αυτό νομίζω το βλέπουμε και με εκφράσεις που ακούστηκαν όπως πρέπει να δουλέψει κάπως πιο σκληρά, να αγωνιστεί περισσότερο κτλ. Πρέπει να επιταχυνθεί η δουλειά της αξιολόγησης. Ε, ευχαριστώ την Επίτροπο για την ιδέα του fitness check, της επαλήθευσης, αλλά εμάς μας ανησυχεί ιδιαίτερος η ταχύτητα και δεν πρέπει να αφήσουμε από το στόχαστρό μα τα θέματα αυτά. Χρειάζονται επενδύσει για όλε τι ουσίε, για όλο το θέμα των ουσιών, το υπογραμμίζουμε στο κείμενο. Ουσίε που χρησιμοποιούνται σε μείγματα χωριστά ή μαζί, τι είδου επιπτώσει μπορεί να έχουν. Και μια και αυτή την εβδομάδα οι βουλευτές χρησιμοποιούν την ευκαιρία της τελευταίας ομιλίας στο στην αίθουσα τη Ολομέλεια. Θα δράξω και εγώ την ευκαιρία για να πω τα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα που μου μένουν ως ευρωβουλευτή. ένα πράγμα για το Brexit. Ένα πράγμα το οποίο έχει μεγάλη σημασία για το θέμα που συζητούμε. Γιατί με το Brexit έμαθα πολλά. Έμαθα ποτέ να μην επιδιώκω έναν στόχο που έχει ιδεολογικό χρωματισμό με παροπίδες. Ποτέ με βάση το ένστικτο ή μία πίστη. Ποτέ με ένα ε, ατονταφέ και χωρίς γνώση των πραγματικών περιστατικών και στοιχείων. Γιατί μετά η πραγματικότητα μας χτυπάει αδυσόπιτα και είναι δύσκολο να γυρίσουμε πίσω. Τι σχέση έχει όλο αυτό με τους διαταράκτες. Πολλά, πολλά πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιδεολογική ιστερία θα έλεγα που έχει ε, αναπτυχθεί σε σχέση με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και σε αυτό, αυτό το βλέπω στην πρώτη τροπολογία ιδιαίτερος που δεν θα υποστηρίξουμε εκ μέρου του ΕΛΚΑ εκεί που αναφέρεται σε ε, υποψίες σε σχέση με, ορισμένου, με τη δράση κάποιων ουσιών ως διαταρακτών χωρίς όμως επιστημονικά δεδομένα. Δεν θα την υποστηρίξουμε λοιπόν. Δεύτερον, το Brexit μας έμαθε ότι πρέπει να παρακολουθούμε τι λένε οι ειδικοί. Το ίδιο και με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, με τρόπο συστηματικό και ψύχρεμο να γίνεται η ανάλυση από τους ειδικού των κριτηρίων. Και με βάση αυτή την ε, αρχή δεν υποστηρίζουμε τις τροπολογίες και ελπίζουμε ότι στην επόμενη ε, περίοδο τη βουλευτική θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντάλη, για δύο λεπτά στους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Η αναβολή δράση όσον αφορά του ενδοκρινικού διαταράκτε είναι κάτι που δεν μα επιτρέπεται. Αυτά τα χημικά ε, ε, είναι συστατικά διαφόρων προϊόντων όπω πλαστικά μπουκάλια, παιδικά παιχνίδια, ε, καλλιντικά και ούτω καθεξή. Αυτέ οι επικίνδυνε ουσίε θα πρέπει να εξαλειφθούν ιδιαίτερα αυτέ που έχουν αποδεδειγμένη επιρροή στου ενδοκρινικού ε, στην ενδοκρινική κατάσταση. Πιστεύουμε όμως πως η Κομισιόν κάνει λίγα και πολύ αργά, γιατί έχουμε το στρατηγικό πλαίσιο, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη συγκεκριμένης δράσης για να δοθεί πλήρη προστασία για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Θα πρέπει, ε, ας πούμε, για τα παιχνίδια και τα καλλιτικά να ε, γίνει δράση. Τελικά έχουμε κατακαιρματισμένες εθνικές προδιαγραφές μπερδεύει τους καταναλωτές που δεν ξέρουν τι είδους προστασία μπορούν να περιμένουν, αλλά και για τους παραγωγούς οι οποίοι ε, υποφέρουν λόγω των διαφορετικών προδιαγραφών. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πορεία εδώ και να βάλουμε πρώτα την υγεία και το περιβάλλον ε, και μένουμε από την Κομισιόν να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογή ώστε να ε, απευθυνθεί και στα χημικά σε ε, προϊόντα όπως παιχνίδια, καλλιτικά και συσκευασίες τροφίμων. Θέλουμε να προστατευτούν οι πολίτες μας. Ε, θέλουμε επίσης μια οριζόντια, έναν οριζόντιο ορισμό σύμφωνο με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει πως το καθημερινό τους περιβάλλον και τα προϊόντα που χρησιμοποιούν δεν βλάπουν την υγεία τους. Και εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκό και το θεμητέ μα ανησυχίε. Είναι πλέον καιρό να αντιμετωπίσουμε του ενδοκρινικού διαταράκτε μια και διαπαντό. Ευχαριστώ. Εξ ονόματο τώρα τη ομάδα της κυρία Ρίση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ε, βρίσκομαι εδώ σε αυτή την Ολομέλεια από το 1999, 20 χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο για του ενδοκρινικού διαταρακτέ έχει εξελιχθεί όταν η επιστήμη η ίδια έχει αλλάξει. Οι ερευνητέ έχουν αποκαλύψει τον αντίκτυπό του στην ανθρώπινη υγεία, την ζωική υγεία και τη σύνδεση με ορισμένε χρόνιε ασθένειε, ορισμένου καρκίνου, τη γονιμότητα, ορισμένα προβλήματα νευρολογική ανάπτυξη. Η σύνδεση αυτή έχει αποδειχθεί. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον, ε, την παγκόσμια αυτή απειλή όπως την ονόμασε το 2013 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή καθυστερούσε στη δράση της, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την καταδίκασε, αλλά ε, δεν έχουμε προχωρήσει πολύ τέσσερα χρόνια μετά και αυτή η νέα στρατηγική ε, αρχίζει να μοιάζει σαν να μην θέλουμε τελικά να μην θέλετε τελικά τελικά να ενεργήσετε. Και στα φυτοφάρμακα ε, αποδιδόταν η ε, επιρροή των ενδοκρινικών διαταραχτών. όμως ε, από ό,τι φαίνεται όλα αυτά τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα θα πρέπει να καταργηθούν και στα καλλιτικά και στα παιχνίδια. Μόνο 8 ουσίες ε, έχουν καταγραφεί ως ενδοκρινικοί διαταράχτες επί τη βάση στη βάση μάλλον των ευρωπαϊκών δεδομένων. Ενώ υπάρχουν πάνω από χίλιες ουσίες. Πριν από λίγες μέρες 90 τέτοιες ουσίες βρέθηκαν σε ένα ποτάμι μόνο στη Γαλλία. Πρέπει να επιταχυνθούν ε, οι, οι, οι δοκιμές, η α αυτή ε, ε, είναι εκτεταμένη η χρήση της στην Ευρώπη. Στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Σουηδία, ε, στην Αυστρία έχουν αρχίσει να νομοθετούν μόνες τους οι χώρες. Εδώ όμως ε, φαίνεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αποκτά όλο της το νόημα. Ακούστε τους ερευνητές. Αυτή η στρατηγική δεν προχωρά αρκετά μακριά. Πρέπει να πάμε πιο γρήγορα και ε, να κάνουμε πιο έντονες δράσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Κονέτσινα τώρα για μισή λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι πραγματικά κρίμα που χρειάζεται και πάλι να απλώς να μιλάμε για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Με την αδράνειά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διακυβεύει την ζωή εκατομμυρίων πολιτών που που παίζουν το, τη ζωή του κορώνα γράμματα. Το 1999 είχαμε την πρώτη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του ενδοκρινικού διαταράκτε. και στο μεταξύ απλώ χάνουμε το χρόνο μα. Ελάχιστη προσπάθεια έχει γίνει και ελάχιστο έργο, όπω είπατε και εσεί. Δεν καταφέραμε να θεσπίσουμε μέτρα για να περιορίσουμε την έκθεση των συμπολιτών μα στις ουσίες αυτέ. Την τελευταία πενταετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε ούτε ένα πράγμα, ούτε μία δράση δεν υιοθέτησε κάτι που έχει ε, ε, προκαλέσει και την επιβλήξη του δικαστηρίου. Είναι παντού ε, οι ουσίες αυτές, στα φάρμακα, στα παιχνίδια, στα τρόφιμα, στα καλλιτικά. Ακόμη και στα παιχνίδια με τα οποία παίζουν τα παιδιά μα, δεν υπάρχουν επιστημονικέ αφιβολίε για τα επιβλαβή αποτελέσματα αυτών των χημικών ουσιών. Έχουμε δώσει αρκετό χρόνο στου παραγωγού να βρουν λύση μόνοι του. Και φυσικά ήταν αναμενόμενο, δεν έκαναν καμία προσπάθεια, δεν βρήκαν καμία λύση. Ενώ εμεί διαπιστώσαμε πώ ε, μα χειραγωγούν και χειραγωγούν και τι επιστημονικέ μελέτε. Η σύγκρουση συμφερόντων των συντακτών των επιστημονικών μελετών είναι ένα πρόβλημα και θα πρέπει να το εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς. Επίση, όπω οι καρκινογόνε και μεταλλαξιογόνε ουσίε ή τοξικέ ουσίε για την αναπαραγωγή, θα πρέπει και οι ενδοκρινικοί διαταράκτε να ε, ρυθμίζονται νομοθετικά και μάλιστα με αυστηρού κανόνε. και θα πρέπει να απαγορεύσουμε τέτοιε ουσίε ολοσχερό σε ένα χρονικό ορίζοντα. Επίση, ε, να καταλήξουμε σε κριτήρια για, το, για τις δοκιμές και τον εντοπισμό τέτοιων ουσιών. Όπω και με τα μεταλλαξιογόνα ή τα καρκινογόνα, ε, δεν υπάρχει καμία ασφαλής οριακή τιμή για την έκθεση στους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Οι οριακές τιμές που έχουμε για τη δυσφενόλη α, για παράδειγμα, είναι υπερβολικά υψηλές. Και έχουμε μελέτες που δείχνουν ε, τα επιζήμια αποτελέσματα της έκθεσης στην δυσφενόλη α και με πολύ χαμηλότερα όρια, κατώτατα όρια και πολύ χαμηλότερες οριακές τιμές. Φυσικά θα υπερψηφίσω το ψήφισμα και να σας ενημερώσω ότι καταθέσαμε πολλές τροπολογίες που το βελτιώνουν γιατί πιστεύω ότι εκφράζουν την απογοήτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω της αδράνειας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και κατά θα ήθελα να πω ότι ακόμη και αν υιοθετήσουμε ένα τέτοιο επικριτικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ψήφισμα και πάλι δεν αρκεί. Ευχαριστώ. Κυρία Ριβαζή, για δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Όντως, διαπιστώνουμε ότι κάθε βουλευτική περίοδος είναι και μια ευκαιρία χαμένη για το θέμα των ενδοκρινικών διαταρακτών. Το είπε και η συνάδελφος, η Διεθνής Οργανώση Υγείας μας λέει το 2013 ότι είναι απειλή για τη δημόσια υγεία και βλέπουμε ότι έχουν συμμετοχή σε πολύ ε, διαδεδομένες ασθένειες όπως η παχυσαρχία, ο διαβήτης, ε, ακόμα και η απώλεια IQ των παιδιών αποδίδεται σε αυτούς. Προβλήματα στην εγκυμοσύνη. Και εσείς τι κάνετε. Το μόνο που κάνετε είναι να προσπαθείτε να κερδίσετε χρόνο. Μία περίοδος ολόκληρη βουλευτική πέραση και είχατε πει ότι υπήρχε στρατηγική για το 19. Ποιος σας έκανε να, να προχωρήσετε στις θέσεις σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια υπουργό από τη Σουηδία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προσέφηγαν κατά της Επιτροπής ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να σας υποχρεώσουν να κάνετε τη δουλειά σας γιατί ήσασταν υποχρεωμένοι να ε, τηρήσετε το δίκαιο και να ορίσετε την περιγραφή του ενδοκρινικού διαταράκτη. Και βεβαίως μεριμνούμε για την προστασία των, ε, της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, εμείς οι βουλευτές. Εσείς από την έλλη μα λέτε «Α, ε, με την αρχή της πρόληψης, ελαχιστοποίηση της έκθεσης κτλ. Αλλά ε, από το γαλλικό ερευνητικό στο ΣΕΝΕΓΕΣ και από άλλα ε, μας λένε ότι υπάρχει αύξηση της παρουσίας και των συνεπειών στον πληθυσμό. Και εσείς το πρόγραμμα δράσης δεν μας προτείνετε. Έχουμε λοιπόν καταθέσει ένα ψήφισμα που σας λέει τώρα και, για, και σε όρους νομοθετικούς προχωρήστε γιατί ούτε ο κοινό οριζόντιο ορισμό δεν έχουμε για το τι μπορεί να είναι στα προσθετικά, στα δοχεία για τρόφιμα, στα παιχνίδια, στα καλλιντικά εκτός από τα βιοκτώνα και τα, τις ουσίες του ρίτς δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός. Και βλέπουμε ότι το ίδιο ισχύει και για όλα τα αιτήματα αδειοδότησης ουσιών. Τι κάνουμε, τι περιμένουμε. Για την προσεχή βουλευτική περίοδο λοιπόν σας καλώ να υιοθετήσετε τις θέσεις των βουλευτών και να εξαλειφθούν όπως και τα καρκινογόνα νευροτοξικά και άλλες ουσίες και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες για τους πολίτες, γιατί δεν έχουμε καθήκον εδώ να υποστηρίξουμε τα λόμπι, αλλά να προστατεύσουμε τους πολίτες. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε τώρα την απάντηση από την Επίτροπο. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σχόλια. Στο 20 χρόνια αφότου εκφράστηκε η πρώτη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς δεταράκτες παραμένουν αυτή πρόβλημα και ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών, όπως όλοι σας επισημάνατε και ενώ έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος ως προς την αντίληψη του τι συνέπειες και τι λειτουργία μπορεί να έχει αλλά και τη διαχείριση του ενδοκρινικού διαταράκτη, συμφωνώ μαζί ότι τώρα πια πρέπει να ανοίξουμε το βήμα και να επιταχύνουμε τις ε, προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη επεσήμανα ότι οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ξεκινήσει την ε, επεξεργασία των προτάσεων που είχαν προεξαγγελθεί από το 2018 για τη στρατηγική. Ταυτόχρονα ε, μελετούμε και τις υφιστάμενες πολιτικές, αυτές που ασκούνται για τους ενδοκρινικούς δεταράκτες ήδη. Αυτό σημαίνει συντονισμό σε διάφορους τομείς πολιτικής, απαραίτητο και στηρίζομαι στην ε, ε, αρρωγή του Κοινοβουλίου για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή προστασία των πολιτών, του περιβάλλοντο αλλά και τη διαφύλαξη τη εσωτερική αγορά, Μια εσωτερική αγορά, η οποία θα κάνει τη δουλειά τη και για να υπηρετήσει τον καταναλωτή, αλλά και να επιτρέψει να ανθίσουν οι επιχειρήσει. Και ολοκληρώνοντα κυρίε και κύριοι, ε, βουλευτές εκ μέρους του συναδέλφου Αντρουκάητης αλλά και προσωπικώς θα ήθελα να ευχηθώ στον κάθε ένα και την κάθε μία από εσά κάθε επιτυχία ε, κάθε καλό σε οποιοδήποτε βήμα ε, επιλέξετε για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Μία πρόταση ψηφίσματο για την ολοκλήρωση του, τη συζήτηση του θέματο αυτού από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών του ECR, ALDE, Πράσινου και Γκουε. Με αυτά ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αργότερα σήμερα. Και στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχουμε την έκθεση της κυρίας Κλούν για, την, για το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Θαλάσσιων Μεταφορών και παρακαλώ την κυρία Κλούν να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και αγαπητοί σκιώδεις ηγητές. Θεωρώ ότι ήταν πολύ θετική συνεργασία μας, πολύ καλή προσπάθειά μας ε, για την αυτιλιακή ενιαία θηρίδα που στόχο έχει να, να διευκολύνει τον κλάδο και τη διακίνηση εμπορευμάτων από τους ευρωπαϊκούς λιμένες. Θέλει να εξασφαλίσει ότι όταν ένα πλοίο λιμενίζεται σε ένα ευρωπαϊκό λιμάνι έχουμε εναρμονισμένες διατυπώσεις που θα πρέπει ο διασαφιστής να εκπληρώνει. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ε, κατακαιρματισμό και δεν είναι εύκολο ο ελιμερισμό σε οποιοδήποτε λιμάνι ή σε κάποια χώρα. Υπάρχει πολύ διαφορετικέ διατυπώσεις για την υποβολή δηλώσεων και μερικέ φορέ σε μερικά λιμάνια έχουμε επιπλέον τέτοιε διατυπώσεις. Θέλουμε λοιπόν μία αναρμόνιση των δεδομένων που απαιτούνται και των στοιχείων που απαιτούνται και αυτό το στόχο έχει η ναυτιλιακή ενιαία θηρίδα και μάλιστα είχα επισκέψει πολλά λιμάνια, είχα συνεργασία με πολλά λιμάνια και είδα και με τα μάτια μου πόσο προχωρημένα είναι μερικά και αλλά όχι τόσο. Θέλουμε λοιπόν όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο χάρη σε μια ενιαία ναυτιλιακή θηρίδα. Όπως σας είπα είχαμε πολύ καλή συνεργασία και στους τριμερείς διαλόγους και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για τις προσπάθειες που έκανε αλλά και τη Ρουμανική Προεδρία γιατί πραγματικά εργαστήκαμε πολύ ομαλά και γρήγορα. Και μάλιστα όλο τυχαίως στην πρώτη συνάντηση που είχαμε ήταν με εκπροσώπους των εφοπλιστών του ναυτιλιακού κλάδου και ενημερώθηκα για τις προκλήσεις τους και χαίρομαι που καταλήγω σε μια πρόταση που θα τους εξυπηρετήσει και θα διευκολύνει και το εμπόριο. Και μάλιστα ε, ε, έχουμε, θα έχουμε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύσεις με τον Κάναδα, έχουμε ήδη υπογράψει συμφωνία και έχουμε και άλλες εμπορικές συμφωνίες και όλοι ε, χρειάζονται και τα λιμάνια και ο ναυτιλιακός κλάδος γενικά χρειάζεται εμπορικές συναλλαγές, κάτι που είναι προς όφελος και των καταναλωτών. Αυτή η νέα ναυτιλιακή θηρίδα θα εξυπηρετεί στους πάντες γιατί εξορθολογίζει το σύστημα και δημιουργεί μια ναυτιλιακή ενιαία θηρίδα, γιατί έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια λιμανισμού το χρόνο στα λιμάνια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μερικές φορές χρησιμοποιείται ακόμη ε, χαρτί ως υπόθεμα, με την μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία θα μειωθούν οι γραφειοκρατικές διατυπώσεις και θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Η αναρμόνιση ε, της υποβολής δηλώσεων θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και θα μειώσει ε, κατά 780 ε, εκατομμύρια μέχρι το 2030 και θα μειώσει κατά το ίμιση το χρόνο υποβολής δηλώσεων χάρη στις αλλαγές της διαδικασίας. Σταθήκαμε σε μερικά θέματα όπως είναι η αναγνώριση των υποδομών που υπάρχουν ήδη στα λιμάνια και η αναβάθμισή τους. Χρησιμοποιούμε ότι ήδη υπάρχει και το βελτιώνουμε. Και επίσης ζητούμε σε έκτακτες προϋποθέσεις να υποβληθούν συμπληρωματικές ε, πληροφορίες, αλλά μόνο υπό όρους. Επίσης η ουδετερότητα η τεχνολογική ήταν μέλημά μας. Αυτό το λάβαμε υπόψη και έχουμε περιλάβει και μια διάσταση διακυβέρνησης. Αυτό επίσης ήταν πολύ σημαντικό και φαντάζομαι θα το αναφέρουν και οι σκιώδεις ηγητές. Το θέμα της διακυβέρνησης ήταν πολύ σημαντικό για μας και για τους ναυτιλιακές εταιρείε. Θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι ο υπεύθυνο, ποιο πρέπει να λογοδοτήσει και πώς θα εντοπιστεί. Πολύ θετική συμφωνία και προσβλέπω στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για να καταφέρουμε πραγματικά να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και το χρόνο που αφιερώνουν ναυτιλιακές εταιρείε στις διατυπώσεις, προκειμένου να διευκολύνουμε την απρόσκοπτη διακίνηση εμπορευμάτων από τους ευρωπαϊκούς λιμένες. Σας ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. Το λόγο έχει επίτροπο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε Βαρβουλευτέ, η Κομισιόν είναι πολύ ικανοποιημένη που οι νομοθέτε έφτασαν σε πολιτική συμφωνία για αυτόν τον κανονισμό που θεσπίζει την το περιβάλλον ναυτιλιακής ενέας θηρίδας. Μπορούμε τώρα να ανταποκριθούμε στο παλιό αίτημα της ε, ναυτιλιακής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία μιας τέτοιας ενιαίας θηρίδας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια κυρία Κλούν, καθώς και τους κοιόδης ε, του, της Επιτροπής Μεταφορών για την εργασία τους και τις αποφασιστικές τους προσπάθειες που επέτρεψαν να φτάσουμε σε μια συμφωνία με ομαλό και ταχύ τρόπο. Σήμερα η ε, μεταφορείς ε, που δαπανούν ε, μια με τρεις ώρες ε, καθημερινά στα λιμάνια για τις αναφορές. Οι νέοι κανόνες θα περικόψουν κατά το ίμιση την διαδικασία και το διοικητικό κόστος κατά δισεκατομμύρια ώρες, εργατόρες. Αυτό θα καταστεί δυνατό μέσω της υιοθέτηση ενός κοινού συνόλου ορισμών και προδιαγραφών της ένταξη των νέων θηριδών σε ένα κοινό οριζόντιο διαλειτουργικό πλαίσιο και έπειτα η πρόβλεψη εναρμονισμένου interface για τις αναφορές. Το νέο περιβάλλον επίσης θα διευκολύνει την ε, διάδοση των δεδομένων και την, και την ε, εκ νέου χρήση αυτών ε, θα εξασφαλιστεί ότι οι αναφορές των πλοίων με τον ίδιο τρόπο θα γίνονται ανεξάρτητα με το ποιο είναι το λιμάνι όπου δένουν. Ε, θα επωφεληθούν επίσης από πιο αποτελεσματική ροή πληροφοριών. Ο τομέας της ναυτιλίας θεωρεί πως αυτός ο κανονισμός είναι από τους πιο, τις πιο σκόπιμες πρωτοβουλίες ε, που στοχεύουν στη βελτίωση της ε, αποδοτικότητας, τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου και έχει ήδη εκφράσει μεγάλη ικανοποίηση με τα συμβαστικά κείμενα. Πιστεύω πως το συμβαστικό κείμενο όχι μόνο ικανοποιεί τα αιτήματα των τριών θεσμών και του ναυτιλιακού τομέα, αλλά επίσης ωφελεί όλο το δίκτυο των ε, ναυτιλιακών μεταφορών μέσω της ψηφιοποίησης και της ευκολότερης ροής των πληροφοριών. Φυσικά αυτό έχει άμεση επιρροή στην ανταγωνιστικότητα και τη δυνατότητα ο ναυτιλιακός τομέας να ενταχθεί στις πολυτροπικές λύσεις μεταφορών. Σας ευχαριστώ και τώρα προχωράμε με τους ομιλητές εξ ονόματος των ομάδων. Ο κύριος Βήμαντε από το ΕΛΚΑ πρώτος. Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, την Δίρντρη, για αυτό το πολύ περίπλοκο ζήτημα. Η ψηφιοποίηση του τομέα των μεταφορών είναι πολύ σημαντική και αν όλα ε, πάνε καλά ε, το σύστημα μεταφορών θα λειτουργήσει πλέον ομαλά. Η ενιαία ναυτιλιακή θηρίδα ε, καλύπτει μια ολόκληρη σειρά θεμάτων. Δεν πρόκειται μόνο, κύριε Πρόεδρε, για χαρτιά που δίνονται στο λιμάνι αλλά και για τα τελωνιακά έγγραφα που αναφέρουν ας πούμε επικίνδυνες χημικές ουσίες και πολλά άλλα πράγματα. Αυτή η οδηγία που υπήρχε πριν από το 2010 ήταν, ε, σχετικ... ήταν πολύ περιορισμένες εμβέλειες και γι' αυτό η ε, Κομισιόν προέβη στη πρόταση αυτή για πιο αποτελεσματικό και διάφανο ε, ε, σύστημα. Εγώ έχω κάποιες ανησυχίες ωστόσο ας πούμε αυτό το Port Community Systems που λέτε, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Εύχομαι η, κυρία Επίτροπος να μεριμνήσει ώστε να λειτουργήσουν ομαλά αυτά τα συστήματα, τα λιμενικά συστήματα. Κυρίες και κύριοι, είναι τελευταία μου ομιλία στο ολομέλη αυτή, στην αίθουσα αυτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις καλές μας σχέσεις και με την ε, κυρία ε, Μπόλση και με τον κύριο Τελίτσκα συνεργαστήκαμε πάντα αγαστά. Μπόρις Βαντερκάμπ, άδειο θα μας φανεί το κοινοβούλιο χωρίς εσάς, κύριε Βαντερκάμπ μου. Ε, Ήσασταν ιδιαίτερα δραστήριος ε, στην Επιτροπή Μεταφορών. Πραγματικά ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστώ μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φλέκενστάιν για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην ε, εισηγήτρια, τους συναδέλφους και εισηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλή συνεργασία στο θέμα αυτό. Ο κύριος στόχος του κανονισμού ήταν ο περιορισμός της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης που οπωσδήποτε έχουμε επιτύχει. Και έχουμε τώρα με τον κανονισμό αυτό λιγότερη γραφειοκρατία για τους εφοπλιστές, ε, για τα πληρώματα, ε, για τη διαχείριση των λιμένων, ανταλλαγή καλύτερη δεδομένων μεταξύ εφοπλιστών και ε, λιμενικών αρχών, αλλά και μεταξύ λιμενικών αρχών διαφορετικών. Και βεβαίως έχουμε να κάνουμε με την ε, στόχευση για καλύτερη κατάρτιση των εργαζομένων στους λιμένες που θα συμμετάσχουν και αναφέρονται και στον κανονισμό, πράγμα το οποίο θα τους ωφελήσει σημαντικά και θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στη δουλειά τους. Ωστόσο, ο κανονισμός δεν φέρνει βελτιώσεις μόνο στη διαχείριση των λιμένων. Τα τελευταία πέντε χρόνια καταφέραμε αρκετά πράγματα δεν είναι ο μόνος ο κανονισμός λοιπόν αυτός. Είχαμε το πακέτο για του λιμένες που πια έχει έρθει η ώρα να υλοποιηθεί σε επίπεδο κρατών μελών με την αποτροπή της υποχρεωτικής απελευθέρωσης, με την διαφάνεια στην, στις συνθήκες εργασίας, με την οδηγία για την εκφόρτωση αποβλήτων που εξασφαλίζει περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, στο τέλος αυτής της θητείας ε, της βουλευτικής περίοδου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία και νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να επενέσουμε τους εαυτούς μας γιατί βοηθήσαμε να ενισχυθεί η Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ιδιαίτερα στο τομέα των λιμένων έχει ωφελήσει την πατρίδα μου την προσωπική, το Αμβούργο. Η κυρία Μάισνερ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, όντως σήμερα Ολοκληρώνω ένα κύκλο γιατί είναι η τελευταία μου ομιλία ως βουλευτού γιατί δεν θα είμαι πια υποψήφια αλλά και γιατί όταν ήρθε το πρώτο πακέτο για τις μεταφορές του 2009 θυμάμαι με τον κύριο Στέρξ, τον Βέλγο συνάδελφο που είχε επεξεργαστεί το προηγούμενο πακέτο δηλαδή την ε, τον κανονισμό για, τα, για την ψηφιακή διαχείριση και ήδη από τότε των λιμένων και ήδη από τότε είχαμε πει ότι χρειάζεται μια μονοθεριδική προσέγγιση κτλ. Και είδαμε ότι η πρώτη αυτή πρόταση δεν είχε φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα στη Γερμανία και αλλού και έτσι τώρα έχουμε προχωρήσει περισσότερο στην ψηφιακή διαχείριση των λιμένων, τουλάχιστον επί χάρτου την έχουμε κατοχυρώσει και αποτελεί ένα, μια σημαντική πρόοδο για την διαχείριση και Κνούτ μου πήρε τα λόγια το στόμα δυστυχώς και οι δυο μας από τη Βόρεια Γερμανία είμαστε. Ήθελα να επισημάνω ότι για, την, για τον τομέα των λιμένων με τη δική σου πρώτα απ' όλα έκθεση Κνούτ Φλέκενστάιν αλλά και χάρη στην πολύ καλή συνεργασία μετά είχαμε την υπόθεση των εκφόρτωση των αποβλήτων, την σημερινή έκθεση πια. Κάναμε πάρα πολλά για τους λιμένες. Και αυτό είναι ορατό πλέον. Και θα ήθελα μια και είναι τελευταία μου ομιλία να εκφράσω ρητά τις ευχαριστίες μου προς όλους και μια και έχω λίγο ακόμα χρόνο, θέλω να πω ότι οι λίγοι που είμαστε εδώ παρόντες, δυστυχώς βέβαια γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα, αλλά οι λίγοι που είμαστε εδώ είμαστε φίλοι καλοί, φίλοι γνωστοί. Αυτά τα 5-10 χρόνια που είμαι εδώ σας έχω γνωρίσει καλά και ελπίζω να ε, έχει ως το δυνατόν καλύτερη πορεία το Κοινοβούλιο, ότι πιο δημοκρατικό υπάρχει στην Ευρώπη, ότι πιο θετικό. Εγώ σταματώ την πολιτική μου δρομία κάτι άλλο θα κάνω. Κυρία Μπούρτσο, ελπίζω να συνεχίσετε κι εσείς ε, καλό ε, δρόμο, εύχομαι σε όλους, καλό δρόμο σε όλους τους φίλους, συναδέλφους από την Επιτροπή των Μεταφορών και καλές θαλάσσιες μεταφορές. Ο Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που είπα στον κύριο Φαντενκάμπ ισχύουν και για σας ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι έχετε αφήσει σημαντικό ίχνος από τη δουλειά σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας ε, αναζητήσουμε, θα μας λείψετε ποτέ. Και τώρα, εκ μέρους της ε, ομάδας EFDD, η κυρία Σέιμουρ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκτιμώ την έκθεση αυτή που είναι πολύ σημαντική και δείχνει πως σημαντικά θέματα έχουν εξορθολογιστεί. Χαίρομαι που το βάρος της γραφειοκρατίας έχει περιοριστεί επιτέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, ανησυχώ για την αποθήκευση των δεδομένων και η παρακολούθηση της συνεχούς τους χρήσης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ισχύ εξαρτάται από την ισχύ του αδύναμου κρίκου της. Οπότε αυτό το θέμα δεν είναι και πολύ θετικό, ειδικά για τα βρετανικά λιμάνια. Η πλειοψηφία των Βρετανικών λιμανιών είναι ιδιωτική ιδιοκτησία. Τώρα, προσωπικά, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η τελευταία μου ομιλία εδώ στην Ολομέλεια και θα ήθελα επ' ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους ε, οδηγούς μεταξύ άλλων που είναι πάντα ε, ευγενέστατοι και πολύ εξυπηρετικοί. Τους ευχαριστώ θερμότατα ανέκαθεν ναι, ήμουν ε, υπέρμαχη των δικαιωμάτων όσων είναι υπέρ του ευρωπαϊκού οράματος, αν είναι αυτή η επιθυμία τη πατρίδα σα. Γνωρίζω ότι πολλοί από εσά ε, πασχίσατε να καταλάβετε γιατί θέλει το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από το ευρωπαϊκό όραμα. Ε, προσπαθήστε να φογκραστείτε και να βρείτε τρόπο να γίνετε καλό γείτονε, γιατί το κόμμα του Brexit ήδη προηγείται στι δημοσκοπήσεις εν ώψη των ευρωεκλογών. Σας ευχαριστώ. Εύχες και σε εσά. Καλή τύχη. Επόμενη ομιλήτρια για δύο λεπτά, η κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μια εύρυθμη λειτουργία των λιμένων ε, βελτιώνει και την εσωτερική αγορά και θα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας ε, ε, να την επιτύχουμε για το καλό όλη της οικονομίας. Ευχαριστώ την εισηγήτρια αλλά και την, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Φάνηκε καθαρά και εξάστερα τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργάζεται και να αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία της. Έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα των λιμένων μας. Και πολύ καλό παράδειγμα των ε, ωφελών της ψηφιοποίησης. Της ψηφιοποίησης στην υποβολή δηλώσεων, στην εποπτεία, στην παρακολούθηση και στην, ε, στις οικονομίες. Ε, θα μειωθεί το κόστος διαχείρισης των λιμένων, ενώ θα αυξηθεί η ποιότητα της διαχείρισης των δηλώσεων. Τα ευρωπαϊκά λιμάνια ήδη είναι πολύ φιλοπεριβαλλοντικά σε σχέση με τα υπόλοιπα λιμάνια του κόσμου. Αλλά με βάση την κυκλική οικονομία θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να έχουμε έναν εναρμονισμένο κατάλογο προσδοκιών από τα λιμάνια μας. Και ε, να δώσουμε έμφαση στην επαραχρησιμοποίηση των υλικών και στους λιμένες, σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο για παράδειγμα, να μην γίνεται αποτέφρωση των ε, λαδιών, αλλά ε, να γίνεται καθαρισμός τους και επαναχρησιμοποίησή τους, αν γίνεται. Επίσης, θα πρέπει να παρακολουθούμε τους στόλους μας, ώστε να εξασφαλίζουμε την τήρηση περιβαλλοντικών προδιαγραφών και κανόνων, είτε για την αλία, είτε για τη διαχείριση των λιμάτων, είτε για τη διαχείριση αποβλήτων που φορέ ή απορριμμάτων που εγκαταλείπονται στα λιμάνια και θα πρέπει να ανακυκλωθούν. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Δεμόντε είναι η ε, ομιλητριά μα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η αύξηση των νέων τεχνολογιών επηρεάζει όλου του τομεί, συμπεριλαμβανομένε και τη κινητικότητα. Έχουμε μεγάλε προκλήσει και πρέπει η Ευρώπη να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία τη στον τομέα αυτό. Πρέπει κάθε φορά που ένα ε, καράβι ελιμενίζεται σε ένα λιμάνι να διεκπεριώσει μια σειρά από διαδικασίες και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε αυτή τη μονοθυριδική προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ των κρατών μελών, πράγμα το οποίο σημαίνει σημαντικό γραφειοκρατικό άχθος ε, για τους εφοπλιστές που Βεβαίω αυτό το άχθο τώρα περιορίζεται σημαντικά με τη μονοθυριδική προσέγγιση και την διασυνδεσιμότητα των διαφόρων συστημάτων που βελτιώνουν και τη χρήση των δεδομένων. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Επίτροπο και το προσωπικό τη. εξαιρετική η δουλειά που έγινε και βεβαίω και όλου του συναδέλφου. Και στα σλοβενικά, τα σβιντένια εμφάλα και στα φριουλάνικα, τη διάλεκτο της περιοχής μου. Σας ευχαριστώ πολύ και ή στο επανεδίν. Uh, Βεβαίως όχι μόνο η τοπική, η, το, πιο λαλιά σας, αλλά και το κρασί της περιοχής σας είναι το φριουλάνο. Κύριε Λιμπεράτης και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, έχω λάβει ερωτήσεις και από εκπροσώπους των λιμένων και από εφοπλιστές. Ε, τι και καινούριο θα επινοήσετε πάλι. Αυτή τη φορά όμως μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι καταλήξαμε σε μια λύση πολύ θετική. Έχουμε μια ενιαία ναυτιλιακή ε, θηρίδα και για το λιμενικό σκέλος και για το ναυτιλιακό σκέλος. Επίσης προτείνουμε ε, μια ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφευθεί ο κατακαιρματισμός. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε καλύτερη ε, διαφάνεια και περιορισμό της γραφειοκρατίας, περιορισμό των γραφειοκρατικών διατυπώσεων. Οπότε θα ε, έχουμε ένα εναρμονισμένο επίπεδο. Πιστεύω όλοι να δουν την ωφέλη αυτή της απλούστευσης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βιμ Βαντενκάμπ, που δυστυχώς έφυγε στο μεταξύ από την αίθουσα, την κυρία Μάισνερ, τον κύριο Φλέκενστάιν για τη συνεργασία και να ευχαριστήσω και τον Μπάβελ για την συνεργασία που είχαμε στην Επιτροπή Μεταφορών και να ευχαριστήσω και την Επίτροπο για αυτή την πενταετή συνεργασία που είχαμε. Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη και σε εσά, κύριε Λιμπεράσκη. θα σας χάσουμε και από την Επιτροπή Μεταφορών και από το Προεδρείο. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ο κύριος Καπούτο, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ εταιρείε ε, θαλασσιών μεταφορών έχουν πάρα πολλέ διαδικασίε να διακπεριώνουν σε κάθε λιμάνι που πιάνουν και επειδή δεν υπάρχει εναρμόνιση αντιμετωπίζουν πολλέ δυσκολίε και επιβάρυνση ανάλογα την περιοχή και το κράτο με κόστο βέβαια σημαντικό για τον κλάδο. Η Επιτροπή μας λέει ότι το προσωπικό των θαλασσιών μεταφορών αφιερώνει 4,6 εκατομμύρια ώρες για να κάνει τις δηλώσεις στα λιμάνια. Έτσι λοιπόν μια ενιαία δήλωση μειώνει σημαντικά τη γραφειοκρατική επιβάρυνση και επιτρέπει την διευκόλυνση του εμπορίου και τον εξυγχρονισμό της κινητικότητας της θάλασσας. Με τον κανονισμό αυτό εξασφαλίζονται οι συνθήκες της μονοθυριδικής και εφάπαξ προσέγγισης με μία μόνο δήλωση σε έναν λιμένα. Πληροφορίες δε που έχουν δοθεί σε αυτήν θα αξιοποιούνται και στους επόμενους ελιμενισμούς. Ευχαριστώ πολύ και κύριε Καπούτο, σε ευχαριστώ και εγώ. Ολοκληρώνω το κατάλογο των αγοριτών. Δεν βλέπω και έτσι κλείνω τη διαδικασία Catch the Eye. Έχω μόνο τον κύριο, έχω τον κύριο Φαρία προς το παρόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν και το πανόραμα της κινητικότητας και οι βιομηχανίες μας πρέπει να γίνουν ηγετικέ όσον αφορά τις μεταφορές. Το ίδιο ισχύει και για τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτός ο κανονισμός είναι ένα απαραίτητο βήμα όσον αφορά την διευκόλυνση των διατυπώσεων που χρειάζονται σε κάθε λιμενισμό του πλοίου. Αυτό μέσω της νέας ε, ε, θηρίδας. Αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να ε, μετατραπούν στην ενιαία θηρίδα ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν τεχνολογικά ε, ο, θαλάσσι, ο των θαλασσίων μεταφορών. Πρέπει να είναι εναρμονισμένη η επικοινωνία, όμως θα πρέπει να έχουμε εναρμόνιση ορισμών και ε, ε, διατυπώσεων. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τον, την Επίτροπο Μπόλς και του συναδέλφους του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα αυτούς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ κύριο Πόσπισιλ για ένα λεπτό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 Ε, φορείς ε, των ε, θαλασσίων μεταφορών με ρώτησαν μήπως τελικά γραφειοκρατικά θα καταστεί πιο δύσκολη κατάσταση. Όμως η ενιαία θηρίδα σημαίνει, είναι λογική. Θα υπάρχουν ξαφείς απαιτήσει από πλευράς των ναυτιλιακών εταιριών. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε, κυρία Επίτροπε, να μην οδηγηθούμε σε μια κατάσταση κατάσταση όπου οι μεταφορείς ε, θα πλημμυρίσουν με περισσότερη ακόμη γραφειοκρατία ε, στην, κατά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Να, μήπως ε, τα, οι απαιτήσει αυτές είναι υπερβολικές. Αν όχι, πιστεύω πως αυτό είναι ο, ο δρόμος να προχωρήσουμε. Να αρμόνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι, φαίνεται να είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ. Thank you, sir. Uh, years ο κύριος ε, πέντε χρόνια μετά που ήρθε εδώ φαίνεται να υπάρχει μια τέλεια συμμετρία. Αρχίσαμε να ακούμε επιχειρήματα για περισσότερη εναρμόνιση, μετά ε, συνδυασμό ε, και συνεργασία στο σχεδί. Στον τελευταία μου ομιλία εδώ ακούμε περισσότερα ακόμα παρόμοια πράγματα. Εγώ πιστεύω πως υπάρχει κάτι ιδιαίτερο ε, όταν ε, κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Ίσως να λειτουργήσει, δεν ξέρω, ίσως να λειτουργήσει. Ε, ενώ λοιπόν τα πράγματα εδώ δεν έχουν αλλάξει και υπάρχει μια συνέπεια εκτός αυτών των το, το, τυχών ωστόσο ένας άνεμος αλλαγής πνέει σε ολόκληρη την Ευρώπη γι' αυτό ε, πρέπει να προσέξουμε ε, ο, αυτός ο άνεμος φυσάει και για τις επόμενες ευρωεκλογέ. όταν θα επανέλθουμε μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός ο κόσμος εδώ και πολύ διαφορετικά τα επιχειρήματα Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία Κατσδιάη και θα ζητήσω από την Επίτροπο Μπούλτση να πάρει και πάλι το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη αυτού του σώματος, καταρχάς σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας που είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τη συνεργασία που μας οδήγησε στο σημείο αυτό. Να τονίσω και πάλι πόσο σημαντική πιστεύω είναι η υιοθέτηση αυτού του κανονισμού ώστε να έχουμε πραγματικά ένα γνήσιο ε, ε, περιβάλλον ναυτιλιακής ενιαίας θηρίδας και έναν ενιαίο χώρο, ναυτιλιακό χώρο. Ε, αυτό θα επιτρέψει, ε, θα ωφελήσει μάλλον ε, το περιβάλλον, θα ωφελήσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και φυσικά η ναυτιλία θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική μια επιπλέον διευκρίνηση ίσως όσον αφορά τα συστήματα κοινότητα, κοινότητας, λιμενικής κοινότητας. Η Κομισιόν δεν θα απαγορεύσει άλλα ε, διόδους αναφοράς με την προϋπόθεση ότι συνδυάζονται και οι ενιαίες θηρίδες και ότι οι φορείς θα, θα, θα έχουν την επιλογή. Από την άλλη πλευρά τα συστήματα ε, λιμενικών κοινοτήτων θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες δεδομένων και θα, δίνουν, θα προσφέρουν προστιθέμενη αξία στα λιμάνια για τους ε, ε, ναυτιλιακούς φορείς, φυσικά εάν συμμορφούνται προς το σύνολο των απαιτήσεων που ορίζονται από αυτόν τον κανονισμό. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τώρα την κυρία Κλούν για τον εξαιρετικό συντονισμό, όλους τους κοιόδης και όλες εσάς συνάδελφοι για την πραγματικά επικοδομητική και στοχευμένη δουλειά που ε, οδήγησε σε αυτό το πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Αγαπητέ Πρόεδρε, σας εύχομαι επίσης ε, καλή επιτυχία για τις επερχόμενες ευρωεκλογέ. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, είναι επίσης η τελευταία μου εμφάνιση ενώπιον του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία ώστε πραγματικά να σας πω πόσο ευγνώμων είμαι για τους όχι πάντοτε εύκολα διαλόγους αλλά πάντοτε επικοδομητικούς διαλόγους και εκτιμώ ότι ποτέ δεν φύγαμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο δύσκολες και αν ήταν αυτές και νομίζω πως αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς όλους τους Ευρωπαίους. Είναι το πνεύμα της δημοκρατίας ότι όσο και δύσκολες και αν είναι κάποιες φορές οι αποφάσεις τελικά τα τελικά πορίσματα πρέπει να τιμούνται ως αποτελέσματα δημοκρατικής διαδικασίας. Να, ήθελα να συνεχίσω σε αυτό το πνεύμα, θέλω να σας καλέσω να συνεχίσετε σε αυτό το πνεύμα όπου και αν ασχοληθείτε και να, ε, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια ανθεκτική, βιώσιμη και δημοκρατική Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν τεράστιο προνόμιο να συνεργαστώ μαζί σας. Σας εύχομαι όλους, σε όλους κάθε επιτυχία σε όποιο δρόμο και να ακολουθήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι το χειροκρότημα μιλάει από μόνο του. Για όλα τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών ε, ήταν πολύ ευχάριστη ε, εμπειρία αυτή η πενταετή συνεργασία μαζί σας από την αρχή και από την ανάληψη των καθηκόντων σας. Ήσασταν και οι πρώτοι που κάνατε την ακρόαση στην Επιτροπή και είχαμε πολύ καλή συνεργασία την πενταετία που πέρασε. Σας εύχομαι καλή τύχη και καλή συνέχεια και νομίζω μιλώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων. Κυρία Ισηγήτρια, κυρία Κλούν, έχετε το τελευταίο δίλεπτο τώρα για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καταλάβατε και από τη συζήτηση και τα σχόλια των συναδέλφων πόσο ευπρόσδεκτη είναι η νομοθετική πρόταση. Γιατί ο κανονισμός αυτός είναι αμοιβαίως υποφιλή, μειώνει το χρόνο υποβολής δηλώσεων κατά 50% είπα εγώ, κατά 60% είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη το καλύτερο. Νομίζω ότι είναι επωφελής για όλους αυτή η πρόταση win-win όπως λέμε, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Ευχαριστώ τους πάντες για τη βοήθεια, την υποστήριξη και το ότι καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ είναι πραγματικά θετικό παράδειγμα το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη όταν ανασκουμπώνεται, ε, όταν συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να κάνουμε πιο ανταγωνιστική την αυθυλία μας και τις, τις συναφείς βιομηχανίες και ε, διευκολύνουμε και την οικονομία και την αγορά θα είναι η τελευταία μου ομιλία στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Ελπίζω όμως να επιστρέψω στην επόμενη και να κάνω και άλλες ομιλίες. Θα εξαρτηθεί από τους ψηφοφόρους μου στην Ιρλανδία και ευχαριστώ την Επίτροπο που με βοήθησε πραγματικά ε, στην Επιτροπή Μεταφορών ε, και με το πακέτο κινητικότητα στα πολυθετική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πρόγραμμα για τα λιμάνια, αλλά και για την ε, οδική ασφάλεια. παρακολούθησε με ενθουσιασμό τις εργασίες σας. Ευχαριστώ τον Βίμβα κάμπ, τον συντονιστή μας, τον ηγέτη μας όπως το λέγαμε, αλλά δεν ε, χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους. Πάντως τον ευχαριστώ γιατί πραγματικά μας καθοδήγησε με στιβαρό χέρι την τελευταία πενταετία ο συντονιστής. Ευχαριστώ την κυρία Μάισνερ για την προσήλωσή της στα ναυτιλιακά και τους εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Νομίζω ότι είναι πολύ θετική αυτή η νότα για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό και την θητεία μας, γιατί πραγματικά κάνουμε κάτι πολύ θετικό και δείχνουμε την υπεπτουσία της Ευρώπης. Πώς μπορούμε χάρη στη συνεργασία να έχουμε θετικά αποτελέσματα και καλά επιτεύγματα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο μέλλον και σε ό,τι καινούριο επιδιώξετε. Ευχαριστώ το αυτό και μας τι ωραίο κλίμα που έχουμε σήμερα. Μακάρι να είναι έτσι όλε οι τελευταίες ε, μέρες πριν από την ε, ολοκλήρωση μιας περίοδου και 200 θα έλεγα τελευταίε. Πάντως και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία στην Επιτροπή των Μεταφορών. Ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει σήμερα και προχωρώ στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. Έκθεση ΤΑΝΓ. για τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αηφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας. Κοιτάω να δω αν έχει έρθει ο κύριος Τάν, μάλιστα. Προχωρούμε ως εκ τούτου. Ε, ε, καλωσορίζω και την ύπατη εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη. Κύριε Τάν, τέσσερα λεπτά για σας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Είχαμε την ε, Ρίτα Τέρνμπερκ, την ε, νεαρή που αγωνίζεται για το κλίμα τις τελευταίες μέρες και μας είπε ότι έχει πιάσει πυρκαγιά και πρέπει να σώσουμε την Παναγία των Παρισίων. Αυτό ακριβώς πρέπει να πούμε. Πρέπει να προχωρήσουμε βέβαια βήμα το βήμα, πέτρα την πέτρα και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σημαντικό ογκόλυθο που μπορεί να μας επιτρέψει να χτίσουμε τη δουλειά αυτή όχι μόνο για μας, αλλά για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τους πολίτες και για τον πλανήτη, για βιώσιμες λύσεις. Η ιδέα ήταν εξ αρχής μια απλή, ριζοσπαστική ιδέα, δηλαδή η αφορία να, γίνει ένα κομμάτι του DNA των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και δεν έχουμε να κάνουμε με τις λύσεις της αηφορίας όσο δυνατόν περισσότερο για κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν, για κάθε λύση, για κάθε είδους αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει. Πρέπει να αξιολογείται ε, η αηφορία αυτή. εύκολο να το πει κανείς, όχι να το κάνει, αλλά βλέπουμε καλά αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις. Έτσι λοιπόν, αηφόρες χρηματοπιστωτικές λειτουργίες δεν μπορεί να είναι κάτι που θα μένει στην άκρη, στη γωνιά. Θα είναι όχι μία δικαιολογία και ένα φιλοσικής για μία αηφόρους επενδύσεις του αντίον. Πρέπει η αηφορία να μπαίνει στο επίκεντρο και στο στόχαστρο και των τραπεζών και των ε, χαρτοφυλακίων και των επενδυτών. Πρέπει δηλαδή να ενσωματώνεται σε κάθε στάδιο λήψεως αποφάσεων χρηματοπιστωτικών. Πρέπει να κινητοποιείται ο κάθε παράγον. Άρα θέλουμε και ευρύ φάσμα και ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, ώστε ο καταναλωτής όταν θέλει να ξέρει τι είδους προϊόν, σε τι είδους προϊόν επενδύει να μπορεί να ενημερώνεται και θέλουμε και ένα ευρύ φάσμα ώστε αυτός ο οποίος παίρνει το ρίσκο και βγαίνει μπροστά ως μπροστάρης να μην ε, τιμωρείται σε σχέση με αυτούς που θα τον ακολουθήσουν. Θέλουμε μια ευρία αντίληψη, δυνατότητες, ε, αξιολόγηση, ευρύ φάσμα αξιολόγησης, δικαιώματα, εκπομπές, συνθήκες εργασίας, όλα αυτά να μπαίνουν μέσα στην αξιολόγηση και ένα πλαίσιο ευρύ αρκετά ώστε να αξιολογεί και τον κίνδυνο αλλά και τον αντίκτυπο σε όρους ε, και αντιμετώπισης και περιορισμού των δυσμενών συνεπειών. Και με τη δέουσα επιμέλεια βεβαίως και θέλουμε και στους, στους τρεις τομείς ε, διαχείρισης της αηφορίας να έχουμε αυτή την εξέταση με ως το δυνατόν ευρύτερο φάσμα επενδυτών, όχι μόνο ένα κομμάτι του χρηματοπιστωτικού τομέα. Άλλωστε, ήδη αυτή την εβδομάδα είδαμε υποχρεωτική ε, επιμέλεια, δέουσε επιμέλεια να ζητούν οι ίδιοι οι φορείς των χρηματοπιστωτικών επενδύσεων, θεωρώντας ότι είναι απαραίτητο να συνδυαστούν, γιατί μπορούν να συνδυαστούν οι οικονομικές ε, αξίες με την αηφορία. Και καλό την Επιτροπή και όλους τους εμπλεκόμενους να ανοίξουν τα θέματα των υποχρεώσεων για ε, ενημέρωση, των, ε, του επίπεδου της δέουσας επιμέλειας και της περιγραφής της και κάθε άλλου στοιχείου που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε προς βιώσιμες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες για τον τομέα τον ίδιο, για βιώσιμες επενδύσεις που δεν χρειάζεται να περιμένουμε να έρθουν από τον ουρανό, αλλά πρέπει να τις καλλιεργήσουμε. Και έτσι, ε, ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω του εκπροσώπου του Κοινοβουλίου, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Συμβουλίου και να, τους και να τους ευχαριστήσω πάνω απ' όλα που μπόρεσαν να ε, γεφυρώσουν τις διαφορές μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα προς όφελος όλων μας. σα ευχαριστώ θερμά. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Τάνκ. Νομίζω ότι είναι αμοιβαία ευχές. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Μαγκερίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση πέρυσι τον Μάρτιο. Ο κανονισμό περί ε, είναι βασικό στοιχείο του σχεδίου δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Και σημαντική πρωτοβουλία στην Ένωση Κεφαλαίου Αγορών για να επιδιώξουμε και να υλοποιήσουμε μέχρι το 2050 μια περιβαλλοντική ουδετερότητα. Επίση, εντάσσεται στην υλοποίηση του στόχου μα του γενικού να συνδέσουμε τα χρηματοοικονομικά με την ανάγκη μια πιο βιώσιμη οικονομία. Οι διαβουλεύσει έδειξαν ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια για το πώ λειτουργούν οι, με, μετέχοντες στη χρηματαγορά και πώς συμπεριλαμβάνουν στις πολιτικές τους ενδικών αντίκτυπο στο περιβάλλον και περιλαμβάνεται αυτό στο, στο ύψο τη αξία των ενεργειακών αποφάσεων, των αποφάσεων για τα περιουσιακά στοιχεία. Και αυτό δημιουργεί κάποια στρέβλαση στι αποφάσει. Έχουμε 185 ε, δισεκατομμύρια κενό επενδυτικό. Φτάνουμε στα 270 δισεκατομμύρια αν περιλάβουμε και τη διαχείριση του ύδατος και των πόρων. Ε, προτείναμε να αφιερωθεί ένα τέταρτο του κοινοτικού προπολογισμού στι συναφεί με το περιβάλλον ε, δράση μέχρι το 2021. Αλλά δεν αρκούν οι κρατικέ δεπάνε. Θα πρέπει και ο ιδιωτικό κλάδο να αναλάβει τι ευθύνε του και να επαναπροσανατολίσει τι κεφαλαϊκέ ροέ προ τη βιώσιμη ανάπτυξη για να αντιστρέψει τι αρνητικέ ε, τροπέ που έχει πάρει η κλιματική αλλαγή. Και γι' αυτό προσθέσαμε κάποιες ε, υποχρεώσεις γνωστοποίησης για αρνητικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα. Έτσι θα περιορίσουμε τα αρνητικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την κοινωνία, άσχετα αν η επενδυτική πολιτική υλοποιεί ένα βιώσιμο στόχο ή όχι. Για παράδειγμα, επενδύσεις προς περιουσιακά στοιχεία που μολύνουν το νερό ή καταστρέφουν την βιοπικιλότητα. Είμαστε υπέρ αυτής της επέκτασης που βελτιώνει σημαντικά την πρόταση γιατί ε, βελτιώνει τη διαφάνεια και την πληροφόρηση των τελικών χρηστών για όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών τη βιωσιμότητα. Με τη συμφωνία αυτή θα αυξηθεί η ποιότητα ε, και των πληροφοριών που δίνονται και επίσης ε, έχουμε μία πειθαρχία στην αγορά και αποφεύγουμε την έκφαση μόνο, την επίφαση μάλλον φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων και στηρίζουμε την οικονομία. Οι χρηματοοικονομικές οντότητε παίρνουν κίνητρα για καλύτερη διαχείριση των κινδύνων βιωσιμότητα. Επίση ενημερώνονται καλύτερα ε, για την βιωσιμότητα των επενδυτικών προϊόντων και των επενδυτικών συμβουλών κάτι που θα αλλάξει την οτροπία των τελικών επενδυτών, των ιδιωτικών επενδυτών. Επίση ε, γίνεται γνωστοποίηση των αρνητικών εξωτερικών ε, αποτελεσμάτων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τις επενδυτικές αποφάσεις. Και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί χάρη στις, στις ε, ταχείες συζητήσεις καταλήξαμε σε συμφωνία και ευχαριστώ τον κύριο Τάνκ γιατί καθοδήγησε τις συζητήσεις αυτές προς ένα πολύ αίσιο αποτέλεσμα. Δεν είναι φυσικά το τελευταίο αυτό βήμα, γιατί συνεργαζόμαστε με τους ε, συνομοθέτες για τα υπόλοιπα τμήματα του ε, της πρότασης για την κλιματική ταξονομία και την εφαρμογή των υπόλοιπων δράσεων που αποτελούν τμήμα του βιώσιμου σχεδίου δράση για τις χρηματοοικονομικές αγορές. Σας ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Το λόγο έχουν οι ομιλητές εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Πιτικά είναι εκ μέρου του ΕΛΚΙΑ για δύο λεπτά. Κάνουμε ένα πραγματικό βήμα προς την πραγματική οικονομία. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε που οδεύουν οι χρηματοοικονομικές ροές. 33 εκατομμύρια είναι το σύνολο, δηλαδή 30.000 δισεκατομμύρια που επενδύονται σε μη βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία ή περιβαλλοντικά επισφαλή επενδυτικά προϊόντα. Και είναι θετικό που μπορούμε πια με την πρόταση αυτή να καθοδηγήσουμε τις επενδύσεις προς ε, τομείς ε, και περιουσιακά στοιχεία που είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Γιατί χρήματα υπάρχουν, θα πρέπει να καθοδηγηθούν σωστά. Και νομίζω ότι το μείζον ζήτημα εδώ είναι η σωστή ενημέρωση, η γνωστοποίηση. Γι' αυτό ο κανονισμός για τις γνωστοποίησεις είναι ε, ο βασικός κανονισμός για οποιαδήποτε ε, προσπάθεια βιώσιμων χρηματοοικονομικών ε, προϊόντων. Θέλουμε όχι μόνο φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, ε, αλλά όλες οι επιδυτικές δράσεις να λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον. Υπάρχει το θετικό, υπάρχει το αρνητικό, αλλά υπάρχει και ένα φάσμα μεταξύ τους. Και δεν μιλούμε μόνο για το κλίμα, αλλά και άλλα ζητήματα, όπως η βιοπικιλότητα για την άμεση χρήση γης, την κατανάλωση του ύδατος, το θέμα του φινικελαίου, η επενδύση στο φινικέλαιο και την κρίση που προκάλεσε. Καταφέραμε να αλλάξουμε τον τροχό και να μεταστρέψουμε την κατεύθυνση των χρηματοοικονομικών προς μια πολύ σωστή πορεία και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους. Ε, το επόμενο βήμα είναι να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή, ώστε να καλύπτει και τι επενδυτικέ επιχειρήσει και οι επενδυτέ να λαμβάνουν τη σωστή ενημέρωση. Και επίση να καλύψουμε όλες τις επενδυτικές επιχειρήσεις, όλ, ανεξαρτήτου μεγέθους, όλα τα επίπεδα της παραγωγικής αλυσίδας, ώστε να ξέρουμε τι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να λαμβάνονται σωστές επενδυτικές αποφάσεις φιλοπεριβαλλοντικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ευχαριστώ συνάδελφε. Δεν βλέπω την κυρία Μπερέση ούτε την κυρία Βιρίνγκ, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρθη εξ ονόματος της ε, ομάδας των Πρασίνων, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πραγματικά ε, που δε, λυπηρό που δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό το φάκελο. Η προοδευτική και ο, ο εισηγητής, που, τον οποίον συγχαίρω, ε, έχουν, ε, οι συντηρητικοί έχουν περιορίσει τόσο πολύ το πεδίο εφαρμογή αυτή τη πρόταση της που τελικά αφορά μόνο μία ελάχιστη αναλογία των, των χρηματοπιστωτικών προϊόντων ε, είναι αποφασισμένοι να μην πάρουν καμία δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Η γνωστοποίηση δεν είναι μέγας κίνδυνος, είναι το μήνυμα που μπορούμε να απαιτήσουμε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα που βλάπτει τόσο την οικονομία μας και το περιβάλλον μας. Θα επαναλάβω, η επιστημονική συνένεση είναι ότι χρειάζεται να δράσουμε για να υπάρξουν μεταβάσεις γρήγορα σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας για να περιοριστεί στον 1,5 βαθμό η παγκόσμια ε, υπερθέρμανση. Μέσα σε 12 χρόνια μόλις οι συντηρητικοί πρέπει να πούμε ότι δεν δίνουν δεκάρα για το μέλλον του πλονίτη μας και σαμποτάρουν το μέλλον των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Ναι, πρόεδρε, εδώ θα μπορούσε να είναι η τελευταία μου ομιλία, αλλά πρέπει να σας πω πως ελπίζω πως η επόμενη θητεία αυτού του Κοινοβουλίου θα χρησιμοποιηθεί ώστε να επανασυνδεθούμε με τους λαού ολόκληρης της Ευρώπης. Θα γίνουν μεγάλες αλλαγέ και θα πρέπει να, ληφθούν, να γίνουν και μεγάλες επιλογές. Να αποφασίσουμε αν θα ε, επιδιώξουμε πραγματική δράση για, το κλίμα ή απλώ θα επιβαρύνουμε τις οικογένειες με τους φόρους ε, ε, να αποφασίσουμε αν θα ε, στηρίξουμε τις οικογένειες ή αν θα συνεχίσουμε να δίνουμε ε, ενθάρρυνση στις τράπεζες και στους πλούσιους. Θα επενδύουμε στα δισεκατομμύρια για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού. Ελπίζω πως θα είμαι ξανά εδώ, αγωνιζόμενος για την Ιρλανδία και αγωνιζόμενος μαζί σας για τη δημιουργία μιας καλύτερης Ευρώπης και καλύτερου μέλλοντος. Ευχαριστώ. Ε, και ζητώ συγγνώμη που είπα ότι είσαι από τους πράσινους. Νομίζω πως ε, αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχω κοιμηθεί και πολύ καλά τις τελευταίες εβδομάδες. Ζητώ και πάλι συγγνώμη. Τώρα θα πάμε στους πρασίνους και με την κυρία Σκοτ Κέτο για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ Πρόεδρε. Με χαρά ακούσαμε το, την, την Κρέτα Τόμπερκ την Τρίτη. Πραγματικά ήταν μαγνητική η ομιλία της, ε, συναρπαστική. Ε, κάλεσε όλους τους πολιτικούς για να προβούν σε δράση. νομίζω πως θα ικανοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη βιώσιμη οικονομία. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ε, εργαλεία για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την κλιματική αλλαγή. Είμαι περήφανη που και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται του κόσμου μέσω των περιβαλλοντικών ε, προδιαγραφών αυτή τη φορά με τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις αηφόρες επενδύσεις, οι πολίτες ε, ε, θα έπρεπε να γνωρίζουν. Όταν ο κόσμος βρήκε ε, ε, κρέας ε, αλόγου στα λαζάνια έγινε χαμός. Θα έπρεπε να γνωρίζουμε και τώρα τι συμβαίνει με τις επενδύσεις. Το Συμβούλιο δεν ανταποκρίθηκε στο δικό μας επίπεδο φιλοδοξίας και εξακολουθεί ε, να πιστεύει πως ο αντίκτυπος των επενδύσεων μπορεί να κρυφτεί από, κρυφτεί από τους ε, πολίτες. Όμως ε, θα πρέπει να μην ε, επιτρέπουμε πια τις επενδύσεις που μολύνουν, αλλά με τις χιλιάδες τους διαδηλωτές ε, στους δρόμους για το κλίμα, καλούμε το Συμβούλιο να, καλέσει, να ακούσει τις επιθυμίες των πολιτών που ζητούν βιώσιμη μετάβαση και τη χρήση του οικονομικού συστήματος για να διευκολυνθεί αυτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι και τώρα εξ ονόματος του EFTD για ένα λεπτό ο κύριος Έθεριτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι επιτέλους τελευταία μου ομιλία. Ας αφήσω τα τυπικά και ας πω ότι πολιτική και οικονομία μαζί δεν πάνε. Το ξέρατε, το είπα. Εντάξει, τελειώσαμε. Και ολοκληρώνοντα, θα θέλω να πω ότι ήταν μεγάλη τιμή που εκπροσώπησα τα δυτικά Midlands, ε, μια περιοχή που αγαπώ σε αυτή την ε, αίθουσα, στις συζητήσεις, πολλούς ανθρώπους τους γνώρισα, τους σέβομαι και Συνεχίζουμε από εδώ και μπρος, όλοι μας, όλοι. Εύχομαι καλή ευημερία σε όλους εσάς, ανεξάρτητα έθνη, ανεξάρτητους ανθρώπους, ανεξαρτησία εύχομαι και πρέπει να πω ότι με όλες τις σχολίες που γνώρισα, ιδιαίτερα είμαι ευγνώμων που είχα τόσο καλούς φίλους και την οικογένεια στο πλευρό μου ιδιαίτερα και δεν θα τραπώ να το πω, τον, μπαμπού, μπαμπά μου και τη μαμά μου που με στά, μου στάθηκαν όλες αυτά, όλα αυτά χρόνια και που ήταν πάντα ασφαλής λιμένας για μένα. Ο πρόεδρος ευχαριστώ πολύ και στους γονείς σας βεβαίως, Του ήρωές σας όπως είπατε και εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Πρόεδρε, η κυρία Βίντερ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον σοσιαλδημοκράτη φίλο και συνάδελφο κύριο Πάουλ Τάνγκ για την πολύ καλή δουλειά του, για την α, ακαταπώνητη προσπάθειά του να εξασφαλιστούν καλές λύσεις. Αγωνιζόμαστε λοιπόν να έχουμε στο μέλλον διαφανείς και α, καλές πληροφορίες από τους οργανισμούς επενδύσεων. Η Γκρέτα Τούνμπερ που ήταν εδώ πριν από δύο μέρε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Περιβάλλοντο μα κάλεσε να αναλάβουμε επιπλέον δράση για να αποφύγουμε κλιματικέ και οικολογικέ καταστροφέ. Ο κύριο Βέμπερ βέβαια δεν είναι εδώ, αλλά θα του πω ότι δεν αρκεί να κάνει κανείς ε, να βγάζει φωτογραφίες για τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ε, για να φαίνεται δίπλα στην Κρέτα, αλλά ταυτόχρονα να μην ε, κάνει τίποτα για να αντιμετωπίσει στην ουσία τα προβλήματα που αυτή επισημαίνει. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν όχι μόνο αναγνώριση των προβλημάτων, αλλά και υλοποίηση των λύσεων. Και αυτό πρέπει να το καταστήσουμε σαφέ στην ε, στον κλάδο. Είναι πολλές οι φορές που κάποια προϊόντα εμφανίζονται ως πράσινα χωρίς να είναι. Δεν έχουμε πια περιθώριο να παίξουμε ούτε με το περιβάλλον ούτε με την κοινωνική αηφορία και στο γραφείο, στο φάκελο για την ταξινομία. Είδαμε ότι είχαμε κάνει εμεί προτάσει όλοι που απέρριψαν οι ε, βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και από τι οποίε θα μπορούσε να προκύψει σαφή ορισμό για το τι μπορεί να είναι αηφόρο ή όχι. Δεν πέρασε αυτό λοιπόν. Ελπίζω στο προσεχές κοινοβούλιο οι συνάδελφοι που θα έχουν τις αρμοδιότητες με την επόμενη επιτροπή να προχωρήσουν περισσότερο. Γίναν σημαντικά βήματα σήμερα, όχι αρκετά αηφόρος οικονομία σημαίνει ότι οι τράπεζες θα αναλάβουν και μέτρα σε σχέση με την διακινδύνευση, εμπλέκοντας και περισσότερο από το ίδιο κεφάλαιο σε επενδύσεις για το περιβάλλον. Αυτό δεν γίνεται ακόμα και βεβαίω σας καλώ να υποστηρίξετε στις ευρωεκλογές του σοσιαλιστές δημοκράτες που αγωνίζονται για την κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική αηφορία. Οι σοσιαλιστές έχουν δύο λεπτά ακόμα με την κυρία Μπέγες. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα από του ε, τελευταίους κανονισμού που θα εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψηφοφορία του. Δεν ξέρω τι θα μπορώ να προβάλλω ως απολογισμό Τη απερχόμενης επιτροπής, αλλά οπωσδήποτε μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τον συσχετισμό, το συνδυασμό των επιτυχή της οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με το περιβάλλον, πράγμα το οποίο οφείλουμε σε πολλούς από τους επιφανείς ε, υπαλλήλου και τα στελέχη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω τον ε, Επίτροπο Ντομπρόφσκη. Και χάρη στην ακαταπώνητη ε, προσπάθεια του Πάουλ Τάνκ, κάναμε σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό. Έχουμε να κάνουμε με ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά το πεδίο εφαρμογή, όπου είχαμε εκφράσει απαιτήσει ώστε κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν να υπάγεται στην υποχρέωση τη ενημέρωση, τη disclosure όπω λέγεται. Αυτό απαιτήσαμε εμεί, αυτό διεκδικήσαμε. Η πρόταση τη Επιτροπή αρχικά στόχευε στην υποχρέωση για το ενεργητικό του τομέα των πράσινων επενδύσεων. Ένα, ένα πρώτο βήμα κατά του greenwashing, του χαρακτηρισμού ως πράσινων επενδύσεων που δεν είναι, αλλά ταυτόχρονα θα άφηνε κάποια περιθώρια μόνο για περιθωριακές επενδύσεις σε κάποιους διαχειριστές χαρτοφυλακίων που θα έδιναν ε, κάτι ψίχουλα στις πράσινες επενδύσεις για να καλύψουν Επιλογέ καθόλου πράσινε στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο. Όχι λοιπόν, καταφέραμε να περάσουμε καλύτερε επιλογέ και κυρίω για τι μεγάλε επιχειρήσει πράσινε επιλογέ και υπογραμμίζουμε ότι πρέπει να αναμορφωθεί όλο ο χρηματοπιστωτικός κλάδο στο, πλαίσιο, στο, στο σύνολό του με το στόχο αυτό, με τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή ενημέρωση για τι συνέπειε των επιλογών που μπορεί να κάνει ο καταναλωτή σε σχέση με το περιβάλλον, τα κοινωνικά και άλλα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα πρέπει να αλλάξουν και οι χρηματοπιστωτικοί παράγοντες στάση για να στηρίζουν καλύτερα την επιλογή την υπέρ του περιβάλλοντο ενό καταναλωτή. Μια σημαντική πρόοδο που θα πρέπει να στηριχθεί και από το επόμενο κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Μπέρε. Και περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. κυρία Γκραπίνη, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Είπατε εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κρίμα που είμαστε τόσο λίγοι στην αίθουσα ενώ συζητούμε έναν τόσο σημαντικό κανονισμό τις βιώσιμες επενδύσεις και τη βιωσιμότητα του χρηματοοικονομικού κλάδου. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι βιώσιμες επενδύσεις στα χρηματοοικονομικά συνδέονται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων ε, στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Είμαστε υπέρ της ε, ε, βιομηχανοποίησης και της πρόθεσης της και είναι ένα θέμα που είναι συναφές με αυτό που συζητούμε. Ελπίζω τελευταία στιγμή έστω να υπερψηφίσουμε το σχετικό κανονισμό γιατί δεν θα πρέπει να έχουμε χρηματοπιστωτικά προϊόντα που δεν θα διέπονται από βιωσιμότητα, αλλά θα πρέπει πρώτα να ενημερώνεται ο καταναλωτή, ο ιδιώτης επενδυτή, να γνωρίζει τα πάντα πριν κάνει τι επενδυτικέ του επιλογέ. Θα πρέπει να γίνει καλύτερη διαχείριση του κινδύνου. Αλλά δεν εννοείται σωστή διαχείριση του μακροπρόθεσμου κυρίω κινδύνου χωρί ενημέρωση για εμπεριστατωμένη απόφαση. Θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και θα αυξηθεί όντω χάρη στον κανονισμό αυτό. έδωσα το λόγο στην κυρία Μπέρες που έφτασε κάπως καθυστερημένα. Θα κάνω το ίδιο και για την κυρία Βίρινγκ εκ μέρους των ε, φιλελευθέρων. Είχαν προγραμματιστεί να μιλήσουν εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, οπότε έχετε δύο λεπτά και εσείς πριν συνεχίσουμε τη διαδικασία του ΚΑΤΣΔΙ που είναι μονόλεπτες παρεμβάσεις. Κυρία Βίρινγκ. Σας ευχαριστώ. Χρειάστηκε πολλούς χρόνους, αλλά επιτέλους καταλήξαμε σε αποτέλεσμα. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επικεφαλεί διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την ψυχραιμία τους, την ιόβια υπομονή τους στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά και για το όραμά τους, αλλά και την επιμονή του και την αιμονή του. Τα τελευταία χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ε, ένας ήταν ο στόχος μας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 180 δισεκατομμύρια ευρώ για να διατηρήσουμε και να υλοποιήσουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχου. Θα τα καταφέρουμε? Μόνο χρόνο θα δείξει. Πάντως προσωπικά πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα βάζουμε τα θεμέλια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, για να υποφεληθούν και οι επερχόμενες γενιές από τις ίδιες δυνατότητες με αυτές που είχαμε εμείς. Οι υπέρμαχοι του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών μας λένε ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει. Ήδη είμαστε κατόπιν εορτής. Θα έπρεπε να είχαμε αναλάβει δράση πριν από 20 χρόνια ήδη και σήμερα δύσκολα θα διορθώσουμε την πορεία που είναι σχετικά μη αναστρέψιμη. Ε, θα πρέπει πάντως ε, να σκεφτούμε ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα στο τέλος αν να κρατήσουμε μια αδιαφανή χρηματοπιστωτική κοινότητα. Θα πρέπει να επιβραβεύονται οι βιώσιμες επενδύσεις και να γίνεται σωστή ενημέρωση. Μόνο έτσι θα διαχειριστούμε την οικονομική, χρηματοπιστωτική και περιβαλλοντική κρίση που διανύουμε. Σας ευχαριστώ και κύριε Σιγητά για τη συνεργασία. Είναι η τελευταία μου ομιλία εδώ και σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία παρόλο που καθυστέρησα να μιλήσω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Είστε πολύ καλή συνάδελφος. Ο κύριος Καπούτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή, τελευταία, αυτή η τελευταία μου παρέμβαση σε αυτή τη θητεία. Και είμαι ικανοποιημένο που παρεμβαίνω για αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την ε, ε, εφορία, την περιβαλλοντική για την οποία έχω εργαστεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτή η συμφωνία προσφέρει εξαιρετικέ ε, ευκαιρίε για επενδύσει. Η πράσινη οικονομία είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία εκατομμυρίων θέσεων εργασία. Σίγουρα αυτή η, οδηγία, το κανονισμός οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση ή ε, γνωστοποιήσεις ε, σχετικά με τους τελικούς επενδυτές ε, είναι πολύ σημαντικοί. Θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν για τις περιβαλλοντικούς κινδύνους, τους κινδύνους διακυβέρνησης μέσα στο πλαίσιο του, καλύτερου, του συμφέροντος των πολιτών. Και όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα την ε, ισότητα των φύλων οδηγούν στην, ε, ε, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Γεια σας σε όλους λοιπόν και στο επανειδήν τον Ιούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως εκ μέρους του Αντιπροέδρου Ντομπρόφσκης, τον οποίο εκπροσωπώ εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Πάουλ Τάνκ και όλους σας για τη συμμετοχή στη συζήτηση, τα σχόλιά σας και ευελπιστώ ότι θα υπερψηφιστεί το ψήφισμα. Συμφωνώ ότι θα είναι σημαντικό βήμα πρόοδου προς τη σωστή κατεύθυνση και πολύ καλός τρόπος να ολοκληρώσουμε ε, την κοινοβουλευτική αυτή θητεία με ένα καλό αποτέλεσμα. Και ελπίζω ε, να τεθεί γρήγορα σε εφαρμογή το νομοθετικό πακέτο που αποτελεί πολιτική προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα τη γνωστοποίηση είναι πολύ σημαντικό. Θα επηρεάσει τι επενδυτικέ επιλογέ υπέρ τη κοινωνία και του περιβάλλοντο και με υψηλά πρότυπα βιωσιμότητα θα αυξήσουμε τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ελκυστικότητα των βιώσιμων επενδυτικών προϊόντων και θα έχουμε και μια ευαισθητοποίηση τη αγορά για θέματα βιωσιμότητα. Θα προωθήσουμε την καινοτομία σε επενδυτικέ στρατηγικέ και το σχεδιασμό των επενδυτικών, χρηματοοικονομικών μάλλον προϊόντων. Πιστεύω ότι με τον κανονισμό αυτό θα έχουμε μια αλλαγή νοοτροπία στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, ελπίζω τουλάχιστον, και στου επενδυτέ και θα προωθήσουμε επενδύσει σε μια πιο βιώσιμη οικονομία. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό βήμα προόδου ε, στο θεματολόγιο μας υπέρ της αηφορίας και της βιωσιμότητας. Σας ευχαριστώ και πάλι και ελπίζω να υπερψηφιστεί το κείμενο αυτό αργότερα. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε και κύριε Τάνκ, κύριε Σιγητά, έχετε το δίλεπτο για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιο δράσης ε, για, τη βιώσιμα, για τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά θέματα. Ήταν πολύ κρίσιμη αλλαγή, ε, ευπρόσδεκτη και χαίρομαι που συμβάλαμε και εμείς ε, στα πρώτα βήματα. Όπω είπαμε είναι τα πρώτα βήματα και όχι το τελευταίο, επουδενή. Και σίγουρα κύριε Καρθή θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να προχωρήσουμε, αλλά κάναμε τα πρώτα βήματα που δίνουν ένα σαφές μήνυμα προς το χρηματοπιστωτικό κλάδο ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι κάνουμε μια μεταστροφή προς πιο βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και αυτό θα ακολουθήσουν και άλλα βήματα και απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αποπτικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειες. Και ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει. Ελπίζω να είμαι και εγώ σε αυτούς που θα το στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και αν μείνω εκτός πάλι θα συμβάλλω στη συνέχιση αυτών των αλλαγών. Σίγουρα πολλά αλλάζουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από την αγγλοσαξονική αμερικανική παράδοση του να σπέβδουμε, να προχωρούμε γρήγορα και να τα σπάμε όλα. Γιατί οι εταιρείε και χρηματοπιστωτικέ οντότητε είναι φορεί μια οικονομία που καθοδηγείται κυρίω από νομισματικά κίνητρα. Θα πρέπει να επανέλθουμε στην ευρωπαϊκή μα παράδοση, να λαμβάνουμε υπόψη τι εταιρείε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που θα λαμβάνουν υπόψη το συμφέρον όλων των ενδιαφερομένων και τη κοινωνία. Να επιστρέψουμε στην στην ευρωπαϊκή παράδοση όπου οι τράπεζε, οι ασφαλιστικές εταιρείε, οι επιδετικέ επιχειρήσεις είναι τμήματα της κοινωνίας μας και με γνώμονα το συμφέρον τη κοινωνίας δρούν. Μεταξύ άλλων, αυτή την αλλαγή χρειαζόμαστε, που ήδη έχει ξεκινήσει. Βλέπω κάποιου πρωτοπόρου ε, και σκαπανεί αυτέ τι αλλαγέ. Βέβαια, ως ε, ε, πολιτικός είμαι αισιόδοξο, αλλά βλέπω πολύ θετικού ιονούς που δείχνουν αυτή την αλλαγή και ελπίζω να συνεχιστεί για να έχουμε μια δικαιότερη και πιο ίση κοινωνία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η συζήτηση ολοκληρώνεται εδώ. Η έκθεση θα ψηφιστεί σήμερα. Το επόμενο θέμα στην ημερησία αφορά, αφορά την Κίνα και ιδιαίτερα τις θρησκευτικέ ε, μειονότητες. Έχω μια σειρά από συντάκτες. Ο κύριος Μπέλτερ, για ένα λεπτό. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. In mijn laatste plenaire bijdrage Στη διάρκεια αυτών των τελευταίων ε, παρεμβάσεων στην Ολομέλεια θέλω ακόμα μια φορά να υπερασπιστώ την ελευθερία των, ε, ε, των στην Κίνα. Υπάρχουν αυταρχικές εκστρατείες τις οποίες στηρίζει ο πρόεδρος ΣΥ τα τελευταία χρόνια που αρνούνται τα ελεύθερα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελεύθερη την ανεξιθρησκεία. Οι χώροι καταστέλλονται, τους κλείνουν σε καταβλισμούς ε, συμμόρφωσης. Πώς ε, μπορούμε εμείς να συνεχίζουμε, ενώ εκατομμύρια χριστιανοί είναι ε, έγκλειστοι και που διώκονται οι χριστιανοί. Πρέπει εδώ αυτό να το καταγγείλουμε. Μιλάμε για άρνηση του πολιτισμού. Οι Κινέζοι έχουν παγκόσμια επιρροή. ευχαριστώ το Θεό για τη βοήθειά του και σας εύχομαι να είναι μαζί σας. Ο Θεός μαζί σας. Ο κύριος Μπουτικόφερ δεν είναι εδώ, οπότε θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Σόλτς. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είπατε εκπρόσωπε σε μια στρατηγική εταιρική σχέση είναι σημαντικό να έχει κανείς την πολιτική βούληση και το θάρρος για να αναφέρεται και να θίγει θέματα τα οποία, στα οποία μπορεί να έχουν οι εταίροι διαφορετικές τοποθετήσεις και προσεγγίσεις και γι' αυτό ε, με γεμίζει ανησυχία όταν ακούω ότι υπάρχουν αλλαγέ ω προς τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μια χώρα την οποία επί δεκαετίε παρακολουθώ με φιλικό πνεύμα. Με ενθαρρύνει βεβαίως η πρόσφατη αποδοχή του χάρτη των ανθρωπινών δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών ε, στην ε, δήλωση ολοκλήρωσης του, της Συνόδου Κορυφής της 9ης Απριλίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνα. Ωστόσο, έχουμε πολλά ζητήματα ανθρωπινών δικαιωμάτων στην περιοχή Σιντζιάνγκ του Νουηγούρων και τα έχουν επισημάνει μέχρι και είπατε τη εκπρόσωπο Μισελ Μπασιλέ των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί η Κίνα να παρετηθεί από την πολυμορφία τη. Χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται να γίνουν προσπάθειε για διερεύνηση των συνθήκων διαβίωση και αντιμετώπιση των Ουιγούρων στην περιοχή του Σιντζιάνγκ ε, σε σεβασμό άλλωστε και άρθρων σημαντικών της, ε, ε, του ίδιου του Κινέζικου Συντάγματος που απαγορεύουν την κράτηση σε στρατόπεδα για, για μακρές χρονικές περιόδους. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να δούμε ότι, ότι συνάδει με την ιδέα της σύγχρονης και ανοιχτή οικονομία τη Κίνα, αυτή η αντίφαση σε σχέση με την ε, κράτηση, μακροχρόνια μάλιστα κράτηση ε, ανθρώπων πάνω σε κατασκευασμένε ή πολύ ισχνέ υποψίε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Μπουτικόφερ, είχαμε ανοίξει τον πληστηριασμό για τη δική σας ομιλία, γιατί Λίπατε, αλλά μια και δεν τη ζήτησε κανείς, περάστε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα λίγα δευτερόλεπτα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, των πολιτικών ομάδων, των διαφόρων πολιτικών ομάδων, για την ε, συνεργασία σε θέματα ανθρωπινών δικαιωμάτων, για το γεγονός ότι ειδικά σε θέματα θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων έχουμε μπορέσει να εκφράσουμε συνένεση και συνενετικές θέσεις εδώ στο Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην τις εκφράζουμε, να μην τις διατυπώνουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πάντα, με τις ίδιες λέξεις, αλλά από κοινού ξέρουμε και ε, προχωρούμε μαζί για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι είναι θεμέλιο στη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας στα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα θεμέλιο το οποίο και για μας, για την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια δεν μπορεί ποτέ να πάρει δεύτερη ή δευτερεύουσα θέση. Και θα ήθελα σε αυτό να αναφερθώ σε δύο ε, προσωπικότητες, τον πρόεδρο Τούσκ, ο οποίος στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας κατέστησε σαφές ότι έτσι βλέπει τα πράγματα ο ίδιος. Μακάρι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ηγέτιδες να είχαν την ίδια στάση και θέλω να το αναφέρω ρητά και επίσης θέλω να μιλήσω και για τον πρόεδρο της Volkswagen, ο οποίος κατά τρόπο στο ενώπιον τον, ε, της κάμερας του BBC δήλωσε ότι δεν έχει ιδέα για τα όσα ανέφερε ο κύριος Σόλτς μόλις τώρα και τις κρατήσεις των Ουιγούρων στην Κίνα. Δεν είναι δυνατό να κάνουμε ότι παραγνωρίζουμε τα ανθρώπινα, ότι αγνοούμε μάλλον τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να τηρείτε αυστηρά το χρόνο σας γιατί έχουμε μεγάλη πίεση. Ο κύριος Λάινεν για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Κυρία Μογκερίνη, θα θυμάστε οπωσδήποτε ότι στην πρώτη συνεδρίαση της ε, πενταετίας αυτής σας είχα παρακαλέσει να προχωρήσετε σε μια νέα στρατηγική για την Κίνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα περιλάμβανε όχι μόνο θέματα οικονομικών συναλλαγών, αλλά και ζητήματα πολιτικών σχέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί το πράξατε. Έχουμε λοιπόν μία νέα στρατηγική, ανανεωμένη στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, ε, η οποία εξετάζει επακριβώς ε, τα τεκτενόμενα στο η μεγάλη αυτή χώρα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα αντιμετωπίσουμε εμείς. Είναι μια τεράστια χώρα έχει κάνει τεράστια βήματα βγάζοντας 700 εκατομμύρια ανθρώπους από συνθήκες φτώχεια, τεράστιο επιτευγμά, αλλά τώρα βλέπουμε δυστυχώς τεράστια οπισθοδρόμηση στον τομέα των ελευθεριών των οποίων χαίρουν οι πολίτες εκεί στο τελευταίο δε συνέδριο του κόμματο. Βλέπουμε ότι μπορεί το κόμμα να ορίζει κάθε λεπτομέρεια της ε, ζωής ε, και βέβαια και τα ζητήματα αυτών των ε, μειονοτήτων πολύ καταπιεστικές συνθήκες, συνθήκες μάλιστα σε σχέση και με τα στρατόπεδα αυτά στους καταβλισμούς που απαγορεύονται από το ίδιο το Σύνταγμα της Κίνας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ξέρουμε ότι είναι αναπαλωτρίωτα, ξέρουμε ότι είναι αδιέρετα, αυτό ισχύει και για την Κίνα και δεν ε, μπορούμε να επιτρέψουμε στην Κίνα επειδή έχει αναλάβει μεγάλη οικονομική και πολιτική ισχύ να αγνοεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να το υπενθυμίζουμε πάντοτε στην Κίνα. Σας ευχαριστούμε κύριε Λάινεν. Επόμενη ομιλήτρια για δύο λεπτά, κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος που επισημαίνει μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες στην Κίνα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το επισημαίνουμε. Είναι απαράδεκτη κατάσταση ε, στην Κίνα για τις μειονότητες αυτές. Η Κίνα, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, με πλούσια παράδοση πνευματική, ε, δυστυχώς καταπατά τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων. Καταφέραμε πάντως να καταλήξουμε σε συμφωνία και ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους γιατί παρά τις διαφορές των απόψεων καταλήξαμε σε συνένεση. Είναι σημαντικό να αποφαινόμαστε με νέα φωνή για τα θέματα της Κίνας. Να ζητήσουμε από την Κίνα να εφαρμόσει το ίδιο της το Σύνταγμα που προβλέπει σεβασμό της ανεξιθρησκείας. Αντίθετα όμως, οι, οι χριστιανοί διώκονται, εκκλησίες ε, καταστρέφονται, θρησκευτικοί ηγέτες ε, συλλαμβάνονται και Φαίνεται ότι γίνεται δίωξη και εθνοτικών μειονοτήτων, όπως των Οιγούρων ή των Θιβετιανών. Έχουν πέσει και αυτοί θύματα του συστήματος ε, στρατοπέδου συγκέντρωσης ε, και ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Ζητούμε άμεση απελευθέρωση όλων των ε, κρατουμένων στα στρατόπεδα αυτά. Επίσης, σίγουροι, οικονομολόγος και ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, ε, από τους Ιγούρους έχουν φυλακιστεί. Θα απελευθερωθούν όπως ο Νέρσο Μαντέλα και ο Βάζελα Χάβελ στην εποχή τους. Ζητούμε να επιβληθούν κυρώσεις σε όσους συμμετείχαν στην καταστολή στην επαρχία Σιντζάνγκ. Και συμφωνούμε και ζητούμε να σταλεί ανεξάρτητη αντιπροσωπεία για να διερευνήσει τις διώξεις στην Επιτροπή Σιντζάνγκ. Σίγουρα ο σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα δεν είναι υψηλό και γι' αυτό θα πρέπει να επιμένουμε. Η διάσκεψη κορυφή με την Κίνα τον Απρίλιο μα άφησε μια πικρή γεύση. Ε, γιατί στο διάλογο μα με το γίγαντα τη την Κίνα, ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικές και θρησκευτικέ μειονότητες δυστυχώ αποσιοποιήθηκε. Και παρόλο που στη διακήρυξη αναφέρεται δειλά ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, αδιέρετα, άρρηκτα συνδεδεμένα αναφέρεται, παρόλα αυτά έχουμε πολύ ανησυχητικές πιέσει στην ελευθερία των ε, μειονοτήτων, είτε κατά των ουηγούρων, είτε με καταστροφές εκκλησιών, είτε με βασανιστήρια ή καταστολές υπό το πρόσημα της κινεζοποίησης, ε, οι καταπιέσεις στην αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ, ε, είχαμε αδιανόητες ε, καταστολές της βάρος των Θιβετιανών. Μάλιστα εμποδίστηκαν διεθνείς δημοσιογράφοι ή παρατηρητές να μεταβούν στην, στην περιοχή, στην αυτόνομη περιοχή του Θιβέτ κάτι που το στυλιτεύσαμε με τον Τόμας Μαν. Το θέμα δεν είναι να δίνουμε μόνο μαθήματα. Είναι αδιαπραγμάτευτα τα ανθρώπινα δικαιώματα Επίσης, ε, δράτω με τι ευκαιρίες και αυτή τη τελευταία ε, ομιλία μου στην Ολομέλεια μετά από τρει διαδοχικέ θητείε, να ευχαριστήσω θερμότατα όλου του συναδέλφου ο... τις καταπληκτικές με τι οποίε συνεργάστηκα και όλο το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία δεκαπενταετία που πέρασα υπηρετώντα την Ευρώπη και που ήταν πολύ πλούσια χάρη στη συνεργασία με όλου αυτού του ανθρώπου. Έδωσα τη μάχη μου υπέρ του ανθρωπισμού και τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Εύχομαι και σε εσά καλή τύχη. Ο κύριος Κέλα με έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε. Είναι από τα τελευταία κατεπήγοντα που εξετάζουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Το μήνυμα όμως είναι κατεπήγον. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η θρησκευτική ελευθερία ε, είναι αντικείμενο καταπίεσης ε, στην Κίνα. Και μάλιστα θρησκευτικές ομάδες ε, υπόκειται σε πολύ αυστηρό έλεγχο. Η ανεξιθρησκεία δεν υπάρχει και 7.000 ε, σταυροί ε, κατέβηκαν από εκκλησίες τον τελευταίο χρόνο. Φαίνεται ότι το κομμουνιστικό κινέζικο καθεστώς θέλει να ασκήσει έλεγχο στις θρησκευτικές πεπιθήσεις και στις εκκλησίες. Επίσης, ανησυχητική είναι η κατάσταση εθνωτικών μειονοτήτων, κυρίως των Ουγγούρων και των Θηβετιανών. Αλλά δεν αρκεί να εκφράζουμε απλώς την ανησυχία μας. Αυτό που επήγει είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα κράτη-μέλη να τηρήσουν την υποχρέωσή τους και να προωθήσουν την ε, δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις εξωτερικές μας σχέσεις, χωρίς καμία εξαίρεση. Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Δεν θα πρέπει να ικανοποιούμε με μια παρήθμιση των κρουσμάτων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί η, η καταστολή στις επαρχές Σιγκιάγκα είναι ε, τρομερή. Θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσει στα υψηλά στελέχη του Κινέζικου κόμματο που είναι υπέτεια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Λυπάμαι που σα κόβω, αλλά πρέπει να τηρήσουμε κάποια πειθαρχία εδώ. Από εδώ και πέρα θα επιμείνω πραγματικά στην πιστή τήρηση του χρόνου αγόρευση. Δεν έχω άλλη επιλογή δυστυχώ. Για ένα λεπτό και για ένα λεπτό και μόνο. Ο κ. Βίντεν Χόλτσερ. Προχωρούν οι σχέσεις μας με την Κίνα και διαμορφώνονται και θα διαμορφώσουν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όρους ε, οικονομικούς αλλά και κοινωνικούς. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε έναν εταίρο στο πρόσωπο της Κίνας αξιόπιστο και ε, στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε δυστυχώς ότι είναι συχνές οι παραβιάσεις ελευθερίας της ε, έκφρασης, της γνώμης και των ελευθεριών. Ιδιαίτερα μας ανησυχεί η συστηματική παραβίαση των ελευθεριών των θρησκευτικών και αυτό αφορά τους πάντες, χριστιανούς, μουσουλμάνους, βουδιστές. Αυτή τη στιγμή οι μουσουλμάνοι Ουιγούροι στην περιοχή Σιντζιάνγκ έχουν αντιμετωπίσει μια κατάσταση αβίωτη με πολύ σκληρά μέτρα καταστολής. Πρέπει να σταματήσει τώρα και μόνο να σταματήσει τώρα μπορούμε να εμποδίσουμε να μετατραπεί αυτό σε μια παράδοση. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η καταστολή των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων δεν είναι κάτι το καινούριο στην Κίνα, αλλά πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια σκληροπυρηνική στρατηγική στην Σινγκζιάνγκ και πολλές μειονότητες έχουν αναγκαστεί να ε, μπουν σε καταβλισμούς για συμμόρφωση και ε, πρόσφατα μα κάλεσαν να επισκεφθούμε την περιοχή, αλλά τέτοια ε, επίσκεψη θα είχε νόημα αν υπήρχε ελεύθερη είσοδο σε αυτούς τους καταβλισμούς. Επίσης, ε, καλό τον ειδικό πεσταλμένο της Ένωση να ζητήσει για τα, την ανεξιθρησκεία να ζητήσει άδεια για να επισκεφθεί την Κίνα. Επίσης θέλουμε να ζητήσουμε πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου που έχει υποχωρήσει δυστυχώς υπό τον πρόεδρο ΣΥ. Σάκε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε πρόσωπε συνάδελφοι. Και την ώρα που μιλάμε, πολλά εκατομμύρια κόσμος έχουν ε, περιοριστεί σε καταβλισμούς που έχουν περιγραφεί από τον ΟΗΕ ως ζώνες ε, χωρίς δικαιώματα. Εμείς ε, δεν θα πρέπει να τυφλωνόμαστε από, την, από το όραμα κέρδους όταν η εταιρείε μα συνεργάζονται με τις κινέζικες. Υπάρχουν διάφορα μέτρα που χρησιμοποιούνται ε, υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων της ε, ιδιωτικής ζωής για αυτόν τον κόσμο. Η νέα στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας είναι ευπρόσδεκτη, όμως θα πρέπει ως πρώτο άξονα να έχει την αντιμετώπιση κοινών θεμάτων, θεμάτων μάλλον κοινών ενδιαφέροντος και αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι πρώτο στο κατάλογο. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από απλά λόγια, ε, Επίσης πιστεύω πως είναι πήγον να εξετάσουμε τον εμπορική αγορά της τεχνολογίας εποπτείας. Ευχαριστώ. Σολέ. Η Κίνα και η καταστολή των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων είναι το τέλειο παράδειγμα της ανάγκης η Ευρωπαϊκή Ένωση να κρατά, δείχνει συνέπεια και δύναμη όταν υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και αν μεγάλος και δυνατός ο ετερός ε, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι καθολικά και οι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι σοβαρότερε ή λιγότερο σοβαρέ ανάλογα με τη χώρα ε, και την οικονομική τη ή πολιτική τη ε, ισχύ. Οπουδήποτε και αν συμβαίνουν οι παραβιάσει, πρέπει εμεί να το καταγγέλουμε και να ενεργούμε αναλόγω. Ε, Δυστυχώ, οι εθνοτικέ, οι θρησκευτικέ και οι γλωσσικέ μειονότητε πιέζονται σε ολόκληρο τον κόσμο ακριβώ επειδή θέλουν να διατηρήσουν την ταυτότητά του. Δεν θα πρέπει να ε, ε, εθελοτυφλούμε ενώπιον τέτοιων ε, πολιτικών. Οι χώρε που επιβάλλουν μια ταυτότητα, μια γλώσσα, μια, ένα πολιτισμό μπορεί να είναι μεγάλε, αλλά δεν είναι δίκαιε ούτε σωστέ. Ευχαριστώ, κύριο Σπρέντα. Ευχαριστώ. Η ομάδα μας σε ολόκληρε προσπάθησε να φέρει ω κατεπήγον το θέμα της Κίνα. και χαίρομαι που επιτέλους, έστω και στην τελευταία ε, σύνοδο τη κοινοβουλευτική μα θητεία, έχουμε ως κατεπήγον αυτό το θέμα για την Κίνα. Έχουμε επανειλημμένω δηλώσει ότι οι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα είναι κατάφορε. Και μάλιστα αναφέρθηκαν ε, ε, προβλήματα. 10 εκατομμύρια Καζάχοι και Ουιγούροι που βρίσκονται σε στρατόπεδα κράτηση και αναμόρφωσης στην επαρχία Σιντζάνγκ. Οι Θιβετιανοί που εξαφανίζονται, ε, βασανιστήρια, ε, καταδίκες χωρίς δίκες, καταδίωξη των θρησκευτικών μειονοτήτων, κυρίως κατά των χριστιανών, καταδεφαρίζονται εκκλησίες, καταστρέφονται σπίτια, φυλακίζονται ιερείς. Όλα αυτά δείχνουν μια πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που θέλει να μεταδώσει ο CG Πινγκ ε, στον κόσμο. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την τελευταία μου παρέμβαση, να ευχαριστήσω την είπατε εκπρόσωπο για το έργο που επιτέλεσε την τελευταία πενταετία και στι εξωτερικέ υποθέσει και σε αυτό το σημαντικό τμήμα, σε αυτή τη σημαντική συνιστόσα της, ε, των εξωτερικών υποθέσεων, τα ανθρώπινα δικαιώματα δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πεμπτουσία τη Ευρώπη το ίδιο ε, και η ποιοτική τη διαφορά. Θα πρέπει να συνεχίσουμε το δρόμο. Επίση, θα ήθελα να πω ε, στο επανειδή στου συναδέλφου, ή μάλλον αντίο, γιατί φεύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, δεν θα Ξανακατεβαλα αλλά χαίρομαι που διατέλεσε Ευρωβουλευτής, γιατί είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό θεσμικό όργανο. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Καλή τυχή. Και σας φαντάζομαι κάποια στιγμή στο μέλλον θα διασταυρωθούν ίσως και πάλι δρόμοι μας. Ο κύριος Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε, εγώ δεν θα σας χαιρετήσω, θα Είμαι και πάλι υποψήφιο στι ευρωεκλογέ από τη Βαρσοβία και είμαι αισιόδοξο. Αλλά σήμερα έχουμε ένα πολύ πιο σοβαρό θέμα από τη συμμετοχή, τη δική μου την προσωπική συμμετοχή σε ευρωεκλογέ. Εδώ μιλούμε για τα δικαιώματα των χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων στην λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων και χαίρομαι που επιτέλου το συζητούμε. Εγώ είμαι υπέρ τη ανάπτυξη των σχέσεων μα με την Κίνα, υπέρ των οικονομικών σχέσεων γιατί πιστεύω ότι θα είναι εποφέλής αλλά δεν μπορούν οι οικονομικές σχέσεις να, γίνονται εις βάρος ε, των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν θα πρέπει να ε, είναι το αντίτιμο τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οικονομικά πλεονεκτήματα που δρέπουμε και δεν θα πρέπει να είναι το τίμημα της σιωπής μας ή της εθελοτυφλίας. Είχαμε συζητήσει ε, πρόσφατα τους Ουγγούρους ε, και ανέφερε και το θέμα των χριστιανών. Ελπίζω να μην έχουμε στο μέλλον ίδιο μέλλον για τους χριστιανούς με τις καταδιάψεις των Ουιγούρων. Πριν ε, από ένα μήνα είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Δαλάη Λάμα. Έχουν περάσει 30 χρόνια που κατέχουν την περιοχή του Θιβέτ οι Κινέζοι, οι Τιβετιανοί βγήκαν στους δρόμους και στην Ινδία ακόμα για να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν τη διαφύλαξη της κουλτούρας και της θρησκείας τους. Είμαστε στην ομάδα την διακομματική για το Θιβέτ και καλούμε τις κινέζικες αρχές να ε, αλλάξουν συμπεριφορά γιατί διαρκώς βλέπουμε ότι επιδεινώνεται η κατάσταση στο Θιβέτ με ε, όλο και πιο σκληρή αντιμετώπιση των Θηβετιανών. Είναι η τελευταία μου ομιλία εδώ σήμερα, ύστερα από 25 χρόνια. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ρίσπεκ, τον κύριο Πρέντα, Τούνμπερκ και πολλούς άλλους συναδέλφους, χάρη στους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν και παραμένει η φωνή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάν, ευχαριστώ και εμείς το καλύτερο όπου σας οδηγήσει ο δρόμος σας, ο κύριος Γιούρεκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση των, χριστιανών στην Κίνα εξακολουθεί να είναι δραματική. Έχουμε πολλαπλά ε, θέματα καταδίωξης. Ε, για παράδειγμα, ε, παρεμπόδιση της θρησκευτική ε, ε, εκπαίδευσης σε πολλές επαρχίες. Επίσης, έχουμε φυλάξει επισκόπων και ιερέων σε πολλές επαρχίες μάλιστα πριν από πολλούς α, μήνες μας έκοψε το κόδωνα του κινδύνου ο επίσκοπος Ζεν. Θα πρέπει να α, στυλιτεύσουμε αυτή την κατάσταση, να δείξουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα και σίγουρα στη διπλωματία έχουν σημασία οι χειρονομίες γιατί θα πρέπει να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η χριστιανική κοινότητα, να έχουμε επαφές με τη χριστιανική κοινότητα. Δεν θα πρέπει να σταχθούμε υπέρ της αδιαφωνίας και της ε, άκαρδης ε, ουδετερότητας. Θα πρέπει η Κίνα να αντιληφθεί ότι η στάση της απέναντι στους ε, χριστιανούς θα επηρεάσει τις διμερείς μας σχέσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέτμαν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, η κατάσταση των, θρησκευτικών, των εθνοτικών μειονοτήτων στην Κίνα και των θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδίω των χριστιανών, Ιγούρων και Καζάχων, είναι ανησυχητική και μάλιστα αναφέρθηκε ως πολιτική ανθρωποκτονία αυτή η δίωξη που κάνει η Κίνα προς εθνοτικές και θρησκευτικές κοινότητες καταπατά τα συνταγματικά τους δικαιώματα ε, και την ελευθερία του συνέρχεσαι και του συνεταιρίζεστε. Ιδιαίτερα ενισχυτική είναι η κατάσταση των Ουιγούρων που έχουν φυλακιστεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τα παιδιά διαχωρίζονται από την οικογένειά τους και υφίσταται μια πολιτική κατήχηση. Ε, και μάλιστα η κατάσταση στην Κίνα δεν αλλάζει, παρόλο που το έχουμε επισημάνει επανειλημμένω. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσει ή να να ε, σε αυτέ τι πρακτικέ. Θα πρέπει να ζητήσουμε άμεση, ε, άμεσο κλείσιμο των, των στρατοπέδων, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων και να επιστρέψουν τα παιδιά στι οικογένειέ του. Ο κύριος Δεμεσμέκερ, για ένα λεπτό. Έχουμε ε, ενημερωθεί για ε, μαζικές ε, συλλήψεις και εγκλισμούς στην Κίνα και θυμάμαι τα πρώτα λόγια ενός γερμανικού τραγουδιού δεν μπορούμε να φυλακίσουμε την σκέψη και αυτό κάνει ακριβώς η Κίνα ότι λίγο αποκλίνει καταστέλλεται βία είναι μια στρατηγική πολύ ρονταρισμένη, μια ε, ε, ήπια εικόνα προς τα έξω ε, που βασίζεται βασικά στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στο εσωτερικό προσπαθούν να θεραπεύσουν από την αρρώστια όσους λίγο αποκλίνουν από τα απαραίτητα. Ε, είναι αμήλικτος ο κρατικός μηχανισμός. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να σταματήσει την καταστολή ε, η κινέζικη κυβέρνηση. Γιατί κύριε Πρόεδρε η ε, σκέψη είναι ελεύθερη και καμιά αρχή δεν μπορεί να την περιορίσει. Ευχαριστούμε κύριε Ντεμεσμάκερ. Τώρα ο συνάδελφος Βόμποντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Σήμερα Φόρεσα επίτηδες κόκκινη γραβάτα. Ε, δεν είναι μόνο εκείνοι που είναι, ε, ε, καταστρέφονται οι εκκλησίες, κατάσχονται οι βίβλοι και ε, ε, το ίμιση των Κινέζων χριστιανών ε, διώκεται. Πρέπει να πηγαίνουν και να δίνουν το παρόν στα αστυνομικά τμήματα σαν να είναι εγκληματίε και άνθρωποι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στις θρησκευτικέ λειτουργίες. Έχουμε ήδη καταδικάσει τις διακρίσεις κατά των χριστιανών στην Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της θα πρέπει να αποκομίσουν τα συμπεράσματα από αυτές τις διώξεις οποτεδήποτε ζητούν άσυλο Κινέζοι πολίτες στην Ευρώπη. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν είμαστε Ευρώπη που να βασίζεται στο σεβασμό των ε, αξιών μας. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την, ε, την το ΚΑΤΣΔΙ, ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ. Κυρία Μογκερίνη, παρά το ότι ο πρόεδρος Τζινπίνγκ προσπαθεί να δώσει μια εικόνα συγχρονιστική για την Κίνα, η πραγματικότητα λέει ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι διώξεις κατά των εθνοτικών μειονοτήτων. Απέναντι σε αυτή τη δράση, τα Υπάρχουν συστήματα ε, μαζικής εποπτείας ε, που φέρουν οι ουγούροι ε, και κλείνονται σε καταβλισμούς αναμόρφωσης στις διάφορες περιφέρειες είναι μεγάλες εκστρατείες ρατσισμού και καταπίεσης. Οι συμφωνίες που υπογράφονται ανάμεσα στην Κίνα και διάφορες χώρες Ένωσης θα πρέπει να επιτρέψουν το χρήμα να μας τυφλώσει απέναντι στις δημοκρατικές μας αξίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ποσπίσιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για το κατεπήγον ψήφισμα για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, που είναι καταστροφική. Αναφέρθηκαν οι Θηβετιανοί, οι Ιγούροι, οι διώξει των χριστιανών. Και μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πράγας πρόσφατα ε, Υποδεχθήκαμε τον εξόριστο Θιβετιανό Πρωθυπουργό και μας ενημέρωσε για την κατάσταση στην αυτόνομη περιφέρεια του, του Θιβέτ και την πραγματική δίωξη και τις μαζικές δολοφονίες Θιβετιανών. Ε, είναι καταστροφική η κατάσταση, τραγική. Θα πρέπει λοιπόν ε, ε, να διατρανώσουμε την φωνή μας υπέρ της υπερασπισής. Εμείς χρειάστηκε συμβολικά να, ε, να υψώσουμε τη σημαία του Θιβέτ στο Δημαρχείο της Πράγας ως ένδειξη συμπαράστασης. Νομίζω ότι είναι ηθικό μας καθήκον να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την υποστήριξή μου στην, ε, στο ψηφίσμα, όπως και οι συνάδελφοι. Η κατάσταση είναι φρικτή, έρχονται πολύ ανησυχητικά μηνύματα, ιδιαίτερα από την περιοχή των Ουιγούρων και θα πρέπει όλοι μας να καταδικάσουμε απερίφραστα τα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει να ε, απευθύνουμε έκκληση για το να στον αποφυλακισμό εκείνων οι οποίοι κρατούνται και να καλέσουμε την Κίνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Δεσμεύσεις που θα πρέπει να υπενθυμίζουμε σε κάθε συνάντηση με τους κοινούς ομολογούς μας και όποτε βρισκόμαστε σε επίσκεψη στην Κίνα ε, δεν πρέπει να φοβούμαστε να μιλήσουμε για τα προβλήματα αυτά γιατί έχω μερικές φορές την εντύπωση πως για λόγους διπλωματίας αποφεύγουμε την αναφορά στα προβλήματα αυτά. Μα αν ευρωβουλευτέ δεν μπορούν να μιλούν, ποιο τότε. Ας το έχουμε αυτό υπόψη και για την επόμενη θητεία. Η κατάσταση στην Κίνα είναι καταστροφική και με το να κλείνουμε το στόμα δεν πρόκειται να την ε, λύσουμε. Ο κύριος Λόπες. Γινόμαστε για άλλη μια φορά μάρτυρες στην υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και στην εργαλειοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως τρόπο τρόπος επέμβασης ε, στις κυρίαρχες χώρες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι γνώμονας ούτε δικαιούται να μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί δείχνει συνενοχή με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία και επιτίθεται ίδια σε άλλες χώρες. Οπότε πώς μπορεί να ισχυρίζεται ότι προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, και δεν θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε εμείς με την πολιτική αντιπαράθεση την παράθεση του Τραμπ απέναντι στην Κίνα. Ε, είμαστε υπέρ ε, της, των δικαιωμάτων και είμαστε υπέρ της συνεργασίας με τρίτες χώρες με σεβασμό της εθνικής του κυριαρχίας και είμαστε κατά της παρέμβασης, όπως φαίνεται και στο χάρτη των Ηνωμένων, των Ηνωμένων Εθνών. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε τα πορτογαλικά συμφέροντα στις σχέσεις με την Κίνα με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αυχόζερ, για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα, μια αυτοκρατορία, αυτοκρατορία του μέσου η αυτοκρατορία αυτή το 19ο αιώνα το καταστρέψαμε εμείς με την πολιτική της κανονιοφόρου. Τους αναγκάσαμε να ανοίξουν τα σύνορα, να βάλουν όπιο. Μετά τον ιδεολογικό μαρξισμό που επίσης συνεισέφερε στην πλήρη καταστροφή της χώρας. Παρ' όλα αυτά η χώρα αυτή ανοικοδομήθηκε. Ανοικοδομήθηκε χάρη σε μια φιλελεύθερη πολιτική που την έχει οργανώσει το κράτος και προσανατολίσει προς την οικονομική ανάπτυξη. Από πού και ως πού τώρα εμείς θα πάμε να δίνουμε μαθήματα στην Κίνα. Ωραία, το Θιβέ, τη Χριστιανή, συμφωνώ. Αλλά από πού και ως πού, εμείς που κάναμε πόλεμο για την ε, Αλσατία και δύο παγκόσμιους πολέμους, εμείς που κάναμε θρησκευτικού πολέμους, ποιοι είμαστε που σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για λόγους πολιτικής πίσω από τη θρησκεία. Εντάξει, δεν λέω να την επικρίνουμε την Κίνα, αλλά μήπως θα ήταν καλύτερο για το Κοινοβούλιο να τηρήσει το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σας ευχαριστώ. Κυρία Αντιπρόεδρε, κυρία Μογκερίνη, έχετε το λόγο αφού τελείωσε η διαδικασία αΐ. Παρακαλώ. Uh, uh, σας ευχαριστώ. Όπως ε, είπατε κάποιοι, ε, Σήμερα είναι η 25η επέτειο της νέας στρατηγική για την ε, Κίνα. Τώρα έχουμε μια νέα σχέση με την Κίνα βεβαίω πιο έντονη αλλά και πιο ειλικρινή και ανοιχτή. Βασισμένη σε λόγια σταράτα, ξεκάθαρα συμφέροντα επίσης. Αλλά βεβαίω, ε, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Προσπαθούμε να υπάρξει κάποια συνέπεια στην προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών οργάνων. Εδώ πέρα λοιπόν θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση σε όλους σας. Εδώ εκπροσωπείτε τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και πολιτικές ομάδες και εθνικά κόμματα. Πολλοί από σας μιλήσατε, ε, είπατε λογικά και σημαντικά πράγματα, οι περισσότεροι θα έλεγα, ανήκετε και σε κόμματα που έχουν ε, ευθύνες κυβερνητικές. Θα ήθελα λοιπόν αυτά τα καθαρά λόγια να τα πείτε και στις δικές σας κυβερνήσεις όταν ε, πρέπει η εταίροι της Κίνας να είναι τόσο ξεκάθαρη όσο είναι και τα θεσμικά όργανα. Όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και εγώ έχουμε απευθυνθεί στους κορυφαίους Κινέζους ηγέτες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ότι για τους Ευρωπαίους τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα. Αντιθέτως, είναι εξίσου σημαντικά, αν όχι πιο σημαντικά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να στέλνουμε συνεπώς και συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Το Κοινοβούλιο, και σας ευχαριστώ γι' αυτό, η Κομισιόν, το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη στις διμερείς του σχέσεις με την Κίνα. Η Κίνα έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στο θέμα οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά η γενικότερη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρατε, συνεχίζει να επιδεινώνεται. Ειδικά όσον αφορά πολιτικά δικαιώματα. Οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων συλλαμβάνονται, θεμελιώδεις ελευθερίες παραβιάζονται. Έχουμε δει όλοι τις εκθέσεις για την κατάσταση στην Τζιντσάνγκ, τα στρατόπεδα πολιτικής επανεκπαίδευσης ε, που αφορούν διάφορες μειονότητες, ε, μαζικές ε, παρακολουθήσεις, περιορισμοί των ταξιδιών και κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις επίσης είναι ζητήματα που έχουμε θίξει και στις διμερείς επαφές και στον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, ε, να απευθυνθώ και στην άλλη πλευρά, ε, για πρώτη φορά προσκαλέσαμε και τους υπουργούς ε, εξωτερικών της Κίνας και με χαρά είδα ότι τα κράτη-μέλη έστειλαν μηνύματα σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών για ζητήματα που είναι σημαντικά για τον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά επίσης θίξαμε αυτά τα ζητήματα και στο πλαίσιο της πολιτικής αντιτρομοκρατίας. Και το τονίζω αυτό, πόσο σημαντικό είναι για εμάς να είμαστε συνεπείς όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί Ίσως υπάρχει η τάση στους συνομιλητές μας, όχι μόνο για την Κίνα, και με άλλους, να σκεφτούν ότι ε, τα θεσμικά όργανα ασχολούνται με αυτά και τα κράτη-μέλη δεν ασχολούνται. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε συνεπείς στα μηνύματα που στέλνουμε. Και νομίζω ότι ίσως ε, σε αυτό το μέτωπο σημειώνεται κάποια πρόοδος ε, απέναντι στους Κινέζους συνομιλητές μας, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτά είναι σημαντικά για κάθε Ευρωπαίο, για κάθε κράτος μέλος, για όλες τις πολιτικές οικογένειες αυτού του Κοινοβουλίου. Δράδομαι και πάλι τη ευκαιρία δημοσίως να ζητήσω από την Κίνα να επιτρέψει πρόσβαση ανεξαρτήτων παρατηρητών στο Xinjiang και να προσθέσω και εγώ την φωνή μου στην έκκληση για ανεξάρτητους παρατηρητές από τον ΟΗΕ και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ανεξιθρησκεία συχνά παραβιάζεται στο Θιβέτ και υπάρχει επίσης, υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση στην ε, περιοχή αυτή για να υπάρξει αμοιβαία πρόσβαση για Ευρωπαίους δημοσιογράφους και διπλωμάτες και τις οικογένειές τους. Τα τόνισα αυτά και στην Σύνοδο Κορυφής, ε, τα έχω λοιπόν πει και δημόσια και ιδιωτικά. Συζητήσαμε την κατάσταση στο Σινζιάνγκ, στο Θιβέτ, την ανεξιθρησκεία και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και στον τελευταίο διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων θέσαμε το ζήτημα του μειωμένου χώρου της κοινωνίας των πολιτών και το νομικό πλαίσιο και την αυτονομία του Χονγκ Κόνγκ επίσης ε, θέσαμε. Ε, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, καμιά φορά είναι πάρα πολύ δύσκολα αλλά το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε με τους Κινέζους εταίρου μας είναι να είμαστε σε επαφή, να είμαστε ξεκάθαροι στα μηνύματα που στέλνουμε και να προωθήσουμε μια αλλαγή πορεία στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλάμε στους Κινέζους με σεβασμό αλλά και ξεκάθαρα. Καμία άλλη παγκόσμια δύναμη δεν το κάνει αυτό. Η παγκόσμια τάση για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική, τα έχουμε πει αυτά εντός Τη αιθούση αυτής πολλές φορέ. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένας λόγος παραπάνω για να μην τα παρατήσουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ω Ευρωπαίοι να σταματήσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιλάμε για την Κίνα, αλλά και ανά τον κόσμο. Και αναμένω τι επόμενε συζητήσει μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μογκερίνη, έχουμε έξι προτάσεις ψηφίσματος από τους πράσινους, την ΚΟΕ, το ΙΣΙΕΡΑ, τους σοσιαλιστές και την ΑΛΔΕ. Ε, ολοκληρώνεται έτσι η συζήτηση για αυτό το θέμα και η ψηφοφορία θα γίνει αργότερα σήμερα. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το Καμερούν. Εδώ έχουμε πέντε συντάκτες ψηφίσματος και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στον κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Καμερούνου. Υπάρχουν πάρα πολλές απειλές εσωτερικές και εξωτερικές και υπάρχει μια αυταρχική διάθεση στη χώρα με πολλούς περιορισμούς. Ο Μόρις, Κάμπτο και 200 ακτιβιστές του κόμματός του της αντιπολίτευσης συνελήφθηκαν ε, μετά από τις εκλογές του 2018. Και αυτό είναι το τελευταίο συμβάν υπάρχουν ε, αντιδράσεις, αντιστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Το Καμερούν είναι φυσικά ένας εταίρος πολύ σημαντικός για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του Μποκοχαράμ για παράδειγμα, που δραστηριοτείται κυρίως στο βορρά της χώρας από το 2012, αλλά υπάρχουν πολλές ανησυχίες για την κατάχρηση που γίνεται στον αντιτρομικό νόμο του 2014. Ακούμε ότι γίνονται εξοδικαστικές δολοφονίες, από τρομοκρατικέ οργανώσει και ακόμα και εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να φροντίζουν για τη συμμόρφωση προ τον νόμο θέτουν σε κίνδυνο του πολίτε. Συγχρόνω, η απάντηση τη κυβέρνηση, στις διαμαρτυρίε των Αγγλόφωνων όπου είναι μια ε, μειοψηφία βορειοδυτικά και, και είναι επίση κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο Ουρμπάν Κρέσπο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στο Καμερούν ο στρατός από ό,τι φαίνεται παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε μεγάλο βαθμό σε βάρος του κόσμου. Κατηγορούνται επίσης ότι αυθαίρετα συλλαμβάνουν διαδηλωτές οι οποίοι ειρηνικά ε, διαδηλώνουν. Στις αγγλόφωνες περιοχές ο στρατός πυροβολεί από ελικόπτερο με αποτέλεσμα εκατοντάδες τραυματίες και πολλούς νεκρούς. Εξοδικαστικά επίσης διώκεται κόσμος. Και υπάρχουν και βίντεο τα οποία δείχνουν πώς στρατιωτικοί από το Καμερούν δολοφόνησαν δύο γυναίκες και τα μωρά τους επειδή υποψιάστηκαν ότι ανήκουν στον Πόκο Χαράν. Χώρε όπω η Ισπανία πουλάνε όπλα στη χώρα. Παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται από το Συμβούλιο ήδη από το 2008 με κοινή θέση. Παρ' όλα αυτά δεν γίνεται τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη προσφέρουν στρατιωτική εκπαίδευση και λογιστική στήριξη, εκατάρτιση, στρατιωτικό εξοπλισμό και ασφάλεια στο Καμερούν. Κάτι το οποίο έχουν σταματήσει να κάνουν άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, ακριβώς γιατί γίνεται κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Καμερούν. Απαιτούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει αυτή η στήριξη, η πώληση όπλων και εξοπλισμού στο Καμερούν όσο δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσο πρόκειται μόνο για λόγια και όχι για πράξεις. Είμαστε συνένοχοι κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζελιάνα Ζόφκο. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμη κυρία Μοκερίνη, ε, πρόεδρε, και την τελευταία μέρα της Συνόδου της θητείας μας παραμένουμε προσιλωμένοι στον αγώνα για ένα δίκαιο και ανθρώπινο κόσμο. Σήμερα αυτό μας φαίνει στο Καμερούν. Πολλοί παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εκθέσεις τους δηλώνουν την υπερβολική βία από πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας και τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πολιτών. Πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης και ο ηγέτης του κόμματος Μωρίς Κάμπτο ε, διώκονται και φυλακίζονται. Οι αρχές επίσης της χώρας επανειλημμένα έχουν περιστέλει ε, τα δικαιώματα και τη ελευθερία της έκφρασης. Αυτό όλα είναι αντίθετα με τις δικές μας αρχές και αξίες τις οποίες προωθούμε και διεθνώς. Συνεπώς, θα πρέπει να δράσουμε αγαπητοί συνάδελφοι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ε, καλέσουμε τις κρατικές αρχές ε, να αφήσουν αμέσως ελεύθερους, ανεφόρων, όλους τους πολιτικούς αντιπάλους και όποιους άλλους πολίτες ε, κρατούνται για λόγους πολιτικούς και μόνο. Θα πρέπει να καταδικάσουμε την έντονη καταστολή και τη βία και να προωθηθούν ελεύθερες και ανεξάρτητες έρευνες η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να κάνει τώρα. Μπορεί να κάνει τη διαφορά, να εκμεταλλευτεί την πολιτική πίεση ε, που δίνουμε από το πρόγραμμα αναπτυξιακής βοήθειας για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Καμερούν. Επίσης, θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως δώσουμε τεχνική βοήθεια και πολιτική υποστήριξη ε, βάσει της εμπειρίας που έχουμε σε άλλες εμπόλεμες σειράξεις και ε, από την αναπτυξιακή βοήθεια για να ενισχύσουμε τη δημοκρατική κοινωνία στο Καμερούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, το παρόν ψήφισμα είναι προ όφελο όλων των πολιτών του Καμερούν και αξίζει την υποστήριξή σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Γιούντιτ Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, εκλογές έγιναν τον Οκτώβριο του 2018 στο Καμερούν και ο πρόεδρος Πολ Μπίγια εξελέγει εκ νέου ο οποίο κυβερνάει από το 1982 κατά τα άλλα. Μα πώς είναι δυνατόν. Και δεν είναι απορία άξιο που διαδηλώνει ο κόσμος και διαμαρτύρεται. Αυτό είναι ο πυρήνας του ψηφίσματος. Να πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον Πολ Μπιγιά άφησε ελεύθερο το Μωρίς Κάμπτο και τους δικούς του. Η δημοκρατική διαμαρτυρία ανήκει σε μια χώρα. Γιατί ε, δικάζονται σε στρατοδικεία οι πολίτες. Οι πολίτες δεν έχουν καμιά δουλειά στα ε, στρατοδικεία. Και γίνονται διακρίσει ει βάρο ανθρώπων που μιλούν διαφορετικέ γλώσσε. Θα πρέπει να τα ακούμε και αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν ασχολείται πολύ συχνά με το Καμερούν. Καλό είναι που έχουμε εστιάσει σήμερα την προσοχή μα και την κατάσταση στα χέρια του έχει ο Πολ Μπιά, ο οποίο μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαργίτσε Σχάκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωποι, συνάδελφοι. Μετά τι εκλογέ που οδήγησαν σε πολλά ερωτηματικά στο Καμερούν, έγιναν ειρηνικέ διαμαρτυρίε και απεργίε, ε, τι οποίε ε, κατέστηλε έντονα η αστυνομία. Εκατοντάδε είναι νεκροί, εκατοντάδε χιλιάδε εκτοπισμένοι και οι ακτιβιστέ ε, συλλαμβάνονται και φυλακίζονται αντιτρομοκρατικοί νόμοι και βαριά μέτρα χρησιμοποιούνται για να πατάξουν αυτές τις διαμαρτυρίες. Ε, Έχουμε βασανιστήρια, ε, εξοδικαστικές ε, εκτελέσεις και διώξεις γενικότερα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα κλιμακώνονται. Καλούμε την κυβέρνηση της χώρας να σταματήσει αυτή τη δυσανάλογη χρήση βίας και να σέβεται τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών. Θα πρέπει να γίνουν έρευνες για τις κατηγορίες για υπερβολική βία στην πάταξη ε, των διαδηλώσεων. Θα πρέπει η Αφρικανική Ένωση να αναλάβει νευτικές συνομιλίες και να βοηθήσουμε και εμείς και να υποστηρίξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και όλοι οι εταίροι μας. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών έχει τώρα το λόγο ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε Μογκερίνη, είπατε εκπρόσωπο. Σε όλη την Αφρική κανείς δεν έχει παραμείνει στην εξουσία περισσότερα χρόνια από όσο ο Πολ μπήγε στο Καμερούν, άντε και στη Ζιμπάμπουε κάτι το οποίο έχει οδηγήσει σε μαζικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις μετά τις τελευταίες εκλογές. Και ο ηγέτης ε, της αντιπολίτευσης, ο Μωρίς Κάμπτο, έχει καταλήξει στη φυλακή με κατηγορίες που θα δικαστούν από στρατιωτικό δικαστήριο και θα είναι το αποτέλεσμα προφανώς η θανατική ποινή ή η σόβια. Οπότε πρέπει να σταματήσει αυτή η βία, αυτή η όχληση των ανθρώπων που διαμαρτύρονται. Πρέπει να υπάρχουν ελεύθερες εκλογές, μεταρρυθμίσεις και κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με την Αφρικανική Ένωση και τις Αφρικανικές χώρες να διαμεσολαβήσουν για να απελευθερωθεί όχι μόνο ο Μωρής Καμπτό αλλά και οι 200 άλλοι ακτιβιστές που συνελήφθησαν μαζί του και κρατούνται. Και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω απ' όλα να πάρει μέτρα για να έχουμε λιγότερη συνεργασία με το Καμερούν εφόσον αυτό δεν συμπεριφέρεται δημοκρατικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσαρνέτσκι έχει τώρα το λόγο εκ μέρους του ECR. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το ερώτημα γιατί ασχολούμαστε με το Καμερούν. Η χώρα αυτή είναι τόσο μακριά από την Ευρώπη. Έχει νόημα όμως. Γιατί είναι μια χώρα η οποία ήταν ε, κάποτε απικία μιας ευρωπαϊκής χώρας και η χώρα αυτή ε, η απικιοκρατική δύναμη δηλαδή είχε κερδίσει προφανώς από αυτή την υπόθεση και δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια στο Καμερούν. Και έχουμε το δικαίωμα λοιπόν να αναμένουμε η χώρα αυτή να πληρεί κάποιες ε, προϋποθέσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει η φωνή μας να είναι δυνατή και αλληλέγγυα. Μόνο έτσι θα ακουστεί στο Καμερούν και σε άλλες αφρικανικές χώρες που ε, έχουν εμπορικές σχέσεις ε, μαζί μας, αλλά ξεχνάνε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ιγνάσιο Κορά Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ το Κάμερουν είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει ταυτόχρονα πολλές βαριές ε, απειλές. Έχουμε την απειλή του Μπόκο Χαράμ, ένοπλη στάση των αγγλόφωνων που θέλουν να αποσχιστούν. Για όλα αυτά χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αυτά με δυσανάλογη χρήση πυρός. Ειδικά καταδικάζουμε έντονα τα βασανιστήρια, τους εξαφανισμένους, τις εξοδικαστικές εκτελέσεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας, κάτι το οποίο είναι ιδιαιτέρως βαρύτατο όταν ε, οι δυνάμεις ασφαλείας κρατούν ε, στην εξουσία έναν άνθρωπο από το 1982. Έχουμε ταυτόχρονα το κλείσιμο του διαδικτύου, φυλάξη πολιτικών αντιπάλων, πράγματα τα οποία ποτέ δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Αυτές λοιπόν είναι οι πιο σοβαρές απειλές που αντιμετωπίζει σήμερα το κομμένο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομάδα του ΕΝΕΦ. E Τον λόγο έχει η κυρία Μπίλντε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίξουμε το στρατό και τους πολίτες του Καμερούν οι οποίοι τα έχουν βάλει με τον Μπόκο Χαράμ. Αυτός ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας είναι κάτι πολύ σημαντικό και ξεπερνάει τα σύνορα του Καμερών. Έτσι λοιπόν ε, με τη συνεργασία που έχουμε με τις χώρες γύρω από την Σαχάρια πρέπει να δράσουμε περισσότερο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για χρόνια χιλιάδες πρόσφυγες από την Ιγυρία που προσπαθούν να αποφύγουν ακριβώς την τρομοκρατία στη χώρα τους έχουν φτάσει στο Καμερούν. Η χώρα αυτή είναι μια σταθερή χώρα σε μια περιοχή με πάρα πολλές εντάσεις. Οπότε δεν πρέπει να απλοποιούμε τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, οι διαφωνίες ανάμεσα στους αγγλόφωνους και τους γαλλόφωνους δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με ανταγωνισμό μεταξύ τους, έχει να κάνει με οικονομικά συμφέροντα. Στις αγγλόφωνες ε, περιοχές είναι που βρίσκονται οι δρογονάνθρακες και οι αρχές ε, βέβαια δεν ε, θέλουν να πάρουν εκείνη περισσότερα κέρδη από αυτά. Η κυβέρνηση του Καμερούν λοιπόν και η Επιτροπή για την Διγλωσία και, και την Ποικιλομορφία στον πολιτισμό είναι που πρέπει να φροντίσουν να πάψουν αυτές οι εντάσεις. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τα δικαστήρια, για τους καθηγητές, τους δίγλωσσους. Η κοινωνία με την ποικιλομορφία της δεν μπορεί να προχωρήσει κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όλοι πρέπει να έχουν τις ίδιες αξίες, τα ίδια σημεία αναφοράς και αγαπάνε την ίδια χώρα. Αυτό το Καμερούν πρέπει και εμείς να στηρίξουμε, χωρίς να μεροληπτούμε, χωρίς να αναμειγνιόμεθα και χωρίς να έχουμε δεύτερη σκέψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος, η κυρία Σεσίλ Κέγκα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Καμερούν έχει κυλήσει στην ε, βία. Η κυβέρνηση του Πολμπιά έχει αποχαλινωθεί και παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυβέρνηση οργανώνει ή κατηγορείται για νοθεία στις εκλογές για να παραμένει στην εξουσία και συλλαμβάνει τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Επίσης, οι δύο αγγλόφωνες επαρχίες είναι σε κατάσταση πολέμου. Στη βόρεια της χώρας εξουσιάζει το Μπόκο Χαράμ. Και υπάρχουν βεβαίως και διάφορες ένοπλες ομάδες. Ο στρατός λοιπόν αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις, τις οποίες οπωσδήποτε καταδικάζουμε, αλλά πρέπει να δούμε τις βαθύτερες αιτίες της καταστροφής αυτής, η οποία λέγεται κυβερνητική ακινησία, γέροντοκρατία, κάκο διαχείριση, νοθεία νεποτισμός και φιλετισμός. Αυτές είναι οι αιτίες καταστροφής χώρας και του μαζικού εκπατρισμού των νεαρών Καμερουνέζων. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μια λύση αντί να γίνεται νοθεία στι εκλογέ και να συλλαμβάνονται ειλικρινεί ηγέτε. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε σε μια στιγμή δύσκολη όπου υπάρχουν εγωισμοί στα κράτη-μέλη και προβλέπεται η επιστροφή των εθνικιστών. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω το προσωπικό μου, το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους διερμηνείς και θα συνεχίσω να υπηρετώ τους Ιταλείς. Ευχαριστούμε. Ε, και ε, το ίδιο ευχόμαστε και εμείς τους Ιταλούς ε, ψηφοφόρους όπως εσείς. Ευχαριστώ κύριο Σαφόζερ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόκειται για την τελευταία μου παρέμβαση εδώ στο Κοινοβούλιο και μιλώ για μια χώρα ιδιαίτερα προσφυλή σε μένα που την έχω διανύσει πολλές φορές και αισθάνομαι και λίγο τέχνο της. Το Καμερούν είναι ψηφιδωτό, πολύ εύθραυστο, εθνικό, θρησκευτικό και κοινωνικό. Σίγουρα υπερέβαλε ο Πόλμπια στη συγκεντρωτική του προσέγγιση, υποδαφλίζοντας ε, τα ε, αισθήματα των ε, Αγγλοφόνων ε, της δύση και των αποσχιστών του Βορρά. Αλλά αυτά υποταβλίζονται ακόμα περισσότερο από εξωτερικές δυνάμεις. 37 χρόνια είναι στην εξουσία ο Πολ Μπιά. Παρ' όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, είναι 37 έτη σταθερότητας και είναι πολύ καλή η θέση του Καμερούν σε σχέση με άλλες χώρες. Σίγουρα δεν μπορεί μέχρι να πεθάνει να μονοπολεί την εξουσία ο πρόεδρος, αλλά ε, είναι εχμάλωτος λογικής εξουσίας και διαδοχής. Ξέρει ότι η δημοκρατική μετάβαση και η αποκέντρωση μαζί με ε, την ασφάλεια και την ανάπτυξη ε, είναι αναπόφευκτα. Θα πρέπει να τον βοηθήσουμε, αλλά με τρόπο χρήσιμο και διακριτικό. Ας αποφύγουμε λοιπόν να αναμειχθούμε σε αυτή τη διαδικασία ε, τους ιδεολόγους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ έχουμε πάντα δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάλογα με την Αφρικανική χώρα και ανάλογα με τα δικά μας συμφέροντα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθεί η διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ τώρα και πρώτος είναι ο κύριος Φαρία. Παρακαλώ. Ο κύριος Πόσπεσιλ, όχι ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συζήτηση που έγινε εδώ ε, δείχνει ε, ακριβώς ε, ποιο είναι το πρόβλημα του Καμερούν. Πολύ ωραία το περιγράψαμε. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπρόσωποι μας. Να αυξήσει την πίεση ε, στον σημερινό πρόεδρα που κυβερνάει από το 82 και να βοηθήσει το λαό του Καμερούν. Έτσι ώστε να αφαιθεί ελεύθερος ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και να μπορέσει να κατέλθει υποψήφιος στις εκλογές και όχι να κρατείτε επειδή τόλμησε να γατεύει υποψήφιο απέναντι στον ίν πρόεδρο. Τι είναι αυτή η καταπίεση και ο εκφοβισμός. Δεν μπορούμε ε, να συζητούμε για κράτος δικαίου στο Καμερούν έτσι όπως έχει η κατάσταση. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλή δουλειά για να βοηθήσουμε και κυρία Επίτροπε νομίζω ότι θα ήταν καλό να πείσουμε ε, την ηγεσία του Καμερού να μην φυλακίζει Σόβια τους ε, πολιτικούς αντιπάλους. Ο κύριος Μαριάς παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σημερινή μου ομιλία είναι η τελευταία μου ομιλία σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Ελπίζω και εύχομαι να είμαστε μαζί ξανά και στην επόμενη θητεία, αλλά αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί από τους ίδιους τους Έλληνες πολίτες κατά πόσο θα μου δώσουν την ευκαιρία να επανεκλεγώ στην επόμενη ευρωβουλή. σε κάθε περίπτωση συμπληρώνω 2.532 ομιλίες και παρεμβάσεις εδώ στην ολομέλεια και θα ήθελα με την αφορμή αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους να ευχαριστήσω το προεδρείο και εσάς κύριε πρόεδρε τους διερμηνείς και όλους τους υπαλλήλους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και να πω βεβαίως ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τον ελληνικό λαό γιατί εγώ παίζω εθνική ελλάδος. από εκεί και πέρα σε σχέση με το θέμα μας πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε το καμερούν πρέπει να επικρατήσει δημοκρατία σε αυτή την αφρικανική χώρα για να μπορέσει πραγματικά να προχωρήσει ο ίδιος ο λαός του καμερούν και να επιληθούν τα προβλήματα. ευχαριστώ πολύ κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Καστάλτο, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, στο Καμερούν η κατάσταση έχει φτάσει σε, αφόρητα, σε αφόρητες καταστάσεις. Βλέπουμε αυθαίρετες συλλήψεις του αρχηγού της αντιπολίτευσης για ειρηνική διαμαρτυρία μετά την ε, νιωστή ε, μπεκλογική αναμέτρηση η οποία νοθεύτηκε. Ε, το ίδιο συμβαίνει επίσης και με λοιπούς ανεξάρτητους ε, δημοσιογράφους και Έχουμε επίσης και ματηρή καταστολή των εξεγέρσεων ε, στα βόρειο-ανατολικά και τα νότια-δυτικά. Και βεβαίως ε, βλέπουμε ότι Συχνά οι στόχοι της καταστολής είναι σχολεία και νοσοκομεία ακριβώς επειδή ξεσηκώνονται μαθητές και φοιτητές. Θα πρέπει να οργανώσουμε το συντομότερο δυνατόν έναν πολιτικό διάλογο για να βρεθεί μια ειρηνική και μόνιμη λύση στην κρίση μεταξύ αγγλόφωνων και γαλλόφωνων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια διπλωματική παρέμβαση για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων. Επίσης ε, θα πρέπει να δούμε θα γίνει σε σχέση με την Συμφωνία του Κότων. Σας ευχαριστώ. Στάνισλαβ Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ότι εδώ συζητάμε στις Ολομέλειες για ανθρώπινα δικαιώματα, στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι πολύ σημαντικό που υψώνουμε την ε, φωνή μας και με μία φωνή μιλάμε για αυτά. Αυτό δείχνει ξεκαθαρά ότι είμαστε ενωμένοι για αυτό το ζήτημα και το εκτιμάω ιδιαίτερα αυτό. Τώρα που μιλάμε για το Καμερούν, προφανώς οι θανατώσεις, οι διώξεις, οι βασανισμοί είναι χωρίς να γίνονται προηγουμένως δίκες, δίκες, είναι κάτι απαράδεκτο. Και γίνεται από το στρατό στον οποίο δίνει οδηγίες ο πρόεδρος, ο οποίος παραμένει στην εξουσία τόσα πολλά χρόνια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και παρόλο που ξέρουμε ότι το Καμερούν μάχεται βέβαια κατά του Μπόκο Χαράμ, παρόλα αυτά δεν μπορεί και να κλείνουμε τα μάτια στις άλλες καταχρήσεις που γίνονται. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που ακούμε ότι συμβαίνουν στο Καμερούν είναι φρικτά, ειδικά στον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και για το ότι φυλακίζεται η αντιπολίτευση χωρίς ε, λόγο, ειδικά ο Μωρίς Καντό. Γι' αυτό είναι σαφές ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ε, καταστέλουν τον ίδιο του το λαό. Πολλοί κόσμος έχει διωχθεί από τα σπίτια του, είναι διεσπαρμένοι στο Καμερούν, σχεδόν μισό εκατομμύρια και 30.000 άλλοι έχουν καταφύγει στην Νιγηρία. Οπότε, σωστό και λογικό είναι να ασκήσουμε πίεση στις αρχές της χώρας πρώτα απ' όλα για να απελευθερώσουν τον Μωρίς Καντό και τους συντρόφους του και κατόπιν για να εδραιωθεί η δημοκρατία στη χώρα και ειδικά για να υπάρξουν ε, ελεύθερα και ανεξάρτητα μήμια. Χωρίς αυτά δεν θα σημειωθεί πρόοδος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιχαέλα Σόιντροβα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Αυτό το καπετεπίγον σαφέστατα υπογραμμίζει στην κυβέρνηση του Καμερούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί την κατάσταση και διαφωνεί με την υπερβολική χρήση βία στην καταστολή των ανθρωπινών δικαιωμάτων και της αντιπολίτευσης, της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και διπλωματικά μέσα στη διάθεσή της και οικονομικά μέσα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Είμαι επεπισμένη ότι θα αντιδράσει η κυρία Μογκερίνη γιατί μας ακούει και τα μελήματά μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους συνάδελφοι σε αυτό το σημείο για τη συνεργασία μας επί μία πενταετία. Συζητούμε αυτά τα κατεπήγοντα, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνεχώς ε, ζητούσαμε την απελευθέρωση των κρατουμένων, των διακομμένων ε, λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων ή της εθνικής τους ε, προέλευσης ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η θητεία. Γι' αυτό θα ε, υπερασπιστώ τη δική μου εντολή και θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι. Ο, ο, ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Σόιντροβα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εκλογές. Ο κύριος Σόγκορ. Just a few weeks ago, the Vice Governor... Πριν από λίγες εβδομάδες η κυβέρνηση του Τιβέτ είπε ότι η κατάσταση είναι καλή, πολύ καλή και πολλοί εκτιμούν τη δουλειά που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα εκεί. Οι Θιβετιανοί ποτέ δεν είχαν μια καλύτερη ανάπτυξη στην οικονομία τους και φροντίζουν ο κόσμος να έχει ό,τι χρειάζεται για να μην πυρποληθούν. Και δεν είναι μόνο οι Θεβετιανοί. Εποφελούνται και από την τεχνητή νοημοσύνη, τις τεχνολογίες για να γίνει η ζωή τους πιο εύκολη και πιο απλή. Να έχουν πρόσβαση σε, σε συστήματα εκπαίδευσης διαβίου επίσης. Με τα ίδια μέτρα μπορούμε να πούμε ότι ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα πάει καλά και προωθεί τις αξίες μας. Συγγνώμη, δεν μπόρεσα να μιλήσω όταν είχα ε, χρόνο στην προηγούμενη συζήτηση. Κάτι τεχνικό πρόκυψε και δεν μπόρεσα. Αυτή είναι η τελευταία φορά που μιλάω μετά από 11 χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, χαίρομαι αγαπητέ ε, Τσάμπα, που είχα την ευκαιρία να σας ε, δώσω το λόγο παρόλα αυτά. Η κυρία Μογκερίνη, παρακαλώ, για να κλείσει η συζήτηση για το Καμερούν. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου είδαμε εντάσεις στη χώρα, ειδικά στις λεγόμενες αγγλόφωνες περιοχές. Καταστολή διαδηλώσεων και περιορισμό του πολιτικού χώρου βασικές μορφές αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί, αντιμετωπίζουν στρατοδικία. Πάνω από 100 διαδηλωτές ε, αντιμετωπίζουν ε, μακροχρόνια κράτηση. Οι δικηγόροι τους λένε πως οι νομικές διαδικασίες του Καμερούν δεν γίνονται σεβαστές. Υπάρχει επίσης de facto απαγόρευση των πόριών και διαδηλώσεων της αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο ξεκάθαρα παραβιάζει το Σύνταγμα του Καμερούν. Παρακολουθούμε την κατάσταση εκ του ε, για λογαριασμό των 28 κρατών μελών. Ζητήσαμε την απελευθέρωση κρατουμένων για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία και να σταματήσει άμεσα η βία, η παραβιάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ρητορική του μίσους. Και επιμένω και σήμερα σε αυτό. Και σας ευχαριστώ που βάλατε αυτήν τη σημαντική συζήτηση στην ημερήσια διάταξη την τελευταία ημέρα της ε, θητείας σας για να τονίσετε αυτό το μήνυμα όσον αφορά την κατάσταση στις αγγλόφωνες περιοχές ε, βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά Έχουμε πει πως ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μια μόνιμη λύση με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Δυστυχώς, οι δολοφονίες ε, και οι ακρότητες ε, εξακολουθούν και από ό,τι φαίνεται περιλαμβάνουν και τις δυνάμεις ασφαλείας ε, και τις αποσχιστικές ομάδες. Η κατάσταση είναι ανησυχητική. Ε, περίπου μισό εκατομμύριο είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι και 32.000 ε, πρόσφυγες έχουν καταγραφεί στην Ιγυρία. Έχουμε ζητήσει αυτοσυγκράτηση και διάλογο από τις αρχές του Καμερούν. Ειδικά παρακολουθούμε εκ του περίπτωση των 47 αγγλόφωνων ηγετών που έχουν φυλακιστεί και ζητάμε δίκαιη δίκη. Αυτά προστίθενται στις συνεχείς επιθέσεις που αναφέρατε του Μπόκο Χαράμ αλλά και στο Τσάντ, ε, τον Νίγηρα και την Ιγυρία. Ξέρουμε πως βεβαίως το Μπόκο Χαράμ δεν είναι ανίκητο, έχει υποφέρει, έχει υποστεί μεγάλες ήττες αλλά βλέπουμε απώλειες αμάχων ε, και ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας. Δεδομένου του ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Νιγηρίας έφτασαν στον βορρά του Καμερούν, θα ήθελα και εγώ να συνταχθώ με την έκκληση της υπατσαρμοστίας του ΟΗΕ για να εφαρμοστεί η αρχή της μη επαναπροώθησης. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να αναλαμβάνουμε και εμείς οι ανθρωπιστικές μας ευθύνες θεωρούμε και τους εσωτερικά εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες ε, που έρχονται από την Ιγυρία και την Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία στην ίδια μοίρα. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο ανθρώπους και νομίζω πως έχουμε ένα ανθρωπιστικό καθήκον και αυτό είναι κάτι βέβαια στο οποίο δεν μπορούμε να ξεχνάμε όταν θα αξιολογούμε τη μελλοντική μας στήριξη στον λαό του Καμερούν. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να ζητάμε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και να διαλευκανθούν πλήρως οι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπατική Πρόσωπε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που παραμένετε μαζί μας και για το επόμενο θέμα έχουμε 8 προτάσεις ψηφίσματος για να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Πάντως από το ΙΣΙΑΡ, την ΚΟΕ, το ΕΛΚ, τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους. Ολοκληρώνω τη συζήτηση εδώ για αυτό το θέμα και θα ψηφίσουμε αργότερα. Ολοκληρώνουμε τι συζητήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Μπρουνέι. Έχουμε τους συντάκτες. Θα δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στην κυρία Μπάρμπαρα Λοφμπίλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη το 2014 το Μπρουνέι ε, εισήγαγε τη Σαρία και στις 3 Απριλίου ε, τι ισχύ με τη τελευταία φάση. Ε, ομόφυλα ζευγάρια, εξωσυζυγικές σχέσεις, εκτρώσεις τιμωρούνται με λιθοβολισμό για την κλοπή κροτηριασμό χεριού, για τη δυσφήμιση του προφήτη Μοχάμετ θανατική ποινή. Τα παιδιά μπορούν να θεωρούνται ε, ότι μπορούν να υποστούν ε, τις συνέπειες του νόμου από την ηλικία των 7 ετών. Ο Σουλτάνος ε, θα πρέπει να σταματήσει αυτή την κατάσταση και να άρει τη Σαρία. Αυτό είναι κατάφορη αντίφαση και απέναντι στο διεθνή νόμο. Πέρα από το φύλλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την προέλευση και τη θρησκεία, οι άνθρωποι είναι ίσοι. Από το 1957 ε, υπάρχει μορατόριο de facto δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή ε, στο Μπρουνέι και θα πρέπει αυτό να οδηγήσει τελικά στην κατάργηση της θανατικής ποινής. Θα πρέπει να αλλάξει τον ποινικό κώδικα των Μπρουνέι ε, και να το ευθυγραμμίσει ε, με τα διεθνή ισχύοντα. Τότε και μόνο τότε θα πρέπει να ξανασκεφτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία. Επίση, θα πρέπει να φροντίσουμε η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπρουνέι, ιδιαίτερα η κατάσταση και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, να εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη του επόμενου διαλόγου Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΣΕΑΝ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Τσάρλ Τάνοκ. Πρόεδρε, αναθεώρηθηκε ο ποινικό κώδικα στο Μπρουνέι της 3 Τετάρτου. Ε, είναι πολύ θλιβερό αυτό. Ε, διευρύνονται τα εγκλήματα ε, που τιμωρούνται με τη θανατική ποινή, όπως είναι οι εκτρώσεις, οι εξωσυγικές σχέσεις, οι σχέσεις τα κτλ ευθυγραμμίζεται με τη Σαρία σύμφωνα με την απόφαση του Σουλτάνου. Επίσης μπορεί κανείς να ακροτηριάζεται μετά από κλοπή. Ε, αυτή ε, μας ανησυχεί πολύ η εξέλιξη, ιδιαίτερα τις σκεφτικές κοινότητες και τους ΛΟΑΤΚΙ που θα κινδυνεύσουν ιδιαίτερα στο Μπρουνέι. Ε, δεν χωράει ένα τέτοιο δρακόντιο ποινικό σύστημα στο σημερινό κόσμο. Έχει δεσμευτεί το Προυνέι διεθνώ. Ω βουλευτή από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανησυχώ πάρα πολύ γιατί είναι και μέλος της κοινοπολιτείας το Μπρουνέι. Ε, είναι η τελευταία μου ομιλία ως Ευρωβουλευτής αυτή η θλιβερή. Μετά από 20 χρόνια που έχω υπηρετήσει εδώ, είναι μεγάλη τιμή και χαρά αυτή η ευκαιρία που είχα να ε, υπηρετώ εδώ και σας λέω ευχαριστώ και μπορεί και στο επαριδίν. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Τάνο, αγαπητέ Τσάρλς. Η Μελίν Μπιόργ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η νομοθεσία στο Μπρουνέι καταδικάζει τους ΛΟΑΔΜΗ και άλλους πολίτες σε βασανισμούς, σε θανατική ποινή και έτσι εγώ με τους συνσυντάκτες του ψηφίσματος καταδικάζουμε αυτή την κατάσταση και την καταγγέλουμε Χρησιμοποιείται η θρησκεία και ο χριστιανισμός πολλές φορές για να διαδοθεί το μίσος, για να καταπιεστούν οι γυναίκες και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΔΜΗ. Για να ενοχλούμε τον κόσμο για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν το σώμα τους. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμβαίνει στον Μπρουνέ ούτε και εδώ. Τι λέει ότι αυτό το καταγγέλουμε, ότι πρέπει να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση, ότι πρέπει να δράσουμε για να διορθωθεί η κατάσταση σε αυτό το αυταρχικό κράτος, αλλά η πολιτική μίσους δεν είναι μόνο εκεί, υπάρχει παντού, το βλέπουμε και στην Κολομβία, όπου και εκεί Έχουμε ακόμα και πολιτικούς από τη Σουηδία που συμβάλλουν στην καταπίεση. Ναι, να υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε άλλες χώρες, αλλά να σκουπίσουμε και μπροστά στην πόρτα μας λιγάκι. Το μίσος κατά της κοινότητας Λουαθμή δεν έχει θέση ούτε εδώ, ούτε πουθενά αλλού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κοράου τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας ε, κυρία Μογκερίνη. Πρώτα απ' όλα ε, θέλω να πω πως ε, πρόκειται για την τελευταία μου παρέμβαση αυτή τη θητεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να είναι στο επίκεντρο των εμπορικών διαπραγματεύσεων μας. Κλείνουμε με το Μπρουνέι που θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο εξόφθαλμες περιπτώσεις. Ένα σουλτανάτο το οποίο ο σουλτάνος μπορεί να έχει πέντε συζύγους ε, και να έχει και διάφορες έσκορτ ε, αλλά στην ίδια χώρα ταυτόχρονα για τους υπόλοιπους επικρατεί θανατική ποινή για τη μοιχεία. Ε, λοιπόν, χαιρόμαστε που διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις με αυτήν την χώρα και θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζουμε να μην επαναληφθούν διαπραγματεύσεις από αυτό. Και μπορούμε βεβαίως να επιτύχουμε και καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι πετύχαμε σε αυτήν την θητεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σοράγια το έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε. Ζούμε μία κρίση Όλος ο κόσμος είναι σε κρίση. Έχουμε την κλιματική κρίση. Έχουμε υπερσυντηρητικές σκοτεινέ δυνάμεις που μας πλησιάζουν στα κοινοβούλια μας. Και έχουμε και μια κρίση δικαιωμάτων των γητεκών, δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ και για τα απλά ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία βρίσκονται υπό επίθεση και στην Ευρώπη και στον κόσμο ο εθνικισμός είναι κρίση για τη δημοκρατία μας. Οπότε θα ήθελα να σας πω σε όλους εσάς τα θεωρία. Είναι η δική σας ευθύνη να διαφυλάξετε τις δημοκρατικές μας αξίες στις 26 Μαΐου. Και σε όλους τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφυλάξετε τις αξίες μας. Όταν μιλάμε για τον Μπρουνέη και την Σαρία που ισχύει ο ποινικό κώδικας είναι κάτι το εξευτελιστικό και απάνθρωπο στοχεύει ανθρώπους που είναι ήδη ευπαθείς, ε, γυναικόπαιδα, ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Και τους στερεί τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, παιδιά ακόμα και 7 ετών μπορούν να μαστιγωθούν. Συνενετικές ερωτικές πράξεις τιμωρούνται με λιθοβολισμό. Στις πολιτισμένες κοινωνίες τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά. Δεν είναι έγκλημα να είναι κανείς ομοφιλόφιλος, λεσβία ή να κάνει έκτρωση. Εγώ απαιτώ άμεσο τερματισμό αυτού του νέου ποινικού κώδικα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στεχόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είπατε εκπρόσωποι μαγερινη και εγώ θέλω να συμφωνήσω με όλους εκείνους που ευχαρίστησαν για τη συνεργασία εδώ τα 5-7 χρόνια για τα κατεπήγοντα. Συχνά λέμε τι θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή κάποιος Ευρωβουλευτής. Όμως χάρη στα κατεπήγοντά μας, χάρη στα ψηφίσματά μας αυτά για τα κατεπήγοντα, καταφέραμε να ελευθερωθούν κάποιοι φυλακισμένοι ή να βοηθήσουμε στην αλλαγή καθεστώτος σε μια χώρα και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, καλά συγκεκριμένα παραδείγματα. Πρόσφατα επικρίναμε την κατάσταση στις Μαλβίδες και το Σεπτέμβριο του 2018 είδαμε να αλλάζουν τα πράγματα και να κερδίζει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον οποίο εμείς στηρίξαμε. Νομίζω λοιπόν ότι η δύναμη του δικού μας έργου μπορεί να αλλάξει την κατάσταση και στον Μπρουνέι. Εγώ έχω επικρίνει όλες τις χώρες που προσπαθούν να επιβάλλουν τη Σαρία για χρόνια. Και ακριβώς γιατί ο νόμος της Σαρίας δεν έχει να κάνει τίποτα με την σύγχρονη δημοκρατία. Δεν έχει καμιά σχέση με τον πλουραλισμό. Αφορά πολλές ομάδες, θρησκευτικέ, μειονότητες, που επειδή κάποιος έχει διαφορετική άποψη από τη δικιά τους, τους επιβάλλει κυρώσεις, τους τιμωρεί, δεν τους σέβεται. Επειδή θα θέλανε κάτι διαφορετικό, θα θέλανε να μπορούν να ακούγονται οι δικές τους οι απόψεις. Λοιπόν, όλοι εμείς πρέπει να αγωνιστούμε για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία για όλους μας, όλους εμάς τους Ευρωπαίους. Ευχαριστούμε, Μερικά Σχάκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε οι εκπρόσωποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν από 10 χρόνια, η πρώτη μου παρέμβαση στην Ολομέλεια αυτή είχε να κάνει με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Οπότε ταιριάζει απόλυτα. Και η τελευταία μου παρέμβαση να είναι πάλι για ανθρώπινα δικαιώματα. Τι παραπάνω μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί θα το κάνουμε εμεί, ποιο θα το κάνει. Η Σαρία στο Μπρουνέι, έτσι όπως εφαρμόζεται, είναι τόσο ακραίο που πλήττει τα παραγωγικά γη, ε, δικαιώματα, την υγεία και βέβαια την κοινότητα ΛΟΑΔΜΗ. Το 2019, μα είναι εξωφρενικό, είναι βάρβαρο. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε τύπου Μακνίσκι κυρώσεις και ήδη βλέπουμε ότι η πίεσή μας φέρνει κάποια αποτελέσματα. Είπατε εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κάνω έκκληση σε εσά να συνεχίσετε να αγωνίζετε για μια ισχυρή Ευρώπη η οποία βάζει πρώτα απ' όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τις παρεμβάσεις των 7 συντακτών ε, ψηφισμάτων και τώρα εκ μέρους των σοσιαλιστών το λόγο έχει η κυρία Τζίλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία εκπρόσωπο. κανείς δεν πρέπει να διώκεται ε, για το ποιο είναι και για το ποιους αγαπάει. Όμως ακούμε ότι στον Μπρουνέι αυτά συμβαίνουν. Η Σαρία, η οποία περιλαμβάνει ακροτηριασμούς, λιθοβολισμούς και διάφορα άλλα τέτοια. Οι νόμοι αυτοί πέρασαν γιατί το ζητούσε ο λαός. Αλλά αυτό γίνεται γιατί η οικονομία καταραίει, το καθεστώς δεν είναι δημοφιλές και τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για να αποσπάσουν την προσοχή του λαού. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να καταδικάσει τις βάρβαρες αυτές ε, πρακτικές ε, για να υπάρξει και στοχευμένη άρνηση βίζας ε, για το καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν να μην εφαρμοστούν αυτά τα δρακόντια μέτρα. Αυτό θα γίνει μόνο με διεθνή καταδίκη και με διάλογο. Είπατε εκπρόσωπε, πρέπει να σταματήσουμε να φρύτουμε μόνο. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Και τέλος, να πω κάποιου συναδέλφου. σω πρόκειται για την τελευταία μου ομιλία και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλου για τη συνεργασία. Ευχαριστώ από την ομάδα των Ευρωπαίων Συνδικών και Μεταρρυθμιστών, ο κ. Δεμέσμακε. Σήμερα και σωστά διατρανώνουμε την έντονη δυσφορία μας ε, σχετικά με την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα στο ε, Μπρουνέι ακροτηριασμός, ε, δημόσια λοθοβολισμοί, ακροτηριασμοί, ε, αυτά είναι μεσαιωνικά πράγματα, αλλά σήμερα τα χρησιμοποιούν για, ως αντίπεινα για ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Ε, τα κράτη είναι υπεύθυνα για τους κανόνες τους, αλλά και οι κανόνες αυτοί ε, την στην καθολικότητα των παγκοσμίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα πρέπει να σεβόμαστε το εθνικό πλαίσιο, λέει, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των γυναικών παιδιών και τη κοινότητα ε, ΛΟΑΤΚΙ, που παραβιάζονται συστηματικά. Συνάδελφοι, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στην τελευταία συζήτηση τη παρούση θητεία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι ποτέ δεν είναι κατακτημένα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόνο η πολιτική πίεση μπορεί να αλλάξει κάτι ε, αν παραβιάζονται κατάφορα όπω το Μπρουνέι. Σήμερα το ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, να πιέσουν για να ε, καταργηθούν αυτά τα δρακόντια μέτρα. Μπορεί να είναι πλούσια, πάμπλουτη χώρα, αλλά πραγματικά ε, η ηθική ένδυα του ηγέτη τη είναι για μένα διαμφισβήτητη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καστάλτο, παρακαλώ. Συνάδελφοι, ο Ασενάλ Μπολκεάλ, ο Σουλτάνος του Μπρουνέη, πιο πλούσιος άνθρωπος ε, του κόσμου για κάποια χρόνια, έγινε διάσημος ε, για το χαρέμι του, για την επιδεικτική σπατάλη του και ταυτόχρονα ο ίδιος άνθρωπος έπιχε επιβάλει την Σαρία. Δεν πρόκειται για παρεξήγηση. Απαγορεύεται λοιπόν μεταξύ άλλων οι ομοφιλοφιλικές σχέσεις, ή ε, εκτρώσεις, και τιμωρούνται με θανατική ποινή. Άλλα πράγματα τιμωρούνται με ακροτηριασμό χεριών και ποδιών και ισχύουν αυτές οι ποινές και για ανηλίκους. Οπωσδήποτε ο κώδικας αυτός θα έπρεπε να εφαρμοστεί ομοιόμορφα. Αν γινόταν αυτό, θα κινδύνευε βεβαίω και η ίδια η βασιλική οικογένεια και ο ίδιο ο Σουλτάνο. Τέλο, αγαπητοί συνάλφοι, θα ήθελα στην ε, τελευταία μου παρέμβαση, να πω αυτό το οποίο είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, να σας ευχαριστήσω όλους για τη δουλειά που κάναμε και για την δύναμη με την οποία υπερασπιστήκαμε τις αξίες μας αυτές, τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν κάνει την Ευρώπη μεγάλη και ελπίζω να είμαι εδώ πέρα και στην επόμενη θητεία για να συνεχίσουμε μαζί να την ε, δράση μας ε, έτσι ώστε η εξωτερική μας δράση, οι εξωτερικές μας σχέσεις να χαρακτηρίζονται πάντα από τους αξίες μας, τα δικαιώματα και τα δικαιώματα ειδικά των πιο ευπαθών. Σας ευχαριστώ από βάθος καρδίας και καλή τύχη σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, αλλά παρακαλώ να σεβόμαστε και το χρόνο μας. Διότι ε, σήμερα δεν χωράει καθυστέρηση. Κυρία, ο κύριος Κολομπιέ. Κύριε Πρόεδρε, ε, στο Μπρουνέι τι κάνουν, έχουν σαρία. Απιστία, θανατική ποινή. Ομοφιλοφιλία, θανατική ποινή των ανδρών. Για τις γυναίκες, 40 ραβδισμοί και φυλάκιση. Ε, περίεργη ε, διάκριση αυτή, αν είσαι άνδρας ή γυναίκες. Πραγματικά τώρα τι, να είναι χειρότερο, το γελίο ή το επαχθές. Ε, η ε, δυσφήμιση του προφήτη θανατική ποινή. Εδώ έχουμε την, ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε μια υπόθεση κατά της Αυστρίας ε, έχει αρνηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα επίκριση στο Ισλάμ. Τέτοια ανεκτικότητα από το δικαστήριο απέναντι στο ε, ριζοσπαστικό Ισλάμ, όσο ισχύει αυτό, εμεί δεν μπορούμε να στρεφόμαστε απέναντι σε τέτοια δεχτή καθεστώτα όπω είναι το Προυνέ. Άλλη μια φορά κυβερνάνε εδώ αδυναμία και υποκρισία. Αφήστε την ελευθερία της σκέψης πρώτα να ε, ανθίσει στην Ευρώπη και να μην κάνουμε μαθήματα σε άλλους. Τελευταία είναι αυτή η ομιλία. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για το έργο που γίνεται εδώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία στους αντικαταστάτες μου για μια Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Ελευθέρων Λαών και των Κυρίαρχων Εθνών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βαλενθιάνο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι πολύ καλά εξήγησαν τι σημαίνει ε, αυτή η σκληρή αντιμετώπιση του Μπρουνέη κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Είναι ένα παράδειγμα το Μπρουνέη, ένα ανάμεσα σε πολλά, σε ολόκληρο τον κόσμο που οι ελευθερίες και τα δικαιώματα οπισθοχωρούν αντί να βελτιώνονται. Πρόκειται για μια οικουμενική αξία τα ανθρώπινα δικαιώματα και για μένα είναι η τελευταία μου παρέμβαση στην Ολομέλη εδώ και θα ήθελα να αφήσω ένα μήνυμα στο όνομα όλων εκείνων που βρίσκονται σε διάφορα δύσκολα σημεία του κόσμου και αγωνίζονται για την ελευθερία, για τη ζωή και ελπίζω το σώμα αυτό να μην τους ξεχάσει ποτέ. Μπορεί να βρίσκονται μακριά, αλλά ακριβώς υποστηρίζουν τις αξίες που και εμείς υποστηρίζουμε εδώ. Λίγοι συμμετέχουμε στις συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζω όλο και περισσότεροι να έρχονται εδώ και να μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όταν ε, εδώ σε αυτό το πολυτελέσιμο κύκλιο ε, σηκωνόμαστε, μην να μιλήσουμε, μην ξεχνάμε τι φυλακέ, μην ξεχνάμε τι γυναίκε που αγωνίζονται για τα δικαιώματά του, μην ξεχνάμε του ομοφυλόφιλου που σφαγιάζονται σε διάφορε χώρε. μην ξεχνάμε σε ποιε αξίε πάνω βασίστηκε η οικοδόμηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και σα ευχαριστώ όλου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βαλενθιάνο. Αγαπητή Ελένα, για αυτήν την τελευταία σου παρέμβαση σε αυτήν τη θητεία. Τώρα περνάμε στις ε, ελεύθερες παρεμβάσεις. Κύριε Φάρια, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, είναι η τελευταία μου παρέμβαση εδώ στο σώμα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο ασχοληθήκατε με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρία Μογκερίνη, μετά από τις νέες ρήτρε αυτές στον ποινικό κώδικα του Μπρουνέη που καταδικάζει διεθνή κοινότητα, ο Σουλτάνος Βολκιά προσπαθεί να τον εφαρμόσει από το Δεκέμβριο που μας πέρασε χωρίς αντιδράσεις. Είναι κάτι που επαναφέρει ε, μέτρα τα οποία χρησιμοποιούνταν το μεσαίωνα, είτε πρόκειται για τον λιθοβολισμό, είτε πρόκειται για τον ακροτηριασμό άκρων μετά από κλοπή. Ακούστηκαν φωνές ολόκληρο τον κόσμο που καταδικάζουν αυτές τις σκληρές και απάνθρωπες πρακτικές ενώ βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Ο Σουλτάνος έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα, οπότε θα έπρεπε να παγώσουμε τα περιουσιακά του στοιχεία και να το βάλουμε στη μαύρη λίστα. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και πρέπει να ανακληθεί και να συμμορφωθεί προς τα διεθνή πρότυπα. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τζούλι Βόρτ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Όταν εξελέγινε το 2014 αποφάσισα να είμαι η φωνή αυτών που δεν είχαν φωνή. Και να είμαι πάλι να χρησιμοποιώ αυτό το εκπληκτικό βήμα για να υπερασπίσω τα ανθρώπινα δικαιώματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σοκαρό, σοκαρίστηκα όταν άκουσα ότι ο Σουλτάνο του Μπρουνέ αποφάσισε να επιβάλλει την θανατική ποινή για μοιχεία και ομοφιλοφιλία. Η θανατική ποινή είναι πάντα απαράδεκτη και πρέπει βεβαίω να είμαστε ενάντια. Αλλά η κατάσταση αυτή είναι ε, ακόμη χειρότερη γιατί είναι κατά των γυναικών. Και δεν επιτρέπεται στα άτομα να αγαπούν αυτούς που θέλουν. Όταν μιλάμε για σεξισμό και ομοφοβία εδώ στην Ευρώπη, πρέπει να θυμόμαστε ότι οποιαδήποτε διάκριση, όσο μικρή και αν φαίνεται, δημιουργεί ένα παγκόσμιο κλίσμα, κλίμα μίσους ε, που οδηγεί σε θανάτους ανθρώπων, ε, είτε στα χέρια του κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού. Πρέπει να συνεχίσουμε να καταπολεμάμε τις διακρίσεις αυτές. Και ζητώ από την ύπατη εκπρόσωπο να χρησιμοποιήσει όλες τις διπλωματικές διάβλους για να πιέσει τις αρχές του Μπρουνέη να ανακαλέσουν αυτούς τους μεσεωνικούς ε, νόμους και να τερματιστεί η θανατική ποινή στη χώρα αυτή και αλλού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Μιράντα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα κομμάτι της δουλειά μου εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορούσε την υπερασπίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων που δεν έχουν φωνή στην Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Μογκερίνη επίσης για τον ε, συμβιβασμό της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να πω πως πρέπει να σταματήσουμε την θανατική ποινή και τις διακρίσεις ε, παντού και στην Ευρώπη. Η δύσκολη κατάσταση του Μπρουνέη όσον αφορά την ομοφοβία ε, σημαίνει ότι πρέπει να υπερασπίσουμε την ε, αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων. Ανήκω στην ομάδα ΛΟΑΤΚΙ του Ευρωπαϊκού με τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είμαι υπερήφανη γι' αυτό, γιατί η μοίρα αυτών των ανθρώπων είναι και δική μας ευθύνη. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να πολεμήσουμε για να υπερασπίσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ε, πρόκειται για την τελευταία μου παρέμβαση αυτήν την θητεία, αλλά θα επανέλθω. Σα ευχαριστώ. Ο ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά τα ίδια ακούμε εδώ. Ε, ε, πεντε 6 άνθρωποι σε ένα-δυο ημικύκλιο υπαγορεύουν στον κόσμο ολόκληρο τι πρέπει να κάνει. Ερωτώ, όλα αυτά τα ψηφίσματα τι επέδωσαν, μια τρύπα στο νερό. Πιστεύετε ότι τα ψηφίσματα αυτά τα διαβάζει κανένας, αυτά που βγάζουμε. Τι θα κάνετε. Ε, αν σας στείλει μαντάτο ο Σουλτάνος του Μπρουνέη, ότι δεν θα πρέπει στην Ευρώπη να σκοτώνετε τις αγέννητες ζωές. Δεν θα τα πάρετε σοβαρά. Ε, ούτε τα δικά σας θα πάρει σοβαρά τις προειδοποιήσεις ο Σουλτάνος του Μπρουνέη. Εδώ συζητάμε για την Κίνα, το Καμερούν, τη Λιβύη, τη Μοζαμβίκη, τον Μπρουνέη και πάει λέγοντας. Και κάνουμε μαθήματα σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Αν δημιουργήσουμε, αν φτιάξουμε μαύρη λίστα, τότε θα μας απομείνουν μερικά κράτη-μέλη που θα είναι εκτός της λίστας. Θα πρέπει να τα σταματήσουμε αυτά, να δίνουμε μαθήματα στον κόσμο ολόκληρο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ε, θα ήθελα να πω ότι ο Σουλτάνος του Μπρουναή εχθές έστειλε επιστολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπάθησε να εξηγήσει σε τι αποσκοπεί με την ομοθεσία αυτή. Παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα συζητούμε την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπρουνέι και τη Σαρία. Βασανισμοί, ε, ομές και ξεφτελιστικές ε, τιμωρίες. Το Μπρουνέι γνωρίζει ότι η Σύμβαση των, Ανθρωπίνων, των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστήριων τα απαγορεύει όλα αυτά. Επανεισαγωγή της αρνητικής ποινής, η ομοφιλοφιλία ε, θα τιμωρείται με θανατική ποινή δια ε, λιθοβολισμού. Αυτά είναι αγριότητες. Το 2015 η Ιρλανδία ήταν η πρώτη χώρα που μετά από δημοψήφισμα νομιμοποίησε το γάμο των ομοφιλοφίλων. Ο κόσμος πάει μπροστά, δεν γυρνάει πίσω. Παντού θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, απευθύνω επίγουσα έκκληση στις αρχές της χώρας να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα, με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών και επιμένω να αποποινικοποιήσει την ομοφιλοφιλία. Ευχαριστώ πολύ και όλες οι χώρες θέλουν το ίδιο μήνυμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ. Η αλλαγή στον ποινικό κώδικα του Μπρουνάη είναι μια ακραία κατάσταση. Πρόκειται για βασανισμό, για σκληρή αντιμετώπιση του κόσμου. Όλα αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λιθοβολισμός, ακροτηριασμοί, ε, για κλοπές ή για σχέσεις ε, μεταξύ ατόμων ιδίου φύλου, ακόμα και συνενετικά. Όλα αυτά γίνονται επειδή τα θέλει ο Σουλτάνος του Μπρουνέη. Δεν ξέρω τι λέει στην επιστολή του ο Σουλτάνος. Νομίζω ότι η κατάσταση είναι υποκριτική αν μας στέλνει επιστολές ε, μετά τα όρια τα οποία διαβάζουμε ότι κάνει στη χώρα του. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εμείς στις συζητήσεις ΑΣΕΑΝ να θέσουμε αυτό το ζήτημα. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η κορονίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι καλό που τα συζητάμε, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος άλλος θα το κάνει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ε, πώς πίσιλ τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να αντιδράσω στον Πολωνό συνάδελφο που αμφισβήτησε την αξία που έχουν αυτές οι συζητήσεις. Εγώ είμαι από την ε, τέως Τσεχοσλοβακία, κομμουνιστική χώρα και εκεί πολλοί αντιφρονούντες που πολεμούσαν, αγωνίζονταν κατά του κομμουνισμού ε, μου έχουν πει ότι πάντα τους ε, άρεσε όταν κάποιος από τις δυτικές χώρες υποστήριζε τον αγώνα τους. Οπότε μην νομίζετε ότι δεν έχει σημασία αυτή η συζήτηση. Έχει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά. Και όταν εμείς υποστηρίζουμε εδώ ανθρώπου οι οποίοι διώκονται σε τρίτε χώρες, έχει νόημα. Έχει σημασία. Οι αντιφρονούντε οι Τσέχοι εκτίμησαν πάρα πολύ το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι δυτικοί τους στήριξαν. Και ακόμα και σήμερα το θυμούνται τη συνάντηση που είχαν με τον τότε πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η συζήτηση και ολοκληρώθηκε και αυτός ο γύρος παρεμβάσεων. Η κυρία Μογκερίνη τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. 3 Απριλίου το Μπρουνέι και ο Σουλτάνος το αποφάσισε για την εφαρμογή του νέου κώδικα. Όπως είπατε, προβλέπει τιμωρίες, ακροτηριασμούς, λιθοβολισμό, πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία θέση στον κόσμο σήμερα. Και επίσης επιτρέπεται και θανατική ποινή. Και ξέρετε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι εντελώς κατά της θανατικής ποινής οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιου είδους τιμωρία. Κανένα έγκλημα δεν δικαιολογεί βασανισμούς, ε, τέτοια βασανιστήρια. Και κανένας δεν θα πρέπει να τιμωρείται επειδή αγαπάει κάποιον άλλον. Ποτέ δεν πρέπει να ερμηνεύεται μια τέτοια αγάπη και σχέση ε, σαν έγκλημα. Πρόκειται λοιπόν για παραβίαση πολλών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το Μπρουνέι διεθνώς. Οι πράξεις αυτές απαγορεύονται από τη Σύμβαση κατά των βασανισμών και κατά ε, απάνθρωπης συμπεριφοράς που έχει υπογράψει η χώρα το 2015. Επίσης, υπάρχει και δήλωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2012 που επίσης παραβιάζεται εφόσον ε, έχει συμφωνήσει με τη σύμβαση αυτή, με τη σύμβαση για την προστασία των παιδιών ή για την καταπολέμηση των παραβιάσεων σε βάρος των γυναικών. Πολλοί από τους διεθνείς εταίρους μας, ο ύπατος αρμοστής ε, Μισελ Μπασλέ για παράδειγμα του ΟΙΕ για τα δικαιώματα των ε, παιδιών έχει καταδικάσει επίσης αυτή την κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να συμμορφωθεί το Μπρουνέι με όλες τις υποχρεώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει συνυπογράψει. Η ευκαιρία της συζήτηση αυτής είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα. Επίσης το μορατόριο όσον αφορά τη θανατική ποινή. Παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση εδώ και χρόνια. Δεν αρχίσαμε να αντιδράμε μόνο πριν από λίγες εβδομάδες. Όταν εγκρίθηκε ο ποινικό αυτός ο κώδικας το 2013, διακόψαμε τις συνομιλίες με τον Μπρουνέη. Και έκτοτε θέτουμε το ζήτημα σε κάθε συνάντηση που έχουμε με τις αρχές της χώρας και στις αιτήσεις εκθέσεις που κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στη χώρα. Είναι βασικό τώρα να φροντίσουμε να μην εκτελούνται τέτοιες τιμωρίες. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε διμερώς τον Μπρουνέη και απευθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μέσω των χωρών μελών. Και η Μαντ Κίλμπερτ, που είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα συνεχίσει να το κάνει αυτό. Επίσης, στο Συμβούλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, όπου γίνεται η αναθεώρηση της έκθεσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα θέσουμε και το θέμα και με τους εταίρους μας από τις χώρες ΑΣΕΑΝ, γιατί πρόκειται για παραβιάσεις στα πλαίσια συμφωνιών που έχει συνυπογράψει το Μπρουνέι. Και θα φροντίσω και εγώ προσωπικά να γίνει αυτό στην επόμενη συνάντηση η ετήσια που έχουμε με τις χώρες ΑΣΕΑΝ τον Αύγουστο που μας έρχεται. Η απαγόρευση τέτοιων τιμωριών δεν έχει να κάνει μόνο με τις ευρωπαϊκές αξίες. Πολλοί το είπατε ότι πρόκειται για οικουμενικές αξίες ε, τις ε, οποίες, ε, στις οποίες πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι, όπου και αν βρίσκονται. Καμία αρχή, καμία χώρα δεν μπορεί να τις παραβιάζει, όπου και αν βρίσκεται. Καμία χώρα δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτές. Πρόκειται για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Και εγώ θα συνεχίσω εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δουλεύω για αυτή την αξιοπρέπεια, προκειμένου αυτή να γίνεται σεβαστή παντού και πρώτα απ' όλα στην Ευρώπη. Είναι η τελευταία συζήτηση εδώ στο σώμα για την θητεία σας αυτή. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη δουλειά που έχετε κάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει βοηθήσει απίστευτα το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα να τον κόσμο και συμφωνώ με αυτούς που υπογράμμισαν ότι στην επόμενη θητεία μακάρι να είναι ακόμα περισσότεροι ευρωβουλευτές οι οποίοι θα ασχοληθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παντού ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε. Νομίζω τα χειροκροτήματα που σας επιφύλαξαν οι συνάδελφοι είναι απόδειξη της αγαστής συνεργασίας την οποία εκτιμούμε πάρα πολύ. Έχω λάβει 7 ψηφίσματα, σχέδια ψηφισμάτων από τις εξής πολιτικές ομάδες. Πράσινη, ΣΥΑΡΓΚΟΕ, EFTD, ε, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Φιλελεύθεροι. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση αυτή. Η ψηφοφορία θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Επευκαιρία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους σας για όλο το διάστημα της συνεργασίας μας. Σας ευχαριστώ που με εκλέξατε αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εύχομαι σε όλους εκείνους που κατέρχονται και πάλι υποψήφοι καλή επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω και τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας και τους διερμηνείς και καλό σας Πάσχα! Να είστε καλά. Λήξη της συζήτησης. Ακολουθούν οι ψηφοφορίες στις 12. president. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Είμαστε συντετριμένοι από το τρομακτικό δυστύχημα με το τουριστικό λεωφορείο στη Μαδέρα όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 29 άνθρωποι και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν. Τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων αυτής της τραγωδίας και θα ήθελα εξ ονόματος του Κοινοβουλίου να ευχαριστήσω τη ε, συνεργεία διάσωσης και παρακαλώ να γερθείτε για να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Φαρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα ακριβώς στην αρχή να πάρω το λόγο πριν τις ψηφοφορίες, γιατί ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε αυτή τη τραγωδία για την οποία μόλις μας μίλησε ο Πρόεδρος. 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ήταν ένα τουριστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε στον κρεμό ε, με Γερμανούς τουρίστες στη Μαδέρα. σε μια πάρα πολύ στενή στροφή και είναι από τα χειρότερα τροχαία δυστυχήματα στη Μαδέρα όλων των εποχών. Με νεκρούς, τραυματίες πολλούς και Πραγματικά θα πρέπει να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων. Και και ενός λεπτού σιγή. Αυτό ήθελα να ζητήσω κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαρία. Ερχόμαστε αμέσω στον κανονισμό, κύριε Καβαδά, μια στιγμή. Οι αρμόδιες γαλλικές αρχές, ε, στα πλαίσια μιας δικαστικής προανάκρισης, ζήτησαν τη ριάση της ασυλίας κυρίας Μαρή Κριστίν Αγνοτού. Σύμφωνα με τον κανονισμό, διαβιβάζεται αρμοδίως στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων το αίτημα αυτό. Μετά την ε, παρέτηση της κυρίας Λίντα Μακάβαν, το Κοινοβούλιο διαπιστώνει τη χειρία της έστης από τις 19 Απριλίου 2019 και ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, δίνω το λόγο στην κυρία Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπα την εκπρόσωπο, την κυρία Μογκερίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ε, ήθιστε να παίρνει κανεί το λόγο εδώ πριν από την ψηφοφορία, αλλά επειδή είναι η τελευταία συνεδρίαση σα κατά τη διάρκεια αυτή τη εντολή, θα ήθελα εκ μέρου ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου προσωπικά να εκφράσω εδώ τις ευχαριστίες μου σε όλους σας, τον καθένα χωριστά και σε όλους μαζί, σε όλες τις πολιτικές ομάδες για πέντε εξαιρετικά χρόνια κοινή δουλειά που κάναμε και δείξαμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν αποτελεσματικά να συνεργαστούν μεταξύ τους με αυτονομία, σεβόμενοι επίσης και τις διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όσους από εσά συνεργάστηκαν μαζί μου σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια, είτε για την επόμενη θητεία σας εδώ, είτε για οτιδήποτε άλλο κάνετε στη ζωή σας μετά. Σίγουρα θα έχετε πάντα την Ευρωπαϊκή Σημαία στην καρδιά σας. Και όσον αφορά εμένα, έχουμε ακόμα λίγους μήνες αυτή την εντολή και θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε πάνω στα καλά αποτελέσματα που είχαμε μέχρι τώρα και στα μαθήματα που πήραμε αυτά τα πέντε χρόνια. Και προσβλέπω σε συνεργασία με τους νέους ευρωβουλευτές από τότε που θα αρχίσει τις εργασίες του το νέο κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μογκερίνη. Νομίζω εξ ονόματος όλου του Κοινοβουλίου μπορώ να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας και να σας ανταποδώσω ειλικρινείς ε, ευχές. Είναι η τελευταία συνεδρίαση σήμερα και έχουν ζητήσει πολλοί συνάδελφοι το λόγο που δεν ξέρω αν έχει άμεση σχέση με τον κανονισμό. Θα προσπαθήσω ε, να τα ξεκαθαρίσω λίγο, να τα ξεδιαλέξω. Έχει ζητήσει το λόγο δύο συνάδελφοι, δύο κυρίες. Γιατί έχουν απευθυνθεί σε μένα και μου είπανε ε, ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Η κυρία Κώστα πρώτη. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θέλω να πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πόλεων τοποθεσιών της UNESCO. Εδώ θυμόμαστε την Παναγία των Παρισίων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφοσιωθήκαμε φέτος στην πολιτιστική ταυτότητα. Είναι αλήθεια ότι ως Κοινοβούλιο σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Συμμετέχουμε σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και πιστεύω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέρφους για αυτά τα χρόνια συνεργασίας. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι για όλα όσα πετύχαμε στην πολιτιστική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέρφους, τον Πρόεδρο και για την καλή συνεργασία που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κώστα, ε, κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ όλους εσάς που φοράτε αυτό το κίτρινο λουδάκι στο πέτο σας. Είναι πέτειος η τρομερή της εξέγερσης του γκέτο της Βαρσοβίας. Για πολλές μέρες χιλιάδες άνθρωποι στην Βαρσοβία ε, κυκλοφορούν με αυτό το λουλουδάκι για να φωνάξουν ποτέ ξανά. Είμαστε στο τέλος αυτής της θητείας. Αυτό το λουλουδάκι μας θυμίζει για ποια Ευρώπη δουλεύουμε, για την ειρήνη και για το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σας ε, εύχομαι σε όλους σας και σας παρακαλώ να συνεχίσετε να υποστηρίζετε τις ίδιες αυτές αξίες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ρωτήσω τώρα, Θέλει κάποιος το λόγο πραγματικά για κάποιο άρθρο του κανονισμού. Πραγματικά όμως. Όχι. Από ό,τι βλέπω. Ωραία. Ο κύριος Καβαντά έχει ζητήσει το λόγο. Υποπτεύομαι περί τίνος πρόκειται. Θα του δώσω το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Καβαντά. Ευχαριστώ, ε, Αντιπρόεδρε του Κοινοβουλίου. Θα είμαι σύντομος, γιατί δεν θέλουμε να μακρηγορούμε. Για 15 χρόνια ε, λίγες φορές έχω πάρει το λόγο και δεν μακρηγορώ συνήθω. Έχω υποσχεθεί στου ψηφοφόρου μου ότι θα δουλέψω σκληρά και ελπίζω να τα έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Ολοκληρώνω τρει θητείε. Θέλω όλου να σα χαιρετήσω και να σα πω ε, και σε εσά ε, πρόεδρε, είσαστε και η γειτονική χώρα της Γαλλίας, κάτι πάρα πολύ απλό. Η Ευρώπη θα ζήσει η Ευρώπη θα ζήσει και θα επιζήσει παρά εκείνους που θέλουν να μας κάνουν να κλειστούμε στον εαυτό μας. Όμως έχουν σωθεί από τον Μπράντι Εβραίοι, από τον κέντρο της Βαρσοβίας. Είναι η Ευρώπη του Πακάλα και όλων αυτών που έσωσαν την Ευρώπη από τον κομμουνισμό, του Σμιτ και του Κόλλο, του Μπλίτσλαφνε, του Σλοβάκου που έσωσε επίσης παιδιά και ηλικιωμένους του Μπακλαβ Χάβελ και της φίλης μου Σιμών Βέιλ. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι που με βοηθήσετε να γίνω καλύτερος πολίτης από ό,τι ήμουν όταν ήρθα, με σκληρή δουλειά. Όλοι κάτι έχουν να μου μάθουν, ακόμα και αντιπαλοί μου. Σας ευχαριστώ πολύ, να ξέρετε ότι σας αγαπάω πολύ. Χρειάζεται σοφροσύνη και μετριοπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. κύριος Πέτερλε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι τελευταίες αποφάσεις που θα πάρουμε σε αυτή τη θητεία και θέλω να σας ευχαριστήσω για πέντε χρόνια ενότητας μέσα στην ποικιλομορφία. Ευθύνη μας είναι να κρατήσουμε μαζί την Ευρώπη, να ξαναχτίσουμε την Παναγία των Παρισίων. Καλό Πάσχα! Ευχαριστώ πολύ κύριε Πέτερλε. Ψηφίζουμε τώρα. Λοιπόν, πρώτο θέμα Κίνα. Έχουμε μια προφορική τροπολογία της κυρίας Σόιντροβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα. Η προφορική μας τροπολογία είναι στην ιδεολογική σκέψη Α. Κίνα έχει εκφράσει ενδιαφέρον για να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους διεθνούς νόμους ε, στην ανάπτυξή της. Είναι η τελευταία φράση σε αυτή την παράγραφο που βλέπετε. Ε, διαφωνεί κανείς με αυτή την προφορική τροπολογία, όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του ψηφίσματος ε, όπως τροποποιήθηκε προφορικά με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Εάν ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Εγκρίθηκε. Καμερούν. Έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος από επτά πολιτικές ομάδες. Η τροπολογία είναι υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Όλο το ψήφισμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μπρουνέι κοινή πρόταση ψηφίσματο 7 πολιτικών ομάδων, τροπολογία 2, ονομαστική κλίση, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφο 11. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Το τμήμα πρώτον υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη D. Η τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Στο recital ε, Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνονται και τα δύο. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Πάμε στην έκθεση Μωράης τώρα. Μία ε, ονομαστική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα και μοναδική. Εάν ψηφίσατε όλοι, προχωρούμε πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση Μπαλάς. Η κυρία Στέβεν θέλει κάτι να ζητήσει τώρα. Αγαπητέ Πρόεδρε, συνάδελφοι, Σύμφωνα το άρθρο 190 εδάφιο 4 του κανονισμού μας, θα ήθελα να προτείνω εξ ονόματο τη ομάδα ECR να αναβληθεί η ψηφοφορία τη έκθεση Μπαλά για του συντονισμού των συστημάτων κοινωνική ασφάλεια για επόμενη σύνοδο. Δεν είναι ακόμα όριμη προς ψήφιση η έκθεση στην Ολομέλεια. Αν ψηφιστεί τώρα, το μόνο που θα κάνουμε είναι να δείξουμε πόσο διχασμένοι είμαστε και πόσο πολλέ διαφορέ έχουμε τελευταία μέρα τη κοινοβουλευτική περίοδου. Θέλω να παραμείνει ανοιχτό αυτό το θέμα για να το διερευνήσει το επόμενο κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε μια καλή και σταθερή συμφωνία, στιβαρή συμφωνία με υπεραξία για τους πολίτες. Ελπίζω να μπορώ να υπολογίζω στην υποστήριξή σας για αναβολή της ψηφοφορίας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Στέβενς, εξ ονόματος της ομάδας ECR. Ε, ο κύριος Μπαλάς, ο εισηγητής, θέλει να μιλήσει κατά αυτού του αιτήματο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το αίτημα αυτό έχει επαναληφθεί, έγινε και τη Δευτέρα να αναβληθεί. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τη συντηρητική δεξιά για να εμποδίσει απλώς μια συζήτηση και μια δημοκρατική ψηφοφορία. Η συζήτηση έγινε, τώρα έφτασε η ώρα να ψηφίσουμε και να μην θέλουμε να κάνουμε σαν σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων ε, σιωπά θα ήταν το ακρονάωτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλάς. Ψηφίζουμε. Το αίτημα της CCR ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία επί του αιτήματος της ε, ομάδας CCR. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην έκθεση Eckhout. Η τροπολογία 90, προσωρινή συμφωνία, ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Εάν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έτσι ολοκληρώνει την πρώτη αναγνώση του Κοινοβουλίου. Έκθεση GZIP. Προσωρινή συμφωνία. Τροπολογία 87 με ονομαστική κλίση που αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση ΣΒΕΦΚΑ. Και εδώ ε, έχουμε την τροπολογία 41 με ονομαστική ψηφοφορία για την προσωρινή συμφωνία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται ούτως η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Έκθεση Ρέγνερ. Και πάλι η προσωρινή συμφωνία, η τροπολογία 340 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση Κρασνοντέψκη. Έχουμε τις τροπολογίες 32 και 48 με ονομαστική ψηφοφορία μου. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 31 CP1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η 6 αναθεωρημένη και η 13 τροπολογία μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 31 CP2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 34 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. τροπολογία 31 CP 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. CP3 ήταν αυτό. 1 CP1 καταπίπτει. 35 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 31 CP4 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 1 CP2D και 31 CP5D. Είναι ταυτόσιμες αυτές. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 36. 37 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Και αν ψήφισαν όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 31 CP6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1 CP3 καταπίπτει. Η τροπολογία 38 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 39 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 με ονομαστική κλίση αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 31 CP7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 42 με ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 και 41 ταυτόσημες με ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 43D με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ένα CP4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 31 CP8 υπέρ, κατά, αποχές. Α, τώρα θέλει Επαλήθευση αυτό τώρα. Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά ήσασταν πολύ διστακτικοί ορισμένοι. Επαληθεύουμε τη 31 CP8, ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίθηκε. 31 CP9, ονομαστική κλίση αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. Η 44 καταπίπτει. 31 CP10 με ονομαστική κλίση έρχεται ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 31 CP11 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 45. Ε, Δεν καταπίπτει, όχι, την ψηφίζουμε ονομαστικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία 45. Ψηφίσαν Πέρας. Απορρίπτεται. Ένα CP5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 CP10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 1 CP6 ονομαστικά αρχίζει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 31 CP11 με ονομαστική κλίση ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Αγκρίνεται. 47 με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 46 με ονομαστική κλίση ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ένα CP7 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται 31 CP12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία και αν ψήφισαν όλοι λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ολοκληρώνεται ούτω η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον ε, κύριο Λούκε Προσωρινή Συμφωνία Τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Άλλη έκθεση του κυρίου Λούκε προσωρινή συμφωνία, τροπολογία 2 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 δήλωση της Κομισιόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου ολοκληρώθηκε. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Φερνάντες και Γκουαλτιέρη. Η κυρία Αντιπρόεδρος, η κυρία Μογκερίνη, έχει ζητήσει τον λόγο εξ Κομψιών. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους συζητητές Γκουαλτιέρη και Φερνάντες για την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει σε αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ και τις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές, ε, τις επί της τις και όλους τους κοιέδες συζητητές που δούλεψαν σκληρά σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πάντα στηρίξατε την πρόταση αυτή, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Χαιρόμαστε για τη συμφωνία στην οποία καταλήγουν οι συνομοθέτες και θέλω να σας διαβάσω την εξή δήλωση, όπως συμφωνήθηκε στις τριμερείς διαβουλεύσεις. Για την εφαρμογή της σταθερότητας και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τις χώρες, για μια χώρα ή για τις τράπεζες εκ μέρους των χωρών μελών σε θεματικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με πλατφόρμες επενδυτικές. Θέλουμε να σημειώσουμε τα άρθρα 5.1 και 6.1 και το 14.16 κάθετος 97 και το άρθρο 3.4 του κανονισμού 14.67-97. Επιπλέον, ε, με την επιφύλαξη του κανονισμού του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρήσει κατά πόσο πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση στο μέλλον και σε τι βαθμό πρέπει να επιφυληθεί η ίδια αντιμετώπιση όπως για το EFSI, για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε το Invest EU όντως να είναι ο διάδοχος του EFSI με τη συμφορά των χωρών ε, μελών για να χρηματοδοτηθεί με το ίδιο ποσό εγγύηση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε. Υπάρχει μερική συμφωνία, τροπολογία 42, Μπούτς και είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Οπότε οι τροπολογίες που είχαν εγκριθεί τον Ιανουάριο αντικαθίστανται, οπότε περνάμε σε ονομαστική ψηφοφορία από της πρότασης της Κομισιόν. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Εγκρίνεται, ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, περνάμε στην έκθεση Κλούν και εδώ πέρα υπάρχει προσωρινή συμφωνία, τροπολογία 63, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε. εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση TANG και εδώ πέρα υπάρχει προσωρινή συμφωνία. Τροπολογία 2 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται, ολοκληρώθηκε η πρώτη αναγνώση του Κοινοβουλίου. Περνάμε στην έκθεση Γκέρλινγκ. Προσωρινή συμφωνία, τροπολογία 44 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Περνάμε στην έκθεση Λάγγεν. Και εδώ πέρα προσωρινή συμφωνία. Τροπολογία 2. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Περνάμε στην έκθεση Χίμπνερ και εδώ πέρα υπάρχει προσωρινή συμφωνία, τροπολογία 2, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην έκθεση Σάντερ και εδώ πέρα προσωρινή συμφωνία, τροπολογία 2, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ολοκληρώθηκε και εδώ η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Περνάμε λοιπόν σε ένα ψήφισμα που αφορά τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο σχετικά με την νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέταση των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Και τέλος Περνάμε στο ψήφισμα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τροπολογία 2, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 7, αρχικό κείμενο με ονομαστικές ψηφοφορίες, μέρος πρώτο άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται μέρος δεύτερο, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές επίσης εγκρίνεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, Περνάμε τώρα στην τελευταία ψηφοφορία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία σας ε, όλα αυτά τα χρόνια και για την υπομονή σας στα θάλη μου. Αν αδίκησα κάποιους ε, συναδέλφους ζητώ συγγνώμη. Σας εύχομαι καλό Πάσχα και εκλογικό αγώνα εάν ξανακατεβαίνετε και όπως είχα ήδη πει μετά τις επιθέσεις του Στρασβούργου πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το θέμα είναι οι πολιτικές απόψεις, η πολιτική κατεύθυνση αλλά ε, ποτέ δεν είναι οι άνθρωποι αντίπαλοι μας στην πολιτική και στη δημοκρατία. Και τέλος, σας παρακαλώ ε, να πάρετε μαζί τις κάρτες όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, σήμερα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί τόσοι πολλοί συνάδελφοι ήθελαν να μας αποχαιρετήσουν και αυτά τα πράγματα βεβαίω ε, τα ακούσαμε αλλά Ε, θα σας παρακαλέσω να φύγετε λίγο γρήγορα για να περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου, ώστε να φύγουν από την αίθουσα. wir werden dann wieder dazu übergehen, dass wir einige Kollegen namentlich nennen, um den. Λοιπόν, ε, θα αναφέρω κάποιους συναδέλφους τώρα για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Κύριε Κασπάρη, κύριε Προύστ, κύριε Κάρας, κύριε Μπούλμαν. Κύριε Καστάλτο, Ένα μωράκι. Κυρία Τσίμερ, κύριε Σόλτς. Κυρία Γκροστέτ. Κυρία Σούιτσα. Σας ευχαριστώ. στο διάδρομο του ΕΛΚ ε, και στο... του ε, Σοσιαλδημοκρατών προχωρείτε στο βάθος παρακαλώ και μην ομιλείτε στον οδηγό. Περνάμε σε επεξηγήσει ε, ψήφου. Ξεκινάμε την έκθεση Μέτσολα. Δίνω τον λόγο στην κυρία Φορέντσα. Α, έφυγε. Έκθεση Eichhout. Σας παρακαλώ. Ε, εκεί η Γκουε. Κύριε Σόλτς. Κύριε Σόλτς. Δεν με ακούει. Δίνω τον λόγο στον κύριο Σόσνερ, όπως και να έχει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την έκθεση αυτή. Δεν ε, συμφωνώ, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τη λογική που χρησιμοποιείται όταν λέμε ότι ένα όχημα μηδέν εκπομπών είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Μα δεν υπάρχει. Πάντα υπάρχουν κάποιες εκπομπές. Συνεπώς, εγώ πιστεύω ότι είναι μια παγίδα. Δυστυχώς, είναι αυτή η οδηγία στην ουσία ε, είναι κάτι που ψηφίσανε οι ευρωβουλευτές χωρίς να ξέρουν στην πράξη πώς θα λειτουργήσει πώς θα λειτουργήσουν όλες οι διατάξεις που περιλαμβάνει. Οπότε δεν πιστεύω καν ότι θα αποφεληθεί το περιβάλλον από ηλεκτρικά ε, οχήματα. Μα μπορεί να μην είναι τα ηλεκτρικά οχήματα τα οποία εκπέμπουν τις ε, ε, εκπομπές αυτές που ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα, αλλά είναι οι σταθμοί όπου παράγεται ο ηλεκτρισμός. Και τι θα γίνει με τις μπαταρίες, τι θα γίνει με τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ηλεκτρικών αυτών μπαταριών. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια οδηγία που θα απαγόρευε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε. Περνάμε τώρα σε επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση ΣΥΜΠ που αφορά την καθαρή ενέργεια των οδικών μεταφορών. Κύριε Μέσιους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ξεκίνησαν αυτά τα μέτρα, εγώ δεν ήμουνα καθόλου ευτυχής, γιατί είναι χαρακτηριστικό εδώ που μιλάμε για περισσότερο κεντρική διοίκηση, πιο άκαμπτη επιβολή και εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα τονίζαμε τόσο πολύ τα ηλεκτρικά οχήματα για να μειωθούν οι εκπομπές. Όμως, αν έχει νόημα η πράσινη οικονομία, πρέπει να ξέρουμε πώς θα αναπτυχθεί η τεχνολογία, κάτι το οποίο δεν ξέρουμε. Και για τους πολιτικούς που βρίσκονται εδώ και προσπαθούν να υπαγορεύσουν πώς η τεχνολογία και πώς η βιομηχανία θα εξελιχθεί, είναι νοησία. Συνεπώς, δουλέψαμε σκληρά με τον εισηγητή, με τους σκιώδεις εισηγητές και καταφέραμε να ενσωματώσουμε πολύ πιο εύκαμπτες διατάξεις και να υπογραμμίσουμε τη δικαιοσύνη, να αφήσουμε την τεχνολογία να εξελιχθεί και θα δούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Τελείωσαν οι επεξηγήσεις ψήφου για αυτή την έκθεση. Περνάμε στην έκθεση της κυρίου Σβιέφκα που αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Και πάλι ο κύριος Μάθιος. Ευχαριστώ πολύ ε, που μου δίνετε το λόγο και για αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι ζωτική σημασίας οι επιχειρήσεις που θέλουν να ε, δρούν διασυνοριακά να μπορούν να το κάνουν ψηφιακά και μπορούν να το κάνουν χωρίς εμπόδια και χωρίς να προσπαθεί κανείς να σταματήσει τον διεθνή ανταγωνισμό. Εγώ προέρχομαι από τις εκδόσεις. Εκδίδουμε πολλά βιβλία, μπορεί οποιοδήποτε να τα κατεβάσει και η κατάσταση συνεχίζεται. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο επιχειρήσεις μπορούν πιο, εύκολη, πιο εύκολα από μακριά να εμπορευτούν στο διαδίκτυο. Και δεν χρειάζεται πια κάποιος να έχει φυσική παρουσία να πάει σε μια άλλη χώρα για να καταγραφεί εκεί κτλ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μάθιος. Τελειώσαμε και με την έκθεση Σβιεύκα. Περνάμε στην έκθεση Ρέγνερ, διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Και πάλι ο κύριος Μάθιους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πάλι ζήτησα να μιλήσω για την ανάγκη που υπάρχει για ελεύθερες μετατροπές συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Χαίρομαι πολύ γιατί είναι πολύ πιο εύκολο πια όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Και πάλι όταν ξεκινήσαμε με αυτά τα μέτρα, αναφερθήκαμε σε ένα σωρό περιορισμού στις επιχειρήσει ότι θα έπρεπε να αποδείξουν το ένα, το άλλο πριν προβούν σε αυτέ τι δραστηριότητε. Ε, λοιπόν, ευτυχώ δεν ισχύει πια αυτό. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα που κάνουμε προ τα μπρο για το διεθνέ εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το διεθνέ εμπόριο ενισχύει την οικονομία και βοηθάει και βοηθάει και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών. Άρα είναι κάτι πολύ θετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάθιος. Ε, αυτά για την έκθεση Ρέγνερ και ερχόμαστε τώρα σε δύο επεξηγήσεις ψήφου του κυρίου Κρασνοντεύσκη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι. Το σύστημα αξιών της ε, πολιτικής ε, κοινότητας φαίνεται από τους αριθμούς. Η απόφαση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνης ίσως να μην είναι ε, μεγάλο, αλλά είναι σαφές ε, βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Λοιπόν, ε, στην αίθουσα αυτή έχει μιλήσει και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Βέμπερ για το θέμα αυτό. Μιλάμε για τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Αλλά αυτή δεν είναι η σωστή κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να πάει η συνεργασία μας. Τα περισσότερα από τα κράτη μας είναι στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, ε, δεν έχουμε έρθει εδώ πέρα για να δημιουργήσουμε μια πολιτική δύναμη, αλλά για να στηρίξουμε αμοιβαία την ανεξαρτησία των κρατών μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να πάμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Φορέντσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα κατά και δαγκωτό ε, για την έκθεση αυτή που λέει ότι η Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση πρέπει να αλλάξει πορεία. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα άτομα, τους ανθρώπους, τη ζωή, όχι τα σύνορα. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ρισκάρει εδώ πέρα να χρεωθεί όλα αυτά τα ναυάγια που γίνονται στη Μεσόγεια κάθε μέρα μετράμε νεκρούς. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει τα άτομα αυτά, να αντιμετωπίσει την φτώχεια, να φτιάξει ένα σύστημα ευρωπαϊκό και προοδευτικό. Αντιθέτως θεωρώ ότι να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού στρατού σημαίνει ότι ρίχνουμε πόρους που στερούμε από τον αγώνα κατά της ε, ανισότητας και θα ρίξουμε βάρος στα σύνορα και όχι στην υποδοχή. Ευχαριστώ κύριε Φορέντσα. Εδώ ολοκληρώθηκαν οι επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση Κρασνοτέψκη και περνούμε στην έκθεση του κυρίου Τάγκ. Γνωστοποίηση σχετικά με τις εφόρες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας. Ε, η κυρία Μέγερ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι η τελευταία Βρετανή που μιλάω εδώ στο κύκλιο νομίζω, αλλά ίσως και όχι για πάντα. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν είναι μόνο κέρδη για τους λίγους και να αγνοεί τις συνέπειες για όλους τους υπόλοιπους. Ως εργατική ευρωβουλευτής θα ήθελα τα χρήματα που επενδύονται να δημιουργούν περισσότερη δικαιοσύνη στην κοινωνία. Σήμερα αυτό που ψηφίζουμε συνδέει το χρηματοπιστωτικό τομέα με την κοινωνική δικαιοσύνη. Τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία ε, ρηπαίνουν, δεν είναι μια καλή επένδυση, δεν ε, βοηθάει ούτε επίση ε, η δουλειά των παιδιών, η εργασία των παιδιών. Οι ασφαλιστικές εταιρείε επίσης θα πρέπει να δούνε όχι μόνο τα κέρδη τους, αλλά να δουν και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, το θέμα της διαφοράς των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών κτλ. Όλοι μαζί λοιπόν χτίζουμε μια πιο δίκαια Ευρώπη για τους πολλούς, όχι για τους λίγους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μαϊέρ. Προχωρούμε στην επόμενη έκθεση. Το ψήφισμα που αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα ε, εξέταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Πόσπισιλ είναι ο μόνος που έχει ζητήσει το λόγο για επεξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι πραγματικά φρικτό το ότι δεν έχουμε ακόμα εκτελεστικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το δικαίωμα σε εξετιστικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι που παλέψαμε όλη αυτή τη θητεία, αλλά δυστυχώ από πλευρά ε, τη Επιτροπή και ακόμα περισσότερο του Συμβουλίου δεν υπήρξε καμία αντίδραση μέχρι το φθινόπωρο. Ήταν αρνητική πάντα. Ε, δεν ε, εξηγούσαν γιατί δεν θέλανε να προχωρήσουμε. Ελπίζω στην επόμενη θητεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αγωνιστεί περισσότερο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για να διορθωθεί η κατάσταση και να μην υπάρχουν πια τέτοια εμπόδια και ούτε πια ψηφίσματα σαν και αυτό που να καταγγέλουμε την κατάσταση. Πρέπει να μπορούμε αποτελεσματικά να κάνουμε τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πόσπιση. Αυτά για το συγκεκριμένο ψήφισμα. Τώρα έχουμε δύο αιτιολογήσει στο σχέδιο ψηφίσματος για το ολοκληρωμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ο κύριος Φαρία πρώτο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δοκιμές που γίνονται για την τοξικότητα ε, ουσιών είναι κάτι που το κάνουμε εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Και πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν ουσίες οι οποίες κυκλοφορούν μεταξύ μας και έχουν δημιουργήσει προβλήματα γονιμότητας, αλλά κάνουν ε, ζημιά και στο περιβάλλον. Έχει γίνει αξιολόγηση παλιότερα για κάθε προϊόν, χωριστά για κάθε ουσία, αλλά δεν υπήρχε κάτι που να μπορούσε να εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις. Η περίπτωση της διφενόλης, τα μπιμπερό για παράδειγμα, ε, ακούστηκε πολύ και συζητήθηκε πολύ στον τύπο. Άρα, ε, τρώγοντας ή με τα καλλιντικά μπορεί κανείς να κάνει κακό στην υγεία του. Συστηματικά λοιπόν πρέπει να αφαιρεθούν όλες αυτές οι ουσίες γιατί τελικά δρούν στο ορμονικό σύστημα. Και πρέπει να δούμε πώς θα αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο στη συνέχεια. Επιπλέον θα ήθελα εδώ πέρα να πω ότι σε όλη αυτή την θητεία έχουμε συζητήσει πολλές φορές για την υγεία και χαίρομαι που πάνω σε αυτό το θέμα είναι και τελευταία μου παρέμβαση εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαρία. Ο κύριος Σόσνετς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό ε, μπορεί εύκολα να συνοψιστεί. Οι ουσίες αυτές είτε είναι επιβλαβείς είτε όχι, δεν ξέρουμε ποιες είναι καν, αλλά σίγουρα μπορούμε να τις ρυθμίσουμε και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το κάνει αυτό με μαϊστρία. Αυτό δείχνει ότι εμείς δεν μάθαμε τίποτα προ Brexit. Είχαν μπουχτίσει οι Βρετανοί από τις υπερρυθμίσεις σας και την αλαζονία σας και αποφάσισαν να σηκωθούν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν καταλαβαίνετε ότι σας έχει βαρεθεί όλη η Ευρώπη, όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι ελίτ στην Ευρώπη θα χάσουν την εξουσία τους. Εγώ δεν ξέρω ποια είναι τα επιτεύγματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σας οδηγούν να έχετε τέτοια αλαζονία στη στάση σας. Και ποιος σας το δίνει αυτό το δικαίωμα. Εδώ πέρα είναι λέσχη ηλικιωμένων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, δεν μπορείτε να αναπαραχθείτε εσείς οι ίδιοι και βγαίνετε και κάνετε κηρύγματα για τον κόσμο ολόκληρο. Εσεί καταστρέψατε την Ευρώπη και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να καταστραφεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόσνιετ. Εδώ ολοκληρώνονται αυτές οι επεξηγήσεις για το συγκεκριμένο ψήφισμα και τώρα κατ' εξαίρεση θα ακούσουμε ε, ε, άλλη μία επεξήγηση από την κυρία Φορέντζα για την έκθεση Μετσόλα. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, κατανόηση. Καταψήφισα το ψήφισμα αυτό γιατί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σώζει και όχι να συνεχίσει να αποκρούει. Πρέπει να σώσει ανθρώπους από την Λιβύη όπου γίνονται βασανιστήριο. Θεωρώ ότι η χώρα μου ειδικά πρέπει να σταματήσει με την ποινικοποίηση των ΜΚΟ που ξαναξεκίνησε η κυβέρνησή μας που θέλει να περάσει μια ειδική οδηγία κατά του πλοίου Μεντιτερανέα. Και υπάρχουν ε, βεβαίως και οι κατά του Open Arms μιας άλλης ε, ΜΚΟ. Ε, πρόκειται για την τελευταία μου παρέμβαση στην Ολομέλεια. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους για αυτά τα πέντε χρόνια, μαθα πάρα πολλά. Θεωρώ ότι έκανα το καθήκον μου να ε, εκπροσωπώ τους ε, αδικημένους ε, και να προσπαθήσουμε λίγο να είναι όλοι ευτυχείς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φορέντσα. Ολοκληρώνονται εδώ οι αιτιολογίε ψήφου. Τα πρακτικά, τα συνοπτικά τη χτεσινή συνεδρία και τα εγκεκριμένα κείμενα διατίθεται. Έχετε αντιρρήσει. Όχι, ούτω και εγκρίνονται αυτά τα συνοπτικά πρακτικά. Ε, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, θα διαβιβάσω αρμοδίω ε, τα ψηφίσματα και τι αποφάσει που λάβαμε. Είναι η τελευταία συνεδρίαση τη περίοδου συνόδου, γι' αυτό προτείνω ε, κατά παρέκκληση του άρθρου 92 να εγκριθούν τώρα τα συνοπτικά πρακτικά και αν δεν διαφωνεί κανείς ούτως εγκρίνονται τα συνοπτικά πρακτικά τα σήμερα, Ε, ευχήθηκα στους συναδέλφους, θέλω να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες για την εργασία τους ε, κατά τη διάρκεια της θητείας και της εβδομάδας αυτής και σας εύχομαι καλό Πάσχα και ευλογημένη επάνωδο ε, στις αιστείες σας. Και με το καλό το νέο κοινοβούλιο από το καλοκαίρι. Διακόπτεται η περίοδος συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λέει τη συνεδρίαση.